Uh, Καλή σας μέρα αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ήδη αργοπορήσει ε, και ε, έχω την αίσθηση, πρέπει να ξεκινήσουμε, έχω την αίσθηση ότι μερικοί συνάδελφοι θεωρούν ότι το πρωί δεν είναι η μέρα εργασίας, σαν να ήταν Δευτέρα. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να σας καλωσορίσω όλους, να σας πω ότι θα πρέπει πρώτα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Το μοναδικό θέμα επ' αυτής ε, είναι ε, η δημόσια ακρόαση όσον αφορά το θεσμικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Συνθήκης της Λισαβόνας και πέρα από αυτά. Ε, θεωρώ ότι έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, δεύτερο σημείο είναι οι ανακοινώσει ε, τη Προέδρου. Δεν έχω τέτοιε ανακοινώσει, επομένω μπορούμε να περάσουμε άμεσα στην συζήτησή μα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα και πολύ σύντομα ε, και πριν ζητήσω από του συζητητέ να παρουσιάσουν τι απόψει του, να πω κάποιε ιδέε οι οποίε είναι οι προσωπικέ μου απόψει βέβαια, αλλά που ελπίζω ότι θα τι ημερίζεστε. Νομίζω ότι τώρα πια μπορούμε να δούμε ε, με ε, σαφήνεια ότι ζούμε δύσκολες, κρίσιμες στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας ε, και πιστεύω ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική ανάγκη για αλλαγή και πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, τα διακυβέρματα της προκλήσεις ε, με την αίσθηση του κατεπήγοντος. <clears throat> Έχουμε τις ε, συνθήκες, περισσότερες από τις, οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές συνθήκες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το θεσμικό έλλειμμα. Θεωρητικώς οι συνθήκες στην ουσία επιβεβαιώνουν του παρελθόν και δεν δημιουργούν έτσι, δεν δίνουν μια νέα όθηση στο μέλλον. Δεν έχουμε πραγματικά συνθήκες εξάντε. Και επομένως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το συζητήσουμε αυτό. Ε, αυτό το κενό θέλουμε τώρα να συζητήσουμε, αυτή την ανάγκη κάλυψης του κενού θέλουμε να συζητήσουμε και ε, να δούμε κατά πόσο να μπορεί ε, και πόσος χώρος υπάρχει για αυτήν την θεσμική ε, προσέγγιση. Έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν για τα θέματα αυτά. Θα έχουμε, έχουμε προβλέψει δύο πάνελς για την σημερινή μας ακρόαση, μια μισή ώρα το καθένα. Το πρώτο, στο το πρώτο πάνελ θα ασχοληθεί ε, με κάποια τομεακά ας πούμε θέματα, θα δει δηλαδή τις διάφορες περιοχές ας το πούμε ε, της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ το δεύτερο πάνελ θα ασχοληθεί με πιο οριζόντια ε, ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν χωρίς καθυστέρηση να ζητήσω από τους εισηγητές Μπρέσοφερ, Χόφστατ και Μπρόκ τους εισηγητές μας να κάνουν τις αρχικές τους ε, παρατηρήσεις. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο τη διαθεσή, μου, παρακαλώ, μας. Παρακαλώ λοιπόν να είσαστε ε, σύντομοι. Δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει πρώτος το λόγο, ποιος θα μιλήσει πρώτος. Ε, κανείς καμιά φορά δεν ξέρει αν είναι καλύτερο να ξεκινήσει ή να μιλήσει τελευταίος. Ο Έλμαρ νομίζω ότι δεν με ακούει καν, δεν με προσέχει. Έτσι κι αλλιώς δεν θέλω να μακρηγορήσω διότι προτιμώ να ακούω και θέλω να ακούσω σήμερα. Σήμερα βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων. που ε, κυρίως είναι υπό το πρίσμα της σημερινής μου αρμοδιότητας εξωτερικών και ασφαλείας και υπάρχουν κάποια ζητήματα ε, που δεν αναφέρονται και δεν εφαρμόζονται. κυρία Μπρέσο και εγώ ασχολούμαστε με την εξάντληση της Λισαβόνας και ο Γκί Φερχόφστατ κάνει προτάσεις ε, για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν και εγώ θα περιοριστώ στο πρώτο να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί ακόμα να εξαντληθεί, δηλαδή να αξιοποιηθεί στο έπακρο η συνθήκη της Λισαβόνας και υπό τις παρούσες συνθήκες ε, καταλαβαίνετε ότι για πολιτικούς λόγους δεν επίκειται αναθεώρηση των συνθήκων μετά τις εξελίξεις στην Πολωνία την Κυριακή, ε, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ενθαρρυντική την κατάσταση για ε, ταχεία πρόοδο. Ε, οι διαπραγματεύσεις που θέλει να διεξαγάγει η Μεγάλη Βρετανία επίσης δεν εμνοούνται σε επίπεδο τροποποίησης των συνθήκων. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς αλλά σε επίπεδο ε, ερμηνείας ας πούμε, των συνθήκων, ε, σε αυτό που λένε closer union, μια πιο κοντινή ε, ένωση. Τι θα πει αυτό, είναι φιλολογικό. Και από ό,τι φαίνεται έπαιξε όμως αποφασιστικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία στην Μεγάλη Βρετανία. Και είναι ενδιαφέρον και αστείο και για το αυτό το Ever Closer Union ε, τα αρχικά βγάζουν Q και ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός ήρθηκε να δεχτεί τη συνθήκη του Μαστρίχτ. Αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι ενδιαφέροντα και έχουν να κάνουν και με την εσωτερική πολιτική, όχι μόνο την εξωτερική, μετανάστευση και άλλε διαστάσεις. Οπότε... Θα πρέπει να δούμε ότι πρέπει να μπει στη συναπόφαση και η πολιτική εσωτερικών και δικαιοσύνης που σε μεγάλο βαθμό έχει κινητικοποιηθεί. Δεν έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες που υπάρχουν. Και θα συζητήσουμε ε, την μετανάστευση. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις και πάλι. Θα πρέπει να απαντήσουμε τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δούμε αυτό το δράμα και την τραγωδία των προσφύγων και των μεταναστών. Ε, ε, δούμε τι δυνατότητες έχουμε. Και από την άλλη η ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ιδιαίτερες επιθυμίες των Βρετανών. Δεν μπορεί ένας Ευρωπαίος πολίτης που τέσσερα χρόνια δουλεύει και πληρώνει φόρους σε μια χώρα, νομικά δεν είναι δυνατόν να διανοηθεί κανείς ότι δεν μπορεί να έχει κάλυψη ασφαλιστική κτλ. Όλα αυτά είναι ζητήματα ε, του πυρήνα ε, των όσων θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την ΟΝΕ. Αναμένεται τώρα ένα έγγραφο των πέντε ε, προέδρων. Υπάρχει, δεν υπάρχει, κυκλοφορεί, δεν ξέρω. Για να δούμε τι θα γίνει στο πλαίσιο των συνθήκων, τι επιτρέπεται για την καλύτερη διακυβέρνηση και για θέματα συντονισμού της οικονομικής πολιτικής καθώς και την επιβολή δημοσιονομικής εξυγίανσης και μεταρρυθμίσεων, έτσι, διαρθρωτικών. Και αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα δεν είναι τόσο πολύ να αξιολογήσουμε ποιος από μας βρίσκεται σε ποια πολιτική παράταξη, τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε, αλλά τι δυνατότητες μας δίνει η συνθήκη, το πλαίσιο, το θεσμικό. Τώρα πώς θα το ερμηνεύσουν, δεν είναι δική μας δουλειά ή πώς θα το αξιοποιήσουν. Εμείς πρέπει να το δούμε από τη θεσμική πλευρά και τη συνταγματική ας πούμε των συνθήκων. Γι' αυτό παρακαλώ να εξετάσουμε επίσης και να ελέγξουμε με ποιο τρόπο θα φέρουμε περισσότερο στο παιχνίδι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή, δυστυχώς, μετά από τη συντακτική συνέλευση και τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, επέμειναν τα κράτη-μέλη και πέρασαν την άποψή τους να εξαιρούνται τα θέματα της ΟΝΕ από τη δικαιοδοσία του ΔΕΚ. Αυτό το θεωρώ πρόβλημα κράτους δικαίου, γιατί δεν ξέρω πώς μπορούμε κάπως κάτι να κάνουμε παρά το κείμενο των συνθήκων. Και αμέσως απορρέει εδώ το επόμενο θέμα. Ήμασταν πάρα πολύ περήφανοι για το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί ο Ευρωπαίος πολίτης και ε, για να μπει στην ΕΣΔΑ η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τότε το ΔΕΚ με νύχια και με δόντια είχε αντιταχθεί στο να είναι εκείνο αρμόδιο για, και να είναι το δίκαιο δοτικό όργανο για το χάρτη των θημελιωδών δικαιωμάτων. Και τώρα ανθίσταται να προσχωρήσουμε στην ΕΣΔΑ γιατί θέλει να είναι ε, αρμόδιο αποκλειστικά το ίδιο. Δηλαδή στροφή 180 μοιρών. Σε σχέση με την προδεκαετία στάση του. Ε, και αυτό θα είχε νόημα να το εξετάσουμε και να το κοιτάξουμε. Και να δούμε ε, πώς θα συναντηθούν στο Στρασβούργο οι εθνικές ε, δικαιοδοσίες και οι ευρωπαϊκοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, αυτά θα χρειαστεί να τα διερευνήσουμε, να τα εξετάσουμε, αλλά θα υπάρξουν και άλλα ελλείμματα, φαντάζομαι, και ανάγκες που θέλω να ακούσω από πλευρά σας για να δούμε πώς θα τα καλύψουμε και πώς θα τα ρυθμίσουμε. Και θέλουμε να ακούσουμε από τους επιστήμονες μας, γιατί εμείς οι βουλευτές δεν είμαστε επιστήμονες, είμαστε κάτι αδαείς βουλευτές εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ελμάρ, η Μερσέντες Μπρέσο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο στόχος αυτής της ακρόασης είναι πρωτίστως να ακούσουμε την άποψη των εμπρογνωμόνων που έχουμε προσκαλέσει και φυσικά όλων των ε, υπολείπων συμμετεχόντων για αυτή τη βιτή σχέση που, τη διτή έκθεση συγγνώμη, που ετοιμάζουμε εμείς οι τρεις ε, εισηγητές που θα έχει ένα κοινό τμήμα που θα αφορά τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δύο ξεχωριστά τμήματα. Μία ε, η έκθεση που υπογράφει ο συνάδελφος Μπρόκ και εγώ και την άλλη έκθεση που υπογράφει ο συνάδελφος Φερχόφστατ αφενός ως προς τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις εκμεταλλευόμενοι στο μέγιστο τη συνθήκη της Λισαβόνας που έχει τεράστιες δυνατότητες ακόμα και αφετέρου στην έκθεση Φερχόφστατ όταν απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις, ε, τροποποίηση των συνθήκων. Οι προκλήσεις λοιπόν που έχουμε εντοπίσει αρχικώς είναι προφανώς το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης, το θέμα της δημοκρατίας και της ε, νομιμότητας της δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θέμα της εξωτερικής πολιτικής, ε, για το οποίο μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο υπήρξε ένα σημαντικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το θέμα των ε, ε, προσαρμογών ε, σε θεσμικό επίπεδο. Εγώ φυσικά εδώ δεν έχω χρόνο να σταθώ σε όλα τα σημεία, αλλά όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση υπάρχουν σαφέστατα μέσα τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε σε επίπεδο συνθήκων, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η ενεργειακή ένωση, η ψηφιακή αγορά, η τραπεζική ένωση υπάρχουν ε, κάποια ζητήματα τα οποία επικαλύπτονται, όπως για παράδειγμα οι φορολογικές δυνατότητες, τη δυνατότητα ε, ελλείμματος στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δεν αναφερόμαστε σε έλλειμμα στα κράτη-μέλη, αλλά σε δυνατότητα έλλειμματος στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Όπως γνωρίζετε ήταν ένα από τα προβλήματα τα οποία ε, αντιμετωπίστηκαν. Και αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν βεβαίω και είναι και θέματα που συζητούμε μεταξύ μας. Όσον αφορά τώρα τα θέματα τα οποία αφορούν τη δημοκρατία, Υπάρχουν ακόμα μια σειρά αποζητήματα τα οποία αφορούν τον εκλογικό νόμο, ε, τα συζητήσαμε και πιο συγκεκριμένα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών, Υπάρχει και όλο αυτό το τεράστιο ζήτημα της ελεύθερης ε, κυκλοφορίας μεν, αλλά ε, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ε, προσέγγιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, επομένως η η τρίτη ηλικία αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες όταν έχουν αποφασίσει ότι θα μπορούν να ζήσουν σε διάφορες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ουσιαστικά τα δύο νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πρέπει να τα συζητήσουν όλα αυτά. Και φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχω χρόνο να θίξω. Ένα τρίτο ζήτημα, η τρίτη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, είναι ένα όλο ένα και πιο περίπλοκο ζήτημα. Είναι ακόμα πιο δύσκολο πλέον να κάνουμε διάκριση μεταξύ εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ε, και γενικότερα μεταναστευτική πολιτική, ε, αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική ασύλου, όλα αυτά τα θέματα αντιμετωπίζονται πλέον συνολικά και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως σύνολο. Η δυνατότητα λοιπόν χρήσης κάποιων μέσων, όπως για παράδειγμα διαρθρωμένη συνεργασία σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί τουλάχιστον ε, κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει να προχωρήσουν και να ε, έχουν κάποιες πολιτικές ασφάλειας και άμυνας και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία βρίσκονται εντός της συνθήκης της Λισαβόνας αλλά πέραν αυτού υπάρχουν και άλλες ε, δυνατότητες εάν φυσικά τροποποιηθεί η συνθήκη. Βάσει συνθήκη πολλά πράγματα όμω μπορούν να επιτευχθούν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα κάλεσε αρκετά κράτη, ε, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν κάποια πιο ενισχυμένη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Τέλος, το θέμα της θεσμικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι διάφορες προκλήσεις έχουν διάφορες συνέπειες όσον αφορά τις θεσμικές, τις πτυχές. Για παράδειγμα, το πώς αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, ο προπολογισμό της Ευρωζώνης, την πιθανή ε, φορολογική πολιτική είτε τη Ευρωζώνης είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η δυνατότητα ή ε, το κατά πόσον θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη ε, μεταβλητής γεωμετρίας. Πρόκειται λοιπόν για ζητήματα τα οποία αφορούν τις θεσμικές πτυχές και συνδέονται με τα θέματα τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Επομένως και για αυτό το ζήτημα αναμένουμε και τις απόψεις σας. Ε, κάτι τελευταίο, ε, κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις δικές μας εκθέσεις, ε, είναι αντικείμενο μιας άλλης έκθεσης, αλλά στα θεσμικά ζητήματα υπάρχουν και κάποιοι προσανατολισμοί που διαβάσαμε από το έγγραφο που λάβαμε μόλις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλύτερη νομοθεσία και κάποια από αυτά τα ζητήματα ίσως θα μπορούν να συζητηθούν και σε, ε, να είναι τμήμα αυτής της θεσμικής συζήτησης γιατί το έγγραφο αναφέρεται και σε κάποια από τα ζητήματα ε, τα οποία απασχολούν και εμάς στην έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε κύριο Φερχόφστατ. Ευχαριστώ πολύ, πολύ σύντομα για την δεύτερη έκθεση για το θεσμικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχέση με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας αρχικά δεν θέλησαμε να δούμε πώς θα μπορούσε να αναθεωρηθεί η ισχύουσα συνθήκη και την όλη διαδικασία απλώς να εντοπίσουμε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα και κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές η έκθεση θα επικεντρωθεί σε τέσσερα ζητήματα. Πρώτον, το θεσμικό οικοδόμημα της Ένωσης, κυρίως το ερώτημα της Βρετανίας και το όλο θέμα που έχει προκύψει και το κατά πόσο είναι δυνατόν να έχουμε διαφορετικούς κύκλους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσους χρειαζόμαστε Διότι αν κοιτάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση προσεκτικά υπάρχουν τουλάχιστον 10 όχι μία ενώσεις με διαφορετικές εξαιρέσεις, διαφορετικές μεταχειρήσεις, διαφορετικές διαδικασίες. Τώρα ίσως είναι η στιγμή αυτά να διορθωθούν, να αποσαφενιστούν. Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η έκθεση. Μετά είναι η οικονομική διακυβέρνηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωζώνης, όπου είναι απολύτως αναγκαίο να προβλέψουμε ένα σύστημα διακυβέρνησης λαμβάνοντας υπόψη και νομισματική ένωση που ήδη ισχύει. Τρίτο πρόβλημα είναι η δημοκρατία και η λογοδοσία. Τι πρέπει να γίνει για το ρόλο του καθενός, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα άλλα θεσμικά όργανα εντό Ένωσης και πώς μπορούμε να αυξήσουμε την, το βαθμό δημοκρατικότητας και λογοδοσίας. Και το τελευταίο ζήτημα είναι η εξωτερική πολιτική και ο γεωπολιτικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε δηλαδή τις περαιτέρω εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της δεύτερης έκθεσης και ίσως ολοκληρώνοντας να θυμίσω ότι το, το ευρωβαρόμετρο του 2014, στα τέλη του 2014, δείχνει σαφώς ότι το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι θέμα κοινή γνώμης, αλλά η έλλειψη τόλμης και οράματος της πολιτικής ελίτ. Αναφέρομαι στη μελέτη του Ευρωβαρομέτρου του 2014, του τέλους του 2014, διότι έδειξε ότι οι πολίτες θέλουν περισσότερη ένωση, περισσότερη ολοκλήρωση. Παρά τις διαφορές και τις αποκλήσεις ευρωζώνης και μελών ευρωζώνης και μη μελών, οι αριθμοί είναι πολύ σαφεί. 56% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπέρ της Οικονομικής και Νοσματική Ένωσης και του ευρώ. 66% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπέρ της ενίσχυσης της κοινή εξωτερικής πολιτικής και 76% του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι υπέρ μιας κοινή πολιτικής άμυνας. Αν είχα τέτοιου αριθμούς ε, και στις εκλογές, τέτοια ποσοστά, 56, 66 και 76, θα ήταν πολύ ωραία. Αλλά είναι σαφής, σαφές το δείγμα. Και με αυτό θέλω να ολοκληρώσω το πρόβλημα με τα θεσμικά όργανα δεν είναι ότι η κοινή γνώμη δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν Αυτό το ακούμε συχνά με το αποτέλεσμα των ε, ευρωεκλογών, ευρωσκεπτικισμός, ε, καχυποψία, έλλειψη εμπιστοσύνη, ότι ο ευρωπαϊκό πληθυσμό δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύει όμω το αντίθετο. Με τέτοιου αριθμού 66% για την ε, Οικονομική Ένωση και 76% για την πολιτική άμυνα, νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να αναλάβουμε τι ευθύνε μα και καλώς το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να συντάξει αυτές τις δύο εκθέσεις. Χαιρόμαστε λοιπόν για τη συμμετοχή των εξαιρετικών εμπειρογνωμόνων μας. Και αναμένουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε στο πρώτο πάνελ. Έχουμε τρεις ομιλητές. Να ξεκινήσω με το Ρενέ Ρεπάζη. Τι να πω για σας, Ρενέ. Συντονίζετε το έργο τριών ε, ε, πανεπιστημίων, του Ρότερνταμ, του, της Δέλφτ και του Λάιντεν. Είστε κοντά στις Βρυξέλλες και έχετε μεγαλύτερη πρόσβαση στη γνώση και τις διάφορες διαφορετικές θεωρήσεις που υπάρχουν για τα θέματα αυτά. Ελπίζουμε λοιπόν να φωτίσετε τις συζητήσει μας και καλώς θα ξεκινήσουμε με εσά τις συζητήσεις μας για το θέμα αυτό, για το μέλλον της Ευρώπης. Έχετε το λόγο, καθηγητά Ρεπαζή. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, ωραία εισαγωγή που κάνατε. Καλημέρα και στα μέλη της Επιτροπής σας. Ευχαριστούμε πολύ που με... Ε, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σε αυτή τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα πλαίσια και πέρα από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω κάνοντας μια, μια αναφορά και μια μικρή σύντομη εισαγωγή ε, όσον αφορά το θέμα και μετά βεβαίως, μια και έχω μόνο 15 λεπτά, ε, θα κάνω κάποιες επιλογές. Θα μιλήσω για τρία θέματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μιλήσω για τον τρόπο ε, επιβολής μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί υπό την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Δεύτερον, θα αναφερθώ στο θέμα της δημοσιονομικής ικανότητας της Ευρωζώνης και τρίτον το θέμα της ενίσχυσης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια αυτής της διακυβέρνηση. Ε, η συνθήκη τη Λισαβόνα δεν άλλαξε την βασική την βασική δομή της Οικονομικής και Νομισματικής ε, Ένωσης ε, η οποία ε, είχε εισαχθεί από τη συνθήκη του Μάστριχτ και είναι υπερεθνική. Αντιτίθεται αρχικά στην παραδοσιακή τεχνοκρατική πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε οι εθνικές δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές να τροποποιηθούν έτσι ώστε να αποκτήσουν ευρωπαϊκή διάσταση. Ε, όμως, ε, κατά αυτή την έννοια δεν υπάρχει μηχανισμός ε, επιβολής αυτών των μέτρων. Ε, από τη στιγμή που τα κράτη-μέλη δεν έχουν την ίδια θέση στις οικονομικές αγορές, ε, ε, οπωσδήποτε θα υπάρξουν τροποποιήσεις οι οποίες θα καταδεικνύονται από την άνοδο ή την πτώση των επιτοκίων. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ούτε ρήτρα bailout, ούτε και ε, δυνατότητα αγοράς των ε, κυβερνητικών ομολόγων από πλευράς των πρωτογενών ε, αγορών βάσει του άρθρου 123 της Συνθήκης Λειτουργίας. Η ο κύριος θεσμός όσον αφορά την Νομισματική Ένωση είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία έχει ανεξαρτησία απέναντι σε θεσμούς και κυβερνήσεις. Ε, απ' την άλλη πλευρά ο κύριος ε, φορέας ε, και θεσμός της Οικονομικής Ένωσης είναι το Συμβούλιο το οποίο συντονίζει όλους τους υπολείπους και όλες τις διαδικασίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά αυτή την έννοια δεν έχει μεγάλο ρόλο στην υπερεθνική Νομισματική ε, Ένωση λόγω ακριβώς ε, της ανεξαρτησίας ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτε και έχει μεγάλο ρόλο να παίξει στην νομισματική πολιτική λόγω ακριβώς της δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όσον αφορά θέματα τα οποία αφορούν την οικονομία ε, υπάρχει ε, ο, ο διεθνής, το διεθνές δίκαιο καθώς επίσης και οι της μορφές ελέγχου. Αυτή η βασική κατασκευή, αυτή η βασική δομή δεν μπορεί να τροποποιηθεί πέρα και χωρίς μια επίσημη τροποποίηση των συνθήκων. Μπορεί να παραχθεί δευτερογενές δίκαιο όπως ας πούμε ήταν το 6-pack ή το 2-pack και επίσης σε διαδικασίες όπως το Fiscal Compact ή ο Μηχανισμός Σταθερότητας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε αυτή την άποψη στην απόφαση της υπόθεσης ε, Pringle όπου αποφάσισε και απεφάνθη ότι ε, ε, οι αποφάσει αυτές είχαν ληφθεί πριν από την θέση εφαρμογή του άρθρου 136 παράγραφος 3 της Συνθήκης Λειτουργίας. Πέρα από αυτήν την αλλαγή των συνθήκων, οπωσδήποτε θα πρέπει ο μηχανισμός σταθερότητας να συμμορφούνται προς τις αρχές της, ε, της αναφερόμενης της συνθήκες έτσι ώστε να είναι ε, νομιμοποιημένος. Και αυτό αναφέρεται στο άρθρο 152 της Συνθήκης Λειτουργίας. Ε, αυτή η ε, ασυμμετρία η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης σημαίνει. Σημαίνει ότι ε, όταν ο συντονισμός των κρατών μελών όσον αφορά τις οικονομικές και δημοσιονομικές τους πολιτικές φτάνει στα άκρα της και στα όρια της θα πρέπει να υπάρχει μια υπερεθνική διάσταση. Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτή η υπερεθνική διάσταση της Οικονομικής Ένωσης θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα μπορούσαν να ε, δοθούν, ε, να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ε, αυτό θα σημαίνει επίσης ότι η συνθήκη αλλάζει με έναν απαρέγκλητο τρόπο έτσι ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση της Οικονομικής Ένωσης. Για να υπάρξει αυτό το δυναμικό και για να μπορέσει να λειτουργήσει στα πλαίσια αυτών των δυνατοτήτων προτείνω ενίσχυση, προτείνω να υπάρχει ε, ενίσχυση της συνθήκης λειτουργίας. Ε, σύμφωνα με το άρθρο 121 της συνθήκης λειτουργίας ε, και έτσι ώστε να μπορέσουν και βάσει του άρθρου 148 της συνθήκης λειτουργίας να εφαρμοστούν κοινέ πολιτικές απασχόλησης θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα γιατί διαφορετικά δεν θα είναι νόμιμες και μόνιμες συγγνώμη, αυτές οι δυνατότητες. Τι, τι εννοούμε όταν λέμε δυνατότητες δυνατότητες ενίσχυσης. Πρώτα απ' όλα θα μπορούσε να υπάρχει η ιδιωτική ενίσχυση έτσι ώστε ε, τα μη συμμορφούμενα κράτη-μέλη να υποχρεωθούν ε, να τροποποιήσουν την οικονομική δημοσιονομική τους πολιτική. Δεύτερον, μπορεί να υπάρχει δημόσια ενίσχυση. Στα πλαίσια αυτής ε, της δημόσιας enforcement μπορεί κανείς να διαλέξει διάφορες πολιτικές. Ένα τρόπο θα μπορούσε να είναι το λεγόμενο naming and shaming, να δείχνεις με το δάχτυλο δάχτυλο τους ε, υπέτειους της ε, ε, και να τους υποχρεώνει να τροποποιήσουν τις αλλαγές, να, να τροποποιήσουν την στάση τους. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι ε, ας πούμε να, ε, υπο, ε, υποχρεωθεί το κράτος μέλος το οποίο παρεκκλίνει στην υποχρεωτική συμμόρφωση αλλά βεβαίως αυτό σημαίνει ότι η υπερεθνική διάσταση της οικονομίας θα πρέπει να γίνει δεκτή από όλους. Αυτή τη στιγμή η πολιτική η οποία ακολουθείται είναι μια συλλογή ας πούμε των στοιχείων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ε, ωστόσο θα πρέπει ε, ε, σε περίπτωση που υπάρχουν παρεκκλίνουσες συμπεριφορές ή λανθασμένες συμπεριφορές τότε θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας πιστικός μηχανισμός επιβολής του νόμου. Οι οικονομικές κυρώσεις είναι αυτές οι οποίες είχαν εισαχθεί από το Six Pack και βασίστηκαν σε κανονισμούς που είχαν βασιστεί με τη σειρά τους στα άρθρα 120 121 παράγραφος 6 και 136 της συνθήκης λειτουργίας ε, σε περίπτωση όπου αναφέρονται οι υπερβολικές ε, αποσταθεροποίησεις όσον αφορά τα ισοζύγια. Ε, στη δεύτερη περίπτωση κατανοούμε ότι το άρθρο 126 παράγραφος 11 αναφέρεται σαφώς σε κυρώσεις οι οποίες ε, ε, ε, καταφέρονται εναντίον κρατών μελών που δεν ακολουθούν την υποχρεωτική διορθωτική πολιτική που προβλέπεται στο Stability Growth Pact. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν κυρώσεις εναντίον κρατών μελών όπου ο πρωτογενής, το πρωτογενές δίκαιο δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να αλλάξουν την οικονομική τους πολιτική. Αυτό με οδηγεί στο τελευταίο μου ε, τμήμα κατά κάποιο τρόπο το οποίο αφορά τα κίνητρα. Ε, από τη στιγμή που δεν μπορούμε ακριβώς να ε, ασκήσουμε κυρώσεις ε, όσον αφορά την μη ε, συμφωνία, ας πούμε, ή συμμόρφωση και από τη στιγμή που έχουμε τον κανονισμό που βασίζεται το άρθρο 121 παράγραφος 6 της Συνθήκης Λειτουργίας θα πρέπει να αλλάξουμε την, τον, τον τρόπο αντιμετώπισης μας. Μία τέτοια, μία τέτοια νομική διευθέτηση δεν θα, θα ερχόταν σε αντίθεση ε, με το πρωτογενές ε, δίκαιο, σε αντίθεση με τις ε, κυρώσεις και ούτε θα μπορούσε να δώσει την δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ζητήσουν οικονομική βοήθεια από τη στιγμή που θα ήταν διαπιστωμένη η μη συμμόρφωση. Σε αυτά τα πλαίσια θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να σας αναφερθώ στην ιδέα της ε, Ενσωμάτωση ε, και του ε, δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην Ευρωπαϊκή Πολιτική είτε πρόκειται για οικονομική είτε για δημοσιονομική όμως τα άρθρα 121 παράγραφος 6 αλλά και το άρθρο 136 δίνει την δυνατότητα αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το θέμα των πληρωμών το οποίο ε, αναφέρθηκε σε σχέση με τα φορολογικά κίνητρα ε, στην ουσία μας οδηγεί στην, σε μια συγκεκριμένη ερώτηση ε, και επομένως οδηγούμεθα εις το δεύτερο τμήμα της παρέμβασής, της παρέμβασής μου κρίνοντας ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια, ένας μηχανισμός υποχρέωσης συμμόρφωσης βάσει βάση κινήτρων, ε, ε, βάσει των άρθρων που ανέφερα προηγουμένως 121.6 και 136, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως δεν είναι δυνατόν να δοθούν τέτοιου είδους κίνητρα. Η απάντηση όμως στην ερώτηση αυτή είναι, ε, θα πρέπει να βρεθεί μάλλον εις την νομοθεσία η οποία διέπει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρεται σε αυτό το θέμα στο γενικό κεφάλαιο της ενότητας του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμμόρφωσή του. Ο, ε, το, το, ο νόμος που αφορά το, ε, ε, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς δίνει αυτήν την σχέση ανάμεσα στον, στις δαπάνες και τα έσοδα ακόμα πιο ε, σημαντικό και ιδίως ε, όταν ε, θυμηθούμε και τις πολύ περίεργες συζητήσεις για τα πολυετή οικονομικά δημοσιονομικά προγράμματα είναι στα πλαίσια αυτών των δημοσιονομικών πολιτών προγραμμάτων να δούμε ακριβώς τον κανονισμό ο οποίος έχει ένα ενδιαφέρον ε, ένα ενδιαφέρον σημείο, το ε, σημείο της αιτιολογικής σκέψης 8, όπου αναφέρει συγκεκριμένα ότι ε, το MFF δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ε, θέμα του προϋπολογισμού τα οποία μπορούν να ε, χρηματοδοτηθούν από συγκεκριμένη ισοδηματική πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε κονδύλι έχει ήδη ταυτοποιηθεί για συγκεκριμένη διαδικασία δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για οτιδήποτε άλλο. Εξορισμού, επομένως, θα πρέπει κάτι τέτοιο να χρηματοδοτηθεί χρηματοδοτηθεί από όλες τις ε, χώρες ε, μέλη. Αυτό αναφέρεται ε, και στα άρθρα τα οποία αναφέρονται στην ενισχυμένη συνεργασία. Κατά την ίδια έννοια όλες οι, όλες οι δαπάνες θα πρέπει να αναφέρονται και να είναι να χρεώνονται κατά κάποιο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και διαφοροποιημένες οικονομικές συμβολές θα πρέπει να θεωρούνται ήδη οι πόροι ε, και επομένως να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και αυτό βάσει του άρθρου 311 της Συνθήκης Λειτουργίας. Ε, ε, ε, εν ε, κατακλείδη, το παρόν πλαίσιο της συνθήκης δίνει την δυνατότητα στην δημιουργία ενός προϋπολογισμού της Ευρωζώνης. Ε, μέσω επιπλέον και ε, επιπλέον οικονομικών συμβολών που θα πρέπει οπωσδήποτε όμως ε, να βασιστούν στο άρθρο 311 αλλά τροποποιημένο. Το τελευταίο σημείο μου αναφέρεται στην εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι γεγονός ότι δεν έχει πάρα πολύ ισχυρό ρόλο ε, στις διαδικασίες στις οποίες μέχρι τώρα έχω αναφέρει. Αυτό απορρέει από τις συνθήκες. Αλλά αν ε, θέλουμε να, αναφέ... να ενισχύσουμε τον ρόλο ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρα από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μπορούμε να κάνουμε τα εξής θα μπορούσε κανείς ε, να θεωρήσει ότι μέσω της ε, επέκτασης ε, της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας θα μπορούσε να τροποποιηθεί αυτή η εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Επίσης θα μπορούσε να υπάρξει εναρμόνιση διαφόρων, διαφόρων νομικών περιοχών βασιζόμενη στα άρθρα 113 και το άρθρο 115 όσον αφορά ας πούμε τους έμεσους ή άμεσους ε, φόρους, καθώς επίσης και όσον αφορά ε, την κοινωνική νομοθεσία, άρθρο 153 της Συνθήκης ε, Λειτουργίας. Θα μπορούσε κανείς βεβαίως να διαλέξει και τροποποίηση της νομικής βάσης χρησιμοποιώντας το άρθρο 332 παράγραφος 2 της Συνθήκης Λειτουργίας που αναφέρεται ακριβώς στο σκοπό της, της βελτίωσης της, της συνήθους διαδικασίας ε, έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο ενισχυμένη ε, συνεργασία, κυρίως ε, για τις χώρες μέλη οι οποίες θέλουν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια ενισχυμένη διαδικασία. Δεύτερον, θα μπορούσε να εισαχθεί μια de facto συναπόφαση μέσω ε, διαθεσμικών ε, συμφωνιών. Η Κομισιόν, ας πούμε, θα μπορούσε ε, να, να πληροφορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις προτάσεις συστάσεων και αποφάσεων ε, ε, βάσει των ε, άρθρων που αφορούν οικονομικά θέματα. Επίσης, τροπολογίες και τροποποιήσεις από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να εισαχθούν ήδη εξ αρχής στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περαίνοντας κυρία Πρόεδρε, ε, μπορώ να πω σε εσά και στα μέλη της ε, Επιτροπής σας ε, ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα ενίσχυσης των, της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια αυτής. Πρόκειται περισσότερο για θέμα πολιτικής βούλησης κατά την άποψή μου παρά ε, θέμα το οποίο περιορίζεται από τους νομικούς περιορισμούς. με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί ενισχυθεί η νομιμότητα ε, ε, και η νομική ασφάλεια. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ε, ότι περιμένω να υπάρξει και μια γόνιμη συζήτηση μετά από τις παρεμβάσεις. Πρόεδρο. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρεπαζή. Είσαστε ο πρώτος ομιλητής, οπότε να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να παρακαλέσω τους υπόλοιπους ομιλητές να ετοιμαστούν ε, και αν μπορούν να μοιράσουν τα έγγραφα με τις ομιλίες τους, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν πολλά σχόλια και πολλές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Η καθηγήτρια Μαρίζ Κρεμόνα τώρα. Έχετε όλη την Ευρώπη στο βιογραφικό σας σημείωμα με τόσα κέντρα που ασχολούνται με τις ευρωπαϊκές σπουδές, αλλά σήμερα έρχεστε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο και ως καθηγήτρια αυτού. Σας δίνω λοιπόν ευθύ αμέσω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Πρόεδρε για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Νομίζω, πρωτού προχωρήσω στις συγκεκριμένα σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ, να πω πολύ σύντομα ότι νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρη η συζήτηση σήμερα. Πέντε χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές υποθέσεις βλέπουμε μια ε, θεσμική προσαρμογή, επαναπροσαρμογή και ευθυγράμμιση σε σχέση με τα θέματα του καθορισμού των ρόλων των θεσμικών οργάνων. Τις διαθεσμικές διευθετήσεις δηλαδή. Βεβαίως δεν έχουν επιληθεί όλα τα ζητήματα. Και αυτή τη στιγμή πρέπει ακριβώς να δούμε πού έχουν φτάσει οι εξελίξεις επίσης. Να παρατηρήσω ότι οι εξωτερικές υποθέσεις είναι ένας τομέας όπου έχει πολύ συγκεκριμένε ιδιότητες η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου μπορεί να χαράξει εξωτερική πολιτική σε πολλά θέματα όπως η ανάπτυξη και το εμπόριο, να αναπτύξει σχέσεις και εταιρικές σχέσεις με χώρες που συμμερίζονται τις γενικούς στόχους της Ένωσης. Και επίσης η συνθήκη ορίζει γενικούς σκοπούς και ένα πλαίσιο. Όμως δεν καθορίζει συγκεκριμένου τελικούς στόχους, επιμέρους στόχους, όπως τη δημιουργία μιας κοινή αγοράς ή στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι. Έχουμε λοιπόν διευρυμένου εξωτερικέ αρμοδιότητες και Κατά συνέπεια έχουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια τα θεσμικά όργανα στο να ερμηνεύουν τι συνθήκε και του στόχου τη για του σκοπούς τη εξωτερική πολιτική. Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση πρέπει να αναπτυχθεί αποτελεσματικά και αποτελεσματικά επίσης να υλοποιείται. Αυτό θέλουμε να δούμε κατά πόσον μπορεί να βελτιωθεί σήμερα. Επίσης, να επισημάνω ότι η Ένωση, όπως ξέρετε, έχει ένα μια μεγάλη γκάμα οργάνων και εργαλείων στην ε, διάθεσή της για την εξωτερική της ε, δράση. Δεν υπάρχει αυτή καθεαυτή αρμοδιότητα μεν, αλλά το σύστημα εξωτερικών υποθέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, όχι μόνο ως προς τη θεσμική ισορροπία, αλλά ω και προ το ρόλο που διαδραματίζουν τα κράτη-μέλη και τα οποία παραμένουν κυρίαρχα στη χάραξη της εξωτερικής τους πολιτικής. Υπάρχουν λοιπόν τα εργαλεία, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο ώστε να είναι συμβατά με τη συνθήκη και επίσης αποτελεσματικά. Και αυτό δεν είναι πάντοτε κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν ιδίω τη διάρθρωση τη δράση τη Ένωση ε, ω προ τη δράση των κρατών μελών. Αυτό πάντοτε αποτελεί, μπορεί να είναι αντιφατικό και ο νόμος, το δίκαιο μπορεί να είναι ε, κάτι που να δημιουργεί δυσκολίε ω προ την ερμηνεία παρά να διευκολύνει τα πράγματα και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για δικηγόρου και νομικού όπω εγώ ίδια. Γι' αυτό θα ήθελα να επικεντρωθώ σε μερικά συγκεκριμένα σημεία εντάχει, ξεκινώντα από τι διεθνεί ε, συμφωνίε έχω διαχωρίσει την παρουσίασή μου σε τομείς αρμοδιότητας σε πρώτη φάση και μετά σε διαδικασίες ως προς τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. Σε ό,τι αφορά τους τομείς ε, δράσης, η συνθήκη της Λισαβόνας σκοπό είχε να δημιουργήσει ένα σύστημα αρμοδιοτήτων ε, και το πώς αυτές εκχωρούνται βάσει των διατάξεών της και αυτό σε έναν βαθμό έχει επιτευχθεί. Αυτό που είδαμε να συμβαίνει στην πράξη Κάτι που δεν αναμενόταν αναγκαστικά ως αποτέλεσμα της θέσης της συνθήκης είναι η αυξημένη χρήση κάποιων βασικών ε, νομικών βάσεων με ευρεία ε, κάλυψη για την ε, σύναψη διεθνών συμβάσεων όπως η εμπορική πολιτική, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και η... το τομέα της ΚΕΠΑ. Εδώ βλέπουμε κάποιες υποθέσεις βέβαια να φτάνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της ευρείας ερμηνείας όλων αυτών των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά, τα αναπτυξιακά και ακόμη και για την ΚΕΠΑ θα έλεγα. Εδώ πρέπει να προσθέσω ότι το δικαστήριο συνεχίζει να δείχνει μια, βάση, μια σαφή προτίμηση για μια ευρία νομική βάση σε ό,τι αφορά τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. Και αυτό έχει επιπτώσεις ιδίως στην ε, ΚΕΠΑ και θα ήθελα να σταθώ αργότερα σε αυτό. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι όλο ένα και περισσότερο να χρησιμοποιούνται λιγότερες και εκπεφρασμένες αρμοδιότητες που εκχωρούνται από τη συνθήκη και δεν θέλω να υπερβάλλω αλλά σε κάποιο βαθμό Υπάρχει μια περιθωριοποίηση των ε, αρμοδιοτήτων που μέσω πλην σαφώς ε, προκύπτουν από την συνδική όπως ε, για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. Αυτό δεν δημιουργεί αναγκαστικά προβλήματα, όμως ενδέχεται να έχει θεσμικές επιπτώσεις ως προς την επιλογή της νομικής βάσης. Άρα, θεωρώ ότι το θέμα είναι πως εξελίσσεται στην πράξη η αναγνώριση όλων αυτών των ε, στοιχείων. Θα επανέλθω σε κάποιες από τις επιπτώσεις που μπορεί να προκύπτουν και που καλό θα ήταν να διερευνηθούν περαιτέρω. ό,τι αφορά τη διαδικασία για τη σύναψη συμφωνιών, λοιπόν, η συνθήκη της Λισαβόνας ενοποιεί τη διαδικασία για την ε, διαπραγμάτευση και τη σύναψη διεθνών συμφωνιών και βελτιώνει τη συνεκτικότητα του συστήματος. Δύο-τρεις παρατηρήσεις ως προς αυτό. Ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου βεβαίως. Μια αλλαγή μείζωνος σημασίας είναι ότι σε πολλές ε, συμφωνίες, όπως τις συμπορικές, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου και σχετική απέτηση για να συναυθεί η συμφωνία. Να γνωρίζετε επίσης η ανάγκη να ενημερώνεται για όλα τα στάδια της διαδικασίας του Ευρωκοινοβουλίου. Θα γνωρίζετε καλύτερα από μένα πόσο καλά αυτό λειτουργεί στην πράξη. Καταλαβαίνω ότι δυσκολίες υπάρχουν ω προς την υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης και τη διάταξη. όμως είναι μια αλλαγή μείζωνο σημασία. Γι' αυτό που θα ονομάζαμε νοοτροπία ε, και τα η ως προς την ε, σύναψη και τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών. Να υπογραμμίσω κάποια συγκεκριμένα θέματα ως προς τη διαπραγμάτευση συμφωνιών που έχουν ιονή νομοθετικό ή θεσμικό χαρακτήρα. Το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι το TTIP βεβαίω, η Συμφωνία Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης. Εδώ θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και άλλες περιπτώσεις όπως η Συμφωνία Άκτα είναι τέτοιου είδους συμφωνία. Νομίζω το πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι η διαδικασία για την κοινοβουλευτική συμφωνή γνώμη στο τέλος της διαδικασίας. Εκεί δεν είναι και ιδανικό το σύστημα. Γιατί δεν αντικατοπτρίζει σωστά την τακτική νομική, νομοθετική διαδικασία όπου το κοινοβούλιο ουσιαστικά διαμορφώνει και επηρεάζει τις νομοθετικές πράξεις με την τοποθέτησή του. Νομίζω ότι πρέπει να μελετήσουμε καλύτερα ε, το όλο θέμα και μάλιστα με δημιουργικό τρόπο για να δούμε πώς μπορούμε να καλέσουμε το Κοινοβούλιο να συμμετέχει περιττέρω. Ε, κάτι που και προηγουμένως υπόθηκε για την δημοκρατική λογοδοσία. Πώς μπορεί να υπάρχει μια πιο διαβριμένη συζήτηση στο επίπεδο του Κοινοβουλίου, στα πρώτα στάδια διαπραγμάτευση μια διεθνή συμφωνία. Ιδίω όπου η συμφωνία, εκεί όπου η συμφωνία μπορεί να έχει τρόπον τεινά νομοθετική ή θεσμική την υπάρχουν ενδείξεις ότι η δημοσίευση τη εντολή για το ΔΤΠ είναι κάτι προ αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα μπορούσε να γίνουν και περισσότερα. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι κάπως ίσως πιο εσωτερικού χαρακτήρα και είναι μάλλον το πώς οι αποφάσεις που ε, καθορίζουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φορείς που ιδρύονται βάσει διεθνούς συμφωνίας ε, διαμορφώνονται σε περίπτωση που οι φορείς αυτοί μπορεί να εγκρίνουν πράξεις με νομικές συνέπειες. Οι φορείς όπως ιδρύονται ή δημιουργούνται ε, λόγω ε, διεθνών συμφωνιών μπορεί να έχουν νομικές επιπτώσεις. Εκεί πώς διαμορφώνεται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι διαδικασίες προβλέπονται σχετικά. Η διαδικασία τι διαδικασιε προβλεπονται σχετικα από το άρθρο 218 εδάφιο 9 με μια απλουστευμένη μορφή της διαδικασίας για την σύναψη διεθνών συμφωνιών. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια δεν είναι συμβαλόμενο μέρος της συμφωνίας, αλλά όπου η συμφωνία επιπτύσσει την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε τα κράτη-μέλη καλούνται να ε, γκρίνουν μια θέση εκ μέρους της Ένωσης πρέπει να οριστεί μια επί της ουσίας νομική βάση για τις διαδικασίες αυτές. Όμως η βάση για τη διαδικασία θα είναι το άρθρο 218 εδάφιο 9 με την ενισχυμένη ψηφοφορία, με την ψηφοφορία μάλλον ενισχυμένη πλειοψηφία στο ε, Συμβούλιο και με παρουσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμη και αν είναι νομική η βάση προβλέπει ομοφωνία, υποχρέωση ομοφωνία, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει άλλη υποχρέωση παρά μόνο το να τηρείται ενήμερο καθ' όλα τα στάδια τη διαδικασία. Οι διαδικασίε αυτέ, οι αποφάσει μάλλον αυτέ, πολλέ φορέ έχουν να κάνουν με ζητήματα που δεν είναι απλώ εθνικού χαρακτήρα, αλλά έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Και ενώ καταλαβαίνω απολύτω την ανάγκη τη απλουστευμένη διαδικασία σε τέτοιε περιπτώσει, δεν είμαι πεπισμένη ότι υπάρχει η, απαραίτητη, η σωστή ισορροπία. Τουλάχιστον προ στιγμή. Νομίζω ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε Το ΠΑΣ θα μπορούσε η ψηφοφορία στις ενισχυμένη πλειοψηφία να σταθμιστεί διαφορετικά. Και ίσω να υπάρχει και μια ε, διαδικασία διαβούλευση για να εξασφαλίζεται η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το τρίτο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ έχει να κάνει με τι μεικτέ συμφωνίε. Μεικτέ, εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι όλοι συμπαλωμένα μέρη. Ε, είναι μια πραγματικότητα πολύ συχνά, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην ε, συνθήκη για τη σύναψη τέτοιου είδου διεθνών συμφωνιών. Υπάρχει ένα βαθμό ευελιξία που προβλέπει η συνθήκη τη Λισαβόνα στο 218 για την έννοια, με την έννοια της διαπραγματευτικής ομάδας της Ένωσης. Εκεί θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα η διάταξη αυτή, προκειμένου να διαρθρωθούν καλύτερα οι ενδεχόμενοι σχηματισμοί τη διαπραγματική ομάδα τη Ένωση σε περίπτωση διαπραγμάτευση τέτοιου είδου συμφωνιών. Όμω αυτή η ευελιξία είναι πιο περιορισμένη σε ό,τι αφορά την απόφαση που προβλέπει την υπογραφή ή την σύναψη τη ε, συμφωνία, την τελική σύναψη. Πρόσφατα υπήρξε απόφαση από το ΔΕΚ όπου θεωρήθηκε ότι οι βρυδικές αυτές αποφάσεις, οι αποφάσεις που συνδυάζουν και την Ένωση και τα κράτη-μέλη που συνεδριάζουν στο Συμβούλιο με τους εκπροσώπους τους, αυτό είναι μια παραβίαση της συνθήκης. Οπότε θα μπορούσε να διευκολύνει το να σκεφτούμε τη δυνατότητα προσθήκη στην όλη διαδικασία λήψη αποφάσεων για τις διεθνείς συμφωνίες κάποιων, ε, κάποιων διατάξεων που να διευκολύνουν αυτή την ε, σύναψη τέτοιου είδους συμφωνιών. Να προχωρήσω στο θέμα της κοινή εξωτερικής πολιτικής ε, ασφάλειας. Ξέρουμε ότι αυτή η πολιτική υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες και κάποιες από τις αλλαγές που ε, εισάγει η συνθήκη της Λισαβόνας ε, καθορίζουν τα όρια μεταξύ της ΚΕΠΑ και άλλων εξωτερικών δράσεων της Ένωσης. Είναι απαραίτητο, αν και πιο δυσκερές, να εφαρμοστούν όλα αυτά με τρόπο απλό. Και θα μπορούσα να προχωρήσω σε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια της συζητησή μας. Όμως, το σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει ακόμη ανάγκη να οριοθετήσουμε την ΚΕΠΑ σε σχέση με τις εξωτερικές δράσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της ΚΕΠΑ. Εδώ θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Εάν λάβουμε υπόψη τον τρόπο που το δικαστήριο ε, ορίζει το θέμα των νομικών βάσεων. Δηλαδή, μπορεί η νομική βάση που έχει επιλεγεί να αιτιολογηθεί. Και αν λάβουμε υπόψη την προτίμηση του δικαστηρίου για μία ενιαία, μία και μόνη νομική βάση, ε, καθίσταται σαφές ότι εφόσον έχει επιλεγεί η νομική βάση της ΚΕΠΑ από την Επιτροπή και το Συμβούλιο τότε είναι πολύ δύσκολο να ε, αμφισβητηθεί η συγκεκριμένη επιλογή. Επίσης φαίνεται ότι η ΚΕΠΑ, ως γνωρίζουμε, ενδεχομένως μπορεί να είναι πολύ ευρεία στην ερμηνεία της. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι ΚΕΠΑ. Δεν υπάρχουν σαφή όρια στις δράσεις της ΚΕΠΑ. Νομίζω ότι αυτό έχει ως συνέπεια την περιθωριοποίηση όλος ιδίως των εξωτερικών διαστάσεων της ε, δικαιοσύνης και των ιστορικών υποθέσεων που έχουν να κάνουν ακριβώς με τα θέματα της αστυνομικής συνεργασίας. Είναι πολύ δύσκολο πάντως να έχει επιλογή νομική βάση για την ε, εξωτερική πολιτική που έχει να κάνει με την ασφάλεια και μετά να αμφισβητηθεί, όπως ε, οι συμφωνίες που έχουν να κάνουν με την τρομοκρατία ή με τον Μαυρίκιο για την ε, μεταφορά υπόπτων ή το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων για άτομα που πρόκειται να δικαστούν στην Αίγυπτο για περιπτώσεις υπεξαίρεσης ε, δημοσίων πόρων. Εδώ η νομική ε, βάση αμφισβητήθηκε και τελικά το δικαστήριο συμφώνησε με την αρχική επιλογή. Είναι δύσκολο λοιπόν να οριοθετήσουμε σωστά τον ρόλο το συγκεκριμένο σημείο πρέπει να τοποθετηθεί η ΚΕΠΑ στην εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του νομικού οικοδομήματο ε, που έχουμε αυτή τη στιγμή ό,τι αφορά τι διεθνεί συμφωνίε. Τώρα η δυνατότητα μια κοινή νομική βάση προβλέπεται, αλλά σπανίω ε, αξιοποιείται. Έχει χρησιμοποιηθεί κάποιε φορέ, αλλά όχι συχνά. Ίσως μια καλή ιδέα θα ήταν να αποσαφινιστεί ότι η νομική δυνατότητα υπάρχει και ότι μπορούμε να την αξιοποιούμε συχνότερα. Σε ό,τι αφορά τις αυτόνομες δράσεις και πράξεις, η συνθήκη λειτουργίας ε, θα έπρεπε να προβλέπει μια τακτική διαδικασία. Ε, το δικαστήριο ε, θεωρεί ότι η κοινή νομική βάση σε αυτές περιπτώσεις δεν είναι μια επιλογή δυνατή. έχουμε λοιπόν ένα ζήτημα που πρέπει να επιληθεί εδώ. Και θα πρέπει να σκεφτούμε τι ρόλο έχει εδώ και το δικαστήριο της Ένωσης, την ΚΕΠΑ. Και θα σταθώ σε κάτι που είπε ο κύριο Μπροκ προηγουμένω. για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτά ήταν από τα βασικά εμπόδια που ε, βρήκε το δικαστήριο για την προσχώρηση και νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. κατά πόσον το δικαστήριο μπορεί να ασχοληθεί με την δικαστική εξέταση κάποιων πράξεων που έχουν ήδη αποφασιστεί για την ΚΕΠΑ. Θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου σε αυτή τη φάση, τις αρχικές μου τουλάχιστον παρατηρήσεις, μια, με ένα τελικό σχόλιο. Έκκληση να ε, σκεφτούμε λίγο ε, εκτός ε, των συνηθισμένων μας απόψεων το κατά πόσον μπορεί να υπάρχει συνένεση στις αποφάσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική. Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα κατά πόσο μπορούμε να ετοιμάζουμε έγγραφα στρατηγικού χαρακτήρα, στρατηγικέ πρωτοβουλίε που να υιοθετούνται από κοινού από τα θεσμικά όργανα. Βεβαίω υπάρχει περιθώριο για το Κοινοβούλιο να έχει τις δικές του αυτόνομες δράσει, ψηφίσματα, αποφάσεις, εκθέσει. Όμως αυτά που από κοινώ εγκρίνονται και έχουν στατοκικό χαρακτήρα για βασικά θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τέτοιου είδους έγγραφα θα ήταν μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Όχι αναγκαστικά τρομερά καινοτόμα, αλλά αυτήν την δυνατότητα θα πρέπει να την εξερευνήσουμε περαιτέρω. Και εκεί σίγουρα δεν θα χρειαστεί και αναπροσαρμογή της συνθήκης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κρεμόνα. Συνήθως δεν χειροκροτούμε. Μη θεωρείτε ότι δεν μας άρεσαν αυτά που είπατε ή δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά δεν συνηθίζεται. Να περάσουμε τώρα στον ε, Δ. Σέρζιο Καρέρα από το Κέντρο Ευρωπαϊκών ε, Σπούδων Πολιτικής, ε, το ΣΕΠΣ, έχετε το λόγο. Θα αναφερθείτε σε θέματα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, από ό,τι κατάλαβα. Good morning. I have a PowerPoint Καλημέρα σας. Έχω μια παρουσίαση σε PowerPoint. Τα θαύματα της τεχνολογίας. Α, ορίστε. Τα καταφέραμε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Καλημέρα σε όλους. Ε, είναι χαρά μου να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να σταθώ σε κάποια ουσιαστικά ζητήματα και κάποιες προκλήσεις ε, που εξετάζουμε όταν εξετάζουμε πολιτική δικαιοσύνη και ιστορικών υποθέσεων. Ίσως θα έπρεπε να τα σκεφτούμε λίγο περισσότερο εν ώψη και των μελλοντικών ε, ε τροποποίησεων της συνθήκης. Στην παρουσίασή μου θα σταθώ σε τέσσερα σημεία. Καταρχάς θα σας δώσω λίγο το υπόβαθρο, ε, το ιστορικό για τις πολιτικές δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων. Στη συνέχεια θα περάσω στις ε, βασικές καινοτομίες που έφερε η συνθήκη της Λισαβόνας στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Κατόπιν θα σταθώ στις βασικές προκλήσεις, ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το παρόν πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας και το κατά πόσον θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και στη συνέχεια θα δώσω και κάποια ε, τροφή για σκέψη για μελλοντικέ προσαρμογές. Επίσης να σας ε, ε, ενημερώσω ότι το κέντρο μας, το ΣΕΠΣ, ετοιμάζει μια νέα μελέτη που ζήτησε η Επιτροπή σας και εξετάζει ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν προκαταρκτικές απόψεις. Όσο θα εμβαθύνουμε στην έρευνά μας θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Ε, λίγα πράγματα για το ιστορικό. Η δικαιοσύνη και ο ιστορικό υποθέσει ε, μπορεί να είναι ένα πολύ τεχνικό ζήτημα, αλλά περιλαμβάνει πάρα πολύ σημαντικούς και ε, ιδιαίτερους τομείς. Μετανάστευση, τρομοκρατία. Τα τελευταία 30 χρόνια η συνεργασία αυτή, παρά το γεγονός ότι είναι ευαίσθητη, ήταν ιδιαίτερα δυναμική. Έχουμε ένα σαφές νομικό πλαίσιο και ένα πλαίσιο πολιτικής, το οποίο έχει αναπτυχθεί σιγά σιγά και έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένε ε, πολιτικές. Η δικαιοσύνη και οι ιστορικέ υποθέσει χαρακτηρίζεται από μια σειρά από ελλείψει. Είναι μια μορφή συνεργασία ε, την οποία υποσκάπτει η λογοδοσία, η ε, μυστικότητα και το γεγονός ότι εκφύσεως κάποια ζητήματα είναι εμπιστευτικά. Ε, ξέρουμε ότι έχουμε θέματα στους διάφορους πυλώνες μεταξύ του πρώτου και του τρίτου πυλώνα. Αυτό βασικά σημαίνει αυτό. Αδιαφάνεια, έλλειψη ε, ε λογοδοσία στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και επίση σημαίνει ότι το Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Ιστορικών Υποθέσεων ε, έχει τα ενία της λήψης αποφάσεων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε κανένα ρόλο να διαδραματίσει. Το δικαστήριο είχε πολύ περιορισμένο ρόλο στην ερμηνεία και την αξιολόγηση της ε, ε, εγκυρότητας των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο σημαίνει ότι μέχρι πρόσφατα υπήρχε έλλειμμα δημοκρατίας και δικαιοσύνης στον τομέα αυτό. Η συνθήκη της Λισαβόνας άλλαξε τα πράγματα αυτά προς το καλύτερο. Καταρχάς ε, δεν έχουμε πλέον αυτούς τους πυλώνες ε, στην δικαιοσύνη και στις υποθέσεις και τουλάχιστον επισήμως έχει ε, επεκταθεί η κοινοτική μέθοδος συνεργασίας. Υπάρχει πλέον ένα τίτλος, ο τίτλος 5, που περιλαμβάνει όλους αυτούς τους τομείς και έχουμε τα συγκεκριμένα κεφάλαια τα οποία αφορούν ε, ε, ελέγχου σύνορους, μετανάστευση, άσυλο, ε, δικαστική συνεργασία σε ποινικά και αστικά ζητήματα και σε εγκλήματα, καθώς επίσης και αστυνομική συνεργασία. Επίσης υπάρχει το δεύτερο τμήμα της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει την ηθαγένεια και τη ρήτρα μη διάκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης δόθηκε και δεσμευτική ισχύ ε, στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που φυσικά είναι γενή σε όλες αυτές τις πολιτικές. Σα ανέφερα προηγουμένω, ότι πέραν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα, ε, συγγνώμη, πριν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα, το Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Εσωτερική ε, Υποθέσεων είχε τα ημεία. Αυτό μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα άλλαξε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτη στι ε, ε, τομεί, αυτούς τομείς. Έχει ενισχυθεί και ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΕΚ έχει πλέον πλήρη δικαιοδοσία να αναθεωρήσει και να ερμηνεύσει νομικέ πράξει χωρίς φυσικά να λησμονούμε και τη δράση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, που ε, είναι σημαντικός παράγων πλέον στους τομείς αυτούς. Το τέλος του 2014 ήταν πολύ σημαντική στιγμή, διότι τελείωσε η μεταβατική περίοδος των 5 ετών από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας Μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο είχαν περιορισμένες εξουσίες για την αναθεώρηση και τον έλεγχο των ε, κρατών μελών και το κατά πόσον τήρουν τις, προ... τις υποχρεώσεις τους. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα και τώρα υπάρχουν πλήρες δυνατότητες εφαρμογής. Το Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρακολουθεί ε, την εφαρμογή ε, από πλευράς ε, αρχών επιβολής του νόμου και αστυνομίας και επομένως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Επίσης αλλάζουν και οι διάφορες ε, συνθέσεις ε, ε, στις μελλοντικές εξελίξεις. Ωστόσο, και αυτό αναφέρθηκε και στο παρελθόν, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικέ υποθέσει είναι ένα ιδιαίτερο τομέα γιατί επιτρέπουν ευελιξία και διαφοροποίηση. Κάτι το οποίο μας οδήγησε σε αρκετές συζητήσεις, όπως για παράδειγμα η ρήτρα opt-out, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το πρώτο, αλλά όχι μόνο, και η Ιρλανδία έχει αυτή τη δυνατότητα. Και η Ιρλανδία μάλιστα διεύρυνε και αυτές τις δυνατότητες για να μην καλύπτει όχι μόνο θέματα συνόρων και μετανάστευσης, αλλά θέματα και ποινική δικαιοσύνη και αστυνομία. Και αυτό το μεταβατικό πρωτόκολλο που σας ανέφερα, το πρωτόκολλο 36, επιτρέπει και στο Ηνωμένο Βασίλειο να πει ή να επιλέξει να μην συμμετέχει σε οποιοδήποτε ε, μέτρο ε, ποινικής δικαιοσύνης και ε, τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να συμμετέχει σε 36 μέτρα ποινική δικαιοσύνη. Και αυτό ενισχύει αυτό το οποίο ανέφερε προηγουμένω κάποιο από του εισηγητέ. Κατά πόσον είναι ακόμα εφικτό, κατά πόσον υπάρχει ακόμα δυνατότητα από πλευρά Ηνωμένου Βασιλείου να επιλέγει να συμμετέχει να μην συμμετέχει όταν εμεί προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό τομέα δικαιοσύνη σε ποινικά ζητήματα. Η δεύτερη πρόκληση που μα έφερε η συνθήκη τη Λισαβόνα είναι η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση σε ευαίσθητου τομεί εθνική κυριαρχία. Καταρχά υπάρχει δυνατότητα να έχουμε αυτέ τι ρήτρε ε, ε, break, δηλαδή να έχουμε επίγοντα μέτρα σε κάποιου τομεί ποινική δικαιοσύνη ή σε κάποια ε, ποινικά αδικήματα και κυρώσεις και σε κάποιες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη αν θεωρούν ότι η έγκριση μιας νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας θα πλήξει σημαντικές πτυχές του ποινικού του συστήματος τότε μπορούν να πούν ότι θα πρέπει να σταματήσει η συνήθις νομοθετική διαδικασία και ε, να υπάρξει μια παύση για να εξετάσουμε ε, προσεκτικά όλες αυτές τις διαδικασίες. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο ε, διαφοροποίησης είναι η δυνατότητα ενισχυμένης συνεργασίας. Και εδώ έχουμε τρεις τομείς που βλέπετε στη διαφάνεια. Ε, ποινική δικαιοσύνη, ποινικά δικήματα και ο Ευρωπαίος εισαγγελέα. Ε, κάτι το οποίο πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά, διότι μπορεί να γίνει μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που θα έχουμε στο μέλλον στη δικαιοσύνη και στις εταιρικές υποθέσεις. Εδώ υπάρχει δυνατότητα εννέα κράτη-μέλη να ε, προχωρήσουν ως μια μικρή ομάδα ενισχυμένης συνεργασίας. Ποιες είναι οι προκλήσεις όμως. Έχουμε αποτελέσματα από την συνθήκη της Λισαβόνα. Έχουμε αυτές τις εξαιρέσεις, έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Ποιες είναι οι προκλήσεις που ε, ε, απομένουν. Καταρχάς, η διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμόρφωση των αποφάσεων. Ναι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης, καθορίζει και την πολιτική στον τομέα αυτό, αλλά πώ λειτουργεί αυτό στην πράξη. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν αλλάξει πραγματικά άποψη όταν συζητούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, αντιμετωπίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτη σε καθημερινή βάση. Και εδώ υπάρχουν κάποια παραδείγματα που μας δείχνουν ότι δεν ισχύει ε, ακόμα πλήρως. Προηγουμένως ε, αναφέρθηκε το θέμα των διεθνών συμφωνιών. Η Διεθνή Συμφωνία είναι εξαιρετικό παράδειγμα ε, ως προς τα προσκόμματα που αντιμετωπίζονται και το γεγονός ότι δεν συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευθύς εξ αρχής στη σύναψη και στις εξελίξεις της Διεθνής Συμφωνίας και αυτό υπήρξε ε, επίμαχο ζήτημα και στη δικαιοσύνη και στις εξωτερικές υποθέσεις και φυσικά στη συμφωνία με τις Ηνωμένες όταν εξετάζουμε πώς ε, λειτουργεί η συνήθις νομοθετική διαδικασία στην πράξη, ε, αντιμετωπίζονται μια σειρά από προβλήματα, τα οποία ίσως θα πρέπει να εξεταστούν όταν ε, σχεδιάζουμε τη μελιγενίστη. Καταρχάς, συμφωνία σε επίσημους τριμερείς διαλόγους. Πώς λειτουργεί αυτό. Υπάρχει κατάλληλη λογοδοσία και συζήτηση των πολύ σημαντικών ε, ε, κάποιων θεμάτων σε κάποιες περιπτώσεις, αποφάσεις ή τροπολογίας. Υπάρχουν ακόμα θέματα διαφάνειας και ίσως αυτό πρέπει να τα εξετάσουμε περαιτέρω. Μια δεύτερη πρόκληση συνέπεια και συνεκτικότητα ή μάλλον έλλειψη ε, συνεκτικότητας μετά από αυτή τη διαφοροποίηση και κάποιες ρήτρες ευελιξίας. Υπάρχει ένας κοινό τομέα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ε, εσωτερικών υποθέσεων ή ε, υπάρχει ένας φαύλος κύκλος και ζούμε μαζί και χώρια ταυτόχρονα σε μια σειρά από πολιτικές που έχουν συνέπειες για όλους και φυσικά για την ελευθερία και τις ελευθερίες όλων. Τη δυνατότητα να υπάρχουν εξαιρέσει. Ε, η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, για παράδειγμα, είναι εξαιρετικό παράδειγμα. Υπάρχουν κάποιε αντιρρήσει από κάποια κράτη-μέλη ε, και θεωρείται ότι μπορεί να περιορίζεται η δημοκρατική λογοδοσία από πλευρά ε, κοινοβουλίων σε σημαντικού τομεί πολιτική, παραδείγματο χάρη στην τρομοκρατία. Κράτο δικαίου. Η Ουγγαρία είναι εξαιρετικό παράδειγμα ε, χρησιμοποιείται πολύ συχνά το επιχείρημα ότι αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα και εσείς δεν έχετε καμία αρμοδιότητα. Και πλέον ε, είναι σπάνιο η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει. Και επίσης υπάρχει το εξή ερώτημα. Αυτές οι αρχές οι οποίες είναι γεγραμμένες στη συνθήκη της Λισαβόνας τίθεται σε εφαρμογή στην πράξη. Ε, στον τομέα της μετανάστευσης, αλληλεγγύη και καταμερισμός ευθυνών. Αυτό περιλαμβάνεται στο άρθρο 80 της συνθήκης. Πώς εφαρμόζεται στην πράξη αυτή ε, η αρχή. Δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγή της συνθήκης, αλλά πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη αυτές οι αρχές. Κάτι αντίστοιχο, αξιολόγηση πολιτικών που ε, είναι ήδη καθιερωμένες. Ε, ποινική δικαιοσύνη και δικαιώματα των ε, θυμάτων στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική πολιτική στην οποία υπάρχουν ε, αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς εφαρμόζεται αυτό στην πράξη. Τα κράτη-μέλη πώς εφαρμόζουν ε, το Ευρωπαϊκό Έγκλημα Σύλληψης, ε, τι γίνεται με τα δικαιώματα των υπόπτων και την οδηγία που σχετίζεται με αυτό. Δεν γνωρίζουμε στην πράξη πώς εφαρμόζονται. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτό δεν είναι μόνο... Ε, θεωρητικό, υπάρχουν σημαντικά ε, συνέπειες του τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι προκλήσεις που ανέφερα προηγουμένως έχουν σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα των ε, ε, Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες στην πραγματικότητα βρίσκονται ενώπιον καταμερισμένων τομέων δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων. Ανεξάρτητα από πού βρίσκεσαι, έχεις, θα έπρεπε να έχεις τα ίδια δικαιώματα, ενώ έχεις διαφορετικά δικαιώματα. Και αυτό θα έπρεπε να ανησυχεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η διαφοροποίηση και αυτή η ενισχυμένη συνεργασία έχει συγκεκριμένες συνέπειες για τις διακρίσεις και την ίση μεταχείριση των Ευρωπαίων πολιτών. Και επίση. ο Ευρωπαϊκός Χάρτης ίσως ακολουθεί τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πώς ακολουθεί ε, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στις διοργανικές σχέσεις ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Δικαιωμάτων. Τελευταία μου διαφάνεια. Μελλοντικέ προσαρμογές. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τρεις προκλήσεις. Καταρχάς, Θέλουμε περισσότερη εργοδοσία, ε, δημοκρατία και διαφάνεια στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Και θα πρέπει να είναι προτεραιότητα να εφαρμοστούν στην πράξη αυτές οι αρχές. Ε, το άσυλο είναι εξαιρετικό παράδειγμα. Υπάρχει ολόκληρη συζήτηση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ε, ποσοστώσεις για την μετεγκατάσταση των ε, τον άσυλο πολλές χώρες εξέφρασαν διαφωνία για αυτές τις ποσοστώσεις. Αλλά πώς θα εφαρμοστεί αυτή ως ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Διότι το σύστημα του Δουβλίνου δεν έχει αποτέλεσμα, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις από αυτού, δεν λειτουργεί το σύστημα του Δουβλίνου, επομένως πώς θα εφαρμόσουμε την αλληλεγγύη, πώς θα υπάρξει κατάλληλος καταμερισμός των ευθυνών. Και τέλος, ε, Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο και ίσως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε εδώ να διαδραματίσει κάποιο ρόλο για να διασφαλίσει ότι θα υπάρξει ένας εξορθολογισμός του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καρέρα. Έχουμε μισή ώρα τώρα για τη συζήτηση. Και ξέρω ότι έχουμε και έναν πρόσωπο της ΕΟΚΕ και τον πρόεδρο της ομάδας 3, ε, τον Λούκα Γιάχερ. Ε, κύριε Γιάχερ, θέλετε να λάβετε το λόγο. Και μετά είναι ο Γιώ Λάιεν ε, μόνο εγγεγραμμένο στον κατάλογο των ομιλητών. Αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο να μας το πει. Κύριε Γιάχερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρχάς επιτρέψτε μου εξ ονόματος του Προέδρου και όλων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής να σας ευχαριστήσω και για την ευκαιρία που μου δίνετε να λάβω εδώ το λόγο κατά τη διάρκεια της παρούσα ακροάσεως, αλλά σας ευχαριστούμε και που μας ρωτήσατε και όλα στη γνώμη μας για τις δύο εκθέσεις πρωτοβουλίας των εισηγητών. Είχα την τιμή να με ορίσει το Προεδρείο της Επιτροπής μας εισηγητή ε, πριν από δύο εβδομάδες και παρά το καλοκαίρι. Μέσα Σεπτεμβρίου αναμένουμε να εγκρίνουμε τη γνωμοδότησή μας. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία αυτή που ανοίξατε στην Επιτροπή σας και άκουσα τα σημαντικότερα στοιχεία που εξέθεσαν οι τρεις εισηγητές. Σίγουρα είναι πολύ πρόσφορη αυτή η συγκυρία για να ξαναρχίσει η συζήτηση. Ε, χρειάζεται ένα μείγμα ρεαλισμού και φιλοδοξίας. Είτε ε, να δούμε τι μπορούμε να ξανανοίξουμε, είτε να δούμε τι ε, δυνατότητες έχουμε στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είναι πραγματικά πρόκληση και ενδιαφέρουσα πρόκληση. Σε αυτή την πρώτη μου παρέμβαση λοιπόν θα ήθελα να ε, αναφερθώ στην οικονομική διακυβέρνηση, κυρίως στην ΟΝΕ, γιατί είναι πολλά τα θέματα και λίγος ο χρόνος. Και να ε, πω ότι υπάρχει ανάγκη να εμβαθύνουμε στην κοινωνική διάσταση ε, των κειμένων συνθήκων. Επανειλημμένως έχουμε πει στην Επιτροπή μας ότι το σύστημα διακυβέρνησης της ΟΝΕ έχει φτάσει στα όρια του. Υπάρχουν όρια δημοκρατίας και λογοδοσίας. Καμιά φορά όμως και αποτελεσματικότητας λόγω των ισχυρών, των διαφόρων ε, πιέσεων, ε, των πολλών οργάνων και των πλαισίων ε, λήψης αποφάσεων. Και ε, ακριβώ επειδή υπάρχουν αυτές οι κακοφωνίες, καμιά φορά είναι σημαντικές οι παρανοήσεις και οι παρεξηγήσεις απέναντι στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και στη συντεταγμένη πολιτεία θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τα διάφορα ε, νομοθετήματα που διέπουν την οικονομική διακυβέρνηση. Τούπακ, ε, ΣΥΚΣΠΑΚ, Τραπεζική Ένωση, όλα αυτά έγιναν σε επίπεδο διακυβερνητικό και δεν επέτρεψαν να ε, συμμετέχει όλη η κοινωνία στην επίλυση της κρίσης και ταυτόχρονα αυξήθηκαν οι καχυποψίες και δυσπιστίες των κοινωνιών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας λοιπόν χρειάζεται να χτίσουμε μια σύγκληση μεταξύ των διαφόρων κρατών στην Ευρωζώνη για να περάσουμε από το σημερινό σύστημα απλού συντονισμού σε ένα πιο σημαντικό σύστημα συναπόφασης για τα βασικά της μακροοικονομικής και μικροοικονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό θα πρέπει να επανέλθουμε στην ε, κοινοτική μέθοδο για την οικονομική διακυβέρνηση, να ζητήσουμε να έχουν ισχυρότερο ρόλο εθνικά και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και διαφοροποιημένη ένταξη. Ε, το περίφημο μοτίβο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δύο ταχυτήτων. Επίσης ένας μηχανισμός αναδιανομής χρειάζεται στην Ευρωζώνη και ένας γνήσιος προϋπολογισμός της Ευρωζώνης. Χρειάζεται ένα νέο άλμα λοιπόν ε, για να δοθεί μια νέα πνοή στην ΟΝΕ, όχι μόνο ευθύνη, ε, λογοδοσία, δημοκρατία, διαφάνεια, αντιπροσωπευτική νομιμότητα και δημοκρατική για να υπάρξει και ένας ουσιαστικός κοινωνικός πυλώνας. Υπό την έννοια αυτή έχουν ε, παραμεληθεί σε μεγάλο βαθμό δύο άρθρα. Το άρθρο 9 για τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει να κάνει με την πλήρη απασχόληση ως προοπτική και την κοινωνική προστασία και το άρθρο 3 στο σύνολό του που η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στα οικονομικά ζητήματα και στην ε, κοινωνική και δαφική συνοχή. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι τον Ιούνιο του 2014 έχει λάβει ε, δεσμεύσει στο Συμβούλιο και ε, έχει χαράξει και γραμμέ με τι οποίε συμφωνούμε πάρα πολύ. Μια ένωση δηλαδή της απασχόλησης, της ανάπτυξης πρέπει να προωθηθεί και να δίνει σε όλου του πολίτες τη δυνατότητα να υλοποιούν τα, τις προσδοκίες τους και να ε, προστατεύονται. Άλλα άρθρα 151-153 έχουν ως προορισμό να υποστηρίξουν ε, μια ε, αηφόρο ανάπτυξη των κρατών μελών και βιώσιμη. Χωρίς να λησμονούμε ε, το χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων που είναι πολύ σημαντικός για τους πολίτες μας. Στα πλαίσια της κείμενης συνθήκης λοιπόν υπάρχουν πολλές δυνατότητες και μέσα. Θα πρέπει να υπάρξουν σε πρώτη φάση κοινωνικοί δείκτες ε, δεσμευτική και παρακολούθηση της κοινωνικής εξέλιξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Να υπάρξει ένα νέο και μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής δράσης, τουλάχιστον στην Ευρωζώνη, για να μην μπω σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερη προστασία των κοινωνικών συστημάτων, ε, πιο στοχευμένες κοινωνικές δράσεις και ε, μεγαλύτερη έμφαση στην ε, ε, βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Ολοκληρώνω. Θα πρέπει με τρόπο πιο αποτελεσματικό να εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας και να αναδεικνύεται καλύτερα η συνεχής αυτόνομη συνεισφορά της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών σε κοινοτικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό και αυτοδιοικητικό. Θα πρέπει όλες οι πολιτικές να λαμβάνουν υπόψη αυτό ε, και μάλιστα τις πέντε οριζόντρες ρήτρες της συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έρθουν πιο κοντά οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές της Ένωσης πιο κοντά στις ανησυχίες των πολιτών. Σταματώ εδώ την ανάγνωση προς το παρόν κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Γιώλα είναι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακούσαμε τρεις ε, εξαιρετικές εισαγωγές που ε, είναι σημαντικές για τις εκθέσεις και της κυρίας Μπρέσο και το συμπέρασμα είναι ότι με τις συνθήκε που έχουμε μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα άλλωστε των εργασιών που είχαν γίνει τότε στην συντακτική συνέλευση. Λέγαμε ότι υπάρχουν ήδη πολλές ε, ρυθμίσεις και μέτρα που επιτρέπουν ε, ευελιξία. Θα είχα να κάνω δύο ερωτήσεις. Ο Ρενέ Ρεπάζη εξήγησε πολύ καλά για το μηχανισμό κυρώσεων στην Ευρωζώνη, ότι είναι σχετικά περιορισμένος και θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ε, μηχανισμός με κίνητρα η δημοσιονομική δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι δεδομένη. Το χρήμα είναι κίνητρο για να κάνεις κάτι που είσαι απρόθυμος να πράξεις. Αν η Ευρωζώνη έχει δικό της προϋπολογισμό, τίθεται το εξής ερώτημα τώρα. Πώς θα αποφασίζουμε εμείς στο Κοινοβούλιο. Και ρωτώ τον ναι, Ρενέ Ρεπάζη, έχει καμιά ιδέα. Γιατί τα χρήματα έρχονται από συγκεκριμένο αριθμό κρατών μελών. Αλλά εμείς είμαστε ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι Κοινοβούλιο Ευρωζώνης. Πώς θα ψηφίζουμε τον προπολογισμό της Ευρωζώνης. Δεύτερο σχόλιο προς την κυρία Κρεμόνα που πολύ ωραία μας εξήγησε ότι έχουμε ένα δημοκρατικό έλλειμμα ε, στη διεθνή παρουσία και δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παρελθόν αυτό ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα και πολιτική της εκτελεστικής εξουσίας και η κοινή γνώμη και τα κοινοβούλια ε, ήταν εκτός. Ε, τώρα ζούμε σε καιρούς ίντερνετ και είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Το βλέπουμε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η συμφωνία TTIP. Η κοινή γνώμη επαγρυπνεί. Η ε, κοινότητα των ΜΚΟ είναι στα κάγκελα. Και ε, θα πρέπει να δούμε τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες μας. Και τίθε λοιπόν το εξής ερώτημα. Στο TTIP, δεν έχουμε δώσει εντολή, κάναμε συζήτηση στο κοινοβούλιο, αλλά όπως βλέπουμε αυτό δεν επαρκεί. Δεν γίνανε ακροάσεις. Πώς να το πω. Είναι πολύ ισοστρεφής η διαδικασία, τα λέμε μεταξύ μας στο μέλλον χρειαζόμαστε κάποιους μηχανισμούς έτσι ώστε ευθύς εξ αρχής ε, να συμμετέχει όσο γίνεται περισσότερο η κοινωνία στη συζήτηση, δημόσια και ανοιχτά. Επίσης, είπε η κυρία Κρυμόνα ότι στα μεγάλα θέματα όπως είναι αναπτυξιακή πολιτική χρειάζεται διοργανική συνεργασία και ή δυνατόν με συμμετοχή της κοινή γνώμης. Εξωτερική πολιτική λοιπόν, εμπορική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική με την έννοια της αναπτυξιακής βοήθειας, όλες αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να εκδημοκρατιστούν. Και θα με διέφερε να μάθω τι κάνουν τα άλλα κοινοβούλια. Το Αμερικανικό Κογκρέσο, ε, ε, που είναι μεγάλο κοινοβούλιο, αλλά τι γίνεται και με τα μικρότερα για εθνικά κοινοβούλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι αρμοδιότητες και εξουσίες έχουν αυτά σε σύγκριση με τόσα εμεί έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ραμόν Χαουρέγγι. Ραμόν Χαουρέγγι. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και τους τρεις για τις παρεμβάσεις και να κάνω δύο συγκεκριμένες για δύο θέματα που νομίζω ότι απασχολούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική κατά κύριο λόγο. Εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή ΤΑΞ που εξετάζει την κατάσταση των ε, συμφωνιών, ξέρετε, των φορολογικών. Ε, και όσο προχωρούμε και διαπιστώνουμε ανάγκη ε, συντονισμού της φορολογικής πολιτικής στα κράτη-μέλη, ταυτόχρονα γίνονται διάφορες συμφωνίες μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων είναι πλήρης αντίφαση αυτό. Από τη μια κάνουμε διάφορα πράγματα και από την άλλη συμβαίνουν κάποια άλλα. Ε, την περασμένη εβδομάδα εγώ κατήγγυλα ότι ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης ήταν στην Ιαπωνία και βγήκαν και δήλωναν στις ιαπωνικές ε, εταιρείες ότι μπορεί να τους ράψουν ένα κουστούμι στα μέτρα τους για να έρθουν να εγκατασταθούν στο Βέλγιο την περασμένη εβδομάδα. Ενώ ταυτόχρονα ε, η ε, Επιτροπή Τάξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχούσε και ήθελε να θέσει ένα τέρμα σε αυτές τις συμφωνίες. Και ρωτώ λοιπόν τον κύριο Ρεπάψ, υπάρχει νομική βάση στις συνθήκες για να δημιουργηθεί ε, ένας ευρωπαϊκός φορολογικός οργανισμός που να αρχίσει να παρακολουθεί, να συντονίζει, να ενημερώνει, να έχει με διαφάνεια, ε, ε, να καταπολεμά την, τον αθέμητο ανταγωνισμό στα φορολογικά. Υπάρχει τέτοια νομική βάση, γιατί νομίζω ότι ένας ευρωπαϊκός φορολογικός οργανισμός θα ήταν η λογική απορία της οδηγίας Μοσκοβισή για να ε, υπάρξει ε, συντονισμός στην ενημέρωση μεταξύ των κρατών μελών. Δεύτερο πρόβλημα, κύριε Καρέρα. Η μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι η τρομοκρατία. Έχουμε ένα πρόβλημα κοινό με τις ίδιες ρίζες και σίγουρα τα ίδια οργανωτικά πλοκάμια και επιτίθεται σε όλους αδιακρίτως στην Ευρώπη. Πριν από δεκά χρόνια και πλέον, το 2004 στην Ισπανία, αρχής γενομένης, ε, ακολούθησαν Λονδίνο, Παρίσι, Βέλγιο ε, και δεν υπάρχει αντίστοιχα απέναντι ευρωπαϊκή αστυνομία. Ερωτώ, υπάρχει βάση ε, στις συνθήκες, όχι για Ευρωπόλ και Ευρωτζάστ, αλλά μια ευρωπαϊκή αστυνομία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μια αντιτρομοκρατική, όχι συντονισμός και συνεργασία εθνικών διοκτικών αρχών, Αγνήσει. ευρωπαϊκή. Υπάρχει τέτοια νομική βάση στις συνθήκες. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ και εγώ από πλευράς μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις εμπειρογνώμονες μας έκαναν τόσες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για την εκθεσή μας. Θα ήθελα και εγώ να θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη προς τον κύριο Ρεπαζή για το θέμα των δυνατοτήτων που έχουμε ως προς τα φορολογικά και τον προπολογισμό της Ευρωζώνης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. εδώ στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας. Υπάρχουν οπωσδήποτε δυνατότητες. Όμως όταν μας λέτε fiscal είναι σαφές τι εννοούμε και δυνατότητες του προπολογισμού θα πρέπει να διασυνδέονται με τις δημοσιονομικές, αλλά και έναν προπολογισμό της Ευρωζώνης που θα χρησιμοποιεί την ενισχυμένη συνεργασία. Δηλαδή θα έχουμε ένα προπολογισμό με κάποιες ε, με τις δυνατότητες ενός πνεύμονα. Δηλαδή ε, για τη δυνατότητα χρέωσης εντός ε, του ισολογισμού μέσω της συνθήκης και μέσω της διαθρωμένης συνεργασίας είναι αυτό εφικτό ή πρέπει να υπάρξει κάποια αναθεώρηση της συνθήκης. Σε δεύτερη φάση και προς τους άλλους δύο εμπειρογνώμονες. εμπειρογνώμονες. Όπως έλεγε ο συνάδελφος, αυτή τη στιγμή η βασική μέρημνα των Ευρωπαίων πολιτών είναι οπωσδήποτε η άμυνα κατά της τρομοκρατίας και η προστασία από τρομοκρατικές επιθέσεις και όχι μόνον διεθνούς και μη προέλευσης και προς τους Ευρωπαίους πολίτες και προς τις χώρες με τις οποίες υπάρχουν διαφορετικών ειδών συμφωνίες συνεργασίας. Και εδώ στη συνθήκη Πώς βλέπετε τη δυνατότητα διαρθρωμένης συνεργασίας. Πώς μπορεί αυτά τα τρία στοιχεία να αλληλοσυσχετιστούν. Από τη μια η εξωτερική πολιτική, η πολιτική άμυνας, που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά προφανώς, διότι η πολιτική κοινή κοινή πολιτική άμυνα μάλλον, σημαίνει ότι από κοινού συνδυάζουμε το δυναμικό μερικών από τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών στρατών. Αλλά υπάρχει και το θέμα της εσωτερικής ασφάλειας, διότι γίνεται όλο και πιο δυσκερές να διακρίνουμε τη μια από την άλλη. δεδομένων των πιέσεων που δεχόμαστε έξωθεν στο εσωτερικό των χωρών μας. Αφού λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι αλληλένδετα, πώς βλέπετε την διαρθρωμένη συνεργασία για τα τρία αυτά θέματα ή τέλο πάντων για αυτό της άμυνας με την πολιτική ασφάλειας. Σας ευχαριστούμε κύριε κύριος Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι μόνο οι σοσιαλιστέ έχουν διάθεση να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση προ στιγμή. Δύο ερωτήσει. Αφού ευχαριστήσω και του τρει ομιλητέ μα. Πρώτον, κύριε Ραπαζή, είπατε ότι η Οικονομική Ένωση έχει διακυβερνητική βάση. Τι εννοούμε όμως οικονομική ένωση, μήπως εννοείται περισσότερο δημοσιονομική ένωση. Αυτό έχει διακυβερνητική διάσταση, διότι έχουμε βασικά εργαλεία όπως την κοινή αγορά, την πολιτική ανταγωνισμού, την κοινή εμπορική πολιτική, τους κοινούς κανόνες για την προστασία των καταναλωτών, και άλλους κοινού κανόνες της κοινή αγοράς που ξεπερνούν το κρατικό επίπεδο. Αυτά είναι βασικά στοιχεία της οικονομικής πολιτικής που χρησιμοποιούνται σε υπερκρατικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική όμως, εκεί υπάρχουν κάποιες λεπτές διαφορές. Όμως, μήπως πρέπει να βρούμε κάποιους κανόνες σε υπερκρατικό επίπεδο. Πάντως, την ουσία της πολιτικής αυτής την ασκούν τα κράτη-μέλη, γιατί σε κάθε περίπτωση το 98% των δημοσίων δαπανών γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Ο προπολογισμός της Ένωσης είναι 2% των ε, κρατικών δαπανών. Εάν διπλασιάζαμε ή τριπλασιάζαμε τις δημόσιες δαπάνες το 94% θα βρισκόμασταν σε υπερκρατικό επίπεδο. Γι' αυτό η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προβλέψει κανόνες για το πώς τα κράτη-μέλη συμπεριφέρονται και ασκούν τις δυνατότητές τους ως προς τον προπολογισμό τους, το χρέος τους, τις δαπάνες τους και πώς αυτό επιδρά στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Όμως, το πώς δαπανούν τα κράτη για την παιδεία, τις συντάξεις, την άμυνα και ούτω καθεξής, τι θα φορολογήσουν, πού θα δαπανίσουν, αυτό είναι κάτι που θα δαπανησουν αυτο ειναι κατι που καθοριζεται σε εσωτερικό επίπεδο. Και προφανώς αυτό είναι και το σωστό. Ίσως σε επίπεδο ευρωζώνη θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιε δημοσιονομικέ δυνατότητε. Δεν διαφωνώ, αλλά πού θα γίνεται η δαπάνη, σε ποια στοιχεία του προπολογισμού. Ποια θα είναι αυτά τα στοιχεία που θα ξεχωρίσουμε και δεν θα βρίσκονται ούτε σε κρατικό ούτε σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο ευρωζώνη. Μήπω πρόκειται για μια δυνατότητα δανεισμού και χρηματοδότηση. Μήπω αυτή τη δυνατότητα πρέπει να ενισχύσουμε και έτσι βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τα χρέη τους. Αυτή είναι η ερώτησή μου προς τον κύριο Ραπαζή. Και τώρα, για τον κύριο Καρέρα. Είπατε κάτι στην παρουσίασή σας ότι οι πολίτες έχουν διαφορετικά δικαιώματα αναλόγως με το που ε, βρίσκονται. Προφανώς όμως πρέπει όλα τα δικαιώματα να είναι πανομοιότυπα ασχέτως με το που διαμένει κανείς. Ας δούμε δύο παραδείγματα. Αν είμαι στο Βέλγιο, είμαι υποχρεωμένος να έχω πάνω μου μια ταυτότητα, ένα δελτίο ταυτότητας ή ένα διαβατήριο. Το ίδιο και σε πολλές άλλες χώρες. Αν βρίσκομαι στις κατοχώρε ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία, δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Τα δικαιώματά μου διαφέρουν. Όμως, επί της ουσίας δεν ε, αλλάζει κάτι, δεν απαιτείται εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο εδώ. Εάν ήμουν ομοφιλόφιλος θα μπορούσα να παντρευτώ σε πολλά κράτη-μέλη, αλλά όχι σε όλα. Ακόμα και στη δική μου χώρα, το Ενωμένο Βασίλειο, θα μπορούσα να παντρευτώ. Εάν ήμουν ομοφιλόφιλος, θα μπορούσα να παντρευτώ έναν άλλον άντρα, στην Αγγλία, την Ουαλία, αλλά όχι στη Βόρεια Ιρλανδία. Μπορεί να διαφέρουν τα δικαιώματα και εντό του ίδιου κράτου μέλου. Σε αυτή την περίπτωση, κρίμα θα ήταν βέβαια, αλλά είναι ανάγκη να έχουμε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή μήπω πρέπει τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στη χάρτα των δικαιωμάτων να προστατεύονται. Και αυτά που τα προστατεύει και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και όχι για το καθένα δικαίωμα ξεχωριστά. Και προς τους συναδέλφους, με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να φύγω στις 11 ε, και 4 Θα πρέπει να μιλήσω για τις ε, τρέλες του Βρετανού Πρωθυπουργού σε μια άλλη συνεδρίαση. Οπότε ζητώ συγγνώμη από όλου. Πρόεδρος. Κάποιος άλλος μήπως θα ήθελε να πάρει το λόγο. Εγώ θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Γενικής φύσεως. Ε, ποια είναι τα όρια της κατακαιρματισμένη Ευρώπης, γιατί ο Γκίφερ Χόστοφ αναφέρθηκε σε αυτές τις πολλέ ε, Ευρώπε. Υπάρχει όριο αυτού του ε, κατακαιρματισμού, ποια είναι η τελική κόκκινη γραμμή. Δεύτερον, αναφερθήκατε ε, στην ε, συνήθη ε, νομοθετική διαδικασία στα πλαίσια των συνθήκων. Δεν θα μπορούσαμε όμως να χρησιμοποιήσουμε μια πασαρέλα ή κάτι άλλο πολλές δυνατότητες. Γιατί, επομένως η ερώτησή μου, γιατί αυτή η επιβολή είναι τόσο, η ενίσχυση είναι τόσο ε, κακή γιατί ξέρουμε ότι ο καθένας στα κράτη-μέλη έχει είδος διαφορετική όρεξη, αλλά δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Ε, ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία γραπτά στις συνδίκες που δεν επιτρέπουν καλύτερη ενδυνάμωση. Επίσης, ο κύριος Ρεπάση αναφέρθηκε ε, στην δυνατότητα χρήση της διαθεσμικής συμφωνίας, ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε εκμεταλλευτούμε καλύτερα, να αξιοποιήσουμε καλύτερα και πληρότερα την συνθήκη. Ε, μπορείτε λίγο να μας πείτε δύο λόγια γιατί αυτή η διαθεσμική συμφωνία θα μπορούσε ε, να βοηθήσει στην πληρέστερη εκμετάλλευση των συνθήκων. Επίσης, ε, υπό τις παρούσες συνθήκες μπορούν να συνενωθούν κάποιες ε, διαδικασίες, ας πούμε, την της Κομισιόν για την Ευρωζώνη ή ε, με κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει αυτού του είδους οι λειτουργίες θα μπορούσαν να συνδυαστούν. Ε, εάν και από τη στιγμή που δεν ζητά κάποιος άλλος το λόγο ε, να απαντήσουν οι τρεις ομιλητές με τη σειρά που αποφασίσουν μεταξύ τους. Ρενέ Δεπασί, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά τα ερωτήματα τα οποία τέθησαν, αλλά ας ξεκινήσω από την αρχή. Την ερώτηση δηλαδή του Γιώλα είναι ποιος θα πρέπει να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό ή τα άλλα κοινοβούλια. Έχω σαφή άποψη. Ε, η οποία βασίζεται σε τρεις ε, ομολογίες των συνθήκων. Πρώτον, το, το ευρώ είναι ε, η, το νόμισμα, το Συμβούλιο εκπροσωπεί την Ευρώπη και, της, και το Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, εάν λάβει κανείς αυτές τις τρεις αρχές, θα καταλάβει ότι θα πρέπει να αποφασίσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την συνολική ε, ε, φορολογική πολιτική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είμαι Γερμανός, ζω ας πούμε στις ε, στις ε, κάτω χώρες και μπορώ να ψηφίσω ευρωπαϊκές εκλογές είτε για τη χώρα από την οποία προέρχομαι ή για την ε, χώρα στην οποία ζω. Εγώ ας πούμε αποφασίζω ότι θα διαλέξω τις, νομι... τις γερμανικές εκλογές ενώ ταυτοχρόνως εγώ φορολογούμε από τις κάτω χώρες. Αυτό συμβαίνει και σε πολίτες που ζουν εκτός Ευρωζώνης αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά αυτήν την έννοια θα πρέπει ο οπωσδήποτε να σκεφτούμε τα πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο σε σχέση με την ε, ηθαγένεια και σχετικά με την υπηκότητα. Η υπηκότητα εκπροσωπεί τις χώρες, οι χώρες εκπροσωπούνται από το Συμβούλιο. Ε, το να, ε, το να, πούμε, το να πούμε ότι μπορούμε να έχουμε ένα δεύτερο κοινοβούλιο για την Ευρωζώνη, όχι. Αυτό δεν ισχύει. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες της δηλαδή, εκπροσωπούνται από το Κοινοβούλιο. Τώρα, εάν θέλουμε υψηλότερη εκπροσώπηση ε, από ορισμένες ε, χώρες ε, μέλη η εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Βεβαίως μπορούν να βρεθούν πολλές λύσεις μέσω υποεπιτροπής που ενδεχομένως και κατά τύχη θα συμμετείχαν σε αυτήν κάποιοι συγκεκριμένοι ευρωβουλευτές. Αλλά εν πάση περιπτώσει το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίζει για, για το σύνολο των αποφάσεων. Δεύτερον, όσον αφορά αυτές τις ε, ε, ειδικέ φορολογικές συμφωνίες, τα tax rulings. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να γίνει, αλλά και δεύτερο τι μπορεί να γίνει στα πλαίσια των συνθήκων. Το ένα θέμα Δεν συζητιέται πολύ για το πώς δηλαδή θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Υπάρχει ήδη ε, μια αρχή, είναι η αρχή, είναι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Η ε, εθνική επιτήρηση είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να λύσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Εάν δει κανείς το θέμα των επιδοτήσεων για υπηρεσίες γενικού οικονομικού ε, ενδιαφέροντος ή συμφέροντος ε, εκεί ε, υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές. Οι ίδιες οι αρχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέματα τα οποία σχετίζονται με τις ειδικέ προλογικές συμφωνίες, tax rulings και βεβαίως το ερώτημα το οποίο με εκπλήσει πάντα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικασία επί για βορολογικά θέματα θέματα επί θεμελιωδών ε, ελευθεριών εδώ και 15 χρόνια. Οπότε έχουμε και μια συγκεκριμένη αρχή αποφάσεων και τιμιγοριών ε, του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αλλά αναρωτιέμαι γιατί δεν έχει προχωρήσει το θέμα αυτό. Δεν ξέρω εάν Έχετε συζητήσει το θέμα αυτό σε κάποια ακρόση, αλλά κατά την άποψή μου η Κομισιόν έχει ακόμα πολλές δυνατότητες τις οποίες αφήνει αχρησιμοποιείται όσον αφορά τη δυνατότητά της ε, να είναι μια φορολογική αρχή. Δεύτερον, ε, δημιουργία πραγματικής ε, ειδική φορολογικής αρχής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό όταν αφορά το, τις, τους άμεσους Η δε νομική βάση θα ήταν το άρθρο 115 αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει το πρόσχημα της ομοφωνίας ε, και πρακτικός ε, ε, θα έπρεπε να υπάρξει ομοφωνία στο Συμβούλιο, πράγμα όχι αυτονόητο. Επί της βάσεως πάντως του άρθρου 115, εναρμονισμένες αρμοδιότητες, ναι, μπορεί να υπάρξει μια τέτοια αρχή. Μάλιστα, και βάσει συνθήκης της νίκης είχαμε, είχε ληφθεί μια μία απόφαση όσον αφορά τις πρακτικές short selling. The treaty as such does not... ε, των ακαλύπτων πωλήσεων. Επίσης, είναι σαφές ε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει χρέος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, μπορούν να υπάρξουν δανειστικές ας πούμε διαδικασίες. αλλά εδώ οδηγούμε και στο ερώτημα του Ρίτσαρτ Κόρμπετ. πρώτα μία σύντομη παρατήρηση όσον αφορά την οικονομική πολιτική. Εγώ αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην, στην ΟΝΕ και στο κεφάλαιο δηλαδή ναι, αλλά έχετε δίκιο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά εσωτερικός νόμος, hard law, έτσι ώστε να ε, μπορέσουμε στην εσωτερική ε, αγορά να έχουμε μια ευρία, ε, ένα ευρύ φάσμα μάλλον διαδικασιών που θα μπορούσε να μας δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και την συνήθη νομοθετική διαδικασία. Αλλά από την άλλη πλευρά βεβαίως το Κοινοβούλιο εξαρτάται από τις προτάσεις της Κομισιόν και μπορεί κανείς να αναρωτηθεί γιατί δεν υπάρχουν προτάσεις έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν τομείς που δεν καλύπτονται από αρμοδιότητες και ακόμα χρησιμοποιούμε την μέθοδο συντονισμού και εκεί θα πρέπει να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου στον συντονισμό ε, και στην επιβολή. Ε, όσον αφορά το δεύτερο και αναφερόμενος ε, και στην προσέγγιση διακινήτρων την οποία ανέφερα στην πρώτη μου παρουσίαση ναι ε, μπορούμε να αποφασίσουμε και βάσει της νομολογίας του δικαστηρίου για το κατά πόσο θα πρέπει να επιλέξουμε την, τις άμεσες αποφάσεις ή την πολιτική δανείζει και δανείζεστε. Ε, όσον αφορά τώρα τα, τα προγράμματα οικονομικής βοήθειας εκεί ε, βασίστηκαν ε, αρχικά στη διαδικασία του δανείζεν και διανύζεστε αλλά επ' αυτής της βάσεως δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ η συζήτηση έφτασε μέχρι τα ομόλογα έργου και τίποτε άλλο. Αυτή είναι βεβαίως μια πολύ γενική τοποθέτηση αυτή που κάνω εδώ. Πάντως ε, υπάρχει μια ενγενής έλλειψη ισορροπίας, γιατί από τη μία πλευρά δεν υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσουμε μέχρι την άκρη του δρόμου και από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα de facto, υπάρχουν de facto τα ε, ευρωομόλογα, γιατί τα κράτη-μέλη είναι όλα ίσα ε, όσον αφορά τις, όσον αφορά τις διασφαλίσεις ε, ε, ε, και τους τίτλους στις ευρωπαϊκές τράπεζες και επομένως ξαναερχόμαστε στο κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε μια κοινή οικονομική πολιτική, αν θα πρέπει να ξαναφτάσουμε σε αυτή τη βασική ερώτηση του κατά πόσο θα πρέπει να επιλέξουμε το δανείζει και δανείζεστε για να φτάσουμε μέχρι την χρήση των ομολόγων. Απ' την άλλη πλευρά ρωτάτε γιατί δεν χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατότητες και γιατί δεν υπάρχει επιβολή Νομίζω ότι ε, η κρίση κατέδειξε σαφώς ότι οι μεμονωμένες προτάσεις και ο ιδιωτικός δανεισμός δεν μπορεί ε, να ε, λύσει, να δώσει λύση στο πρόβλημα και έστω και αν υπάρχουν και εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές οικονομικές και φορολογικέ ε, ε, πολιτικές, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Το όλο οικοδόμημα μέχρι τώρα απέτυχε και το είδαμε αυτό στην περίοδο της κρίσης. Ε, και χρησιμοποιήθηκαν κάποιες μεθόδους τύπου blaming and shaming μαζί με ιδιωτικό δανεισμό, αλλά τελικά είδαμε ότι δεν προχώρησε πολύ το σύστημα. Οι περισσότεροι αντιμετώπισαν μέσω κυρώσεων, αλλά οι κυρώσεις είναι μόνο οικονομικές και επομένως επίσης δεν μας ε, προωθούν ε, πάρα πολύ ε, και σίγουρα δεν οδηγεί την σταθερότητα και την ανάπτυξη. Και είδαμε και σε χώρες που διανύουν κρίση ότι οι οικονομικές κυρώσεις δεν οδήγησαν και πουθενά. Ε, και είναι σαφές πλέον ότι ε, βασιστήκαμε σε εσφαλμένες αρχές οι οποίες με τη σειρά τους είχαν βασιστεί σε, στις, ε, στις, στη γενική τοποθέτηση των, των χρηματοπιστωτικών αγορών και που οδήγησαν τελικά σε εσφαλμένες κυρώσεις. Τώρα, όσον αφορά το άλλο ζήτημα, εάν δείτε, τον συντονισμό της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής πολιτικής ε, και την διαδικασία επιτήρησης του προϋπολογισμού διαρκώς ε, υπάρχουν συστάσεις ε, της Κομισιόν ενώ το μόνο όργανο που μπορεί να αποφασίσει τελικά είναι το Συμβούλιο. Πριν γίνουν, στην ουσία η Κομισιόν είναι αυτή η οποία αποφασίζει τι θα περιλάβει στις προτάσεις της και τις συστάσεις της πριν τις προτείνει, πριν τις ε, προωθήσει ε, το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει επί ενός ψηφίσματος, μετά απευθύνεται στην Κομισιόν έτσι ώστε να κάνει μια δευτερολογία πρότασης επί της αρχής προτάσεως αν θέλετε και μετά η Κομισιόν δέχεται ή όχι τις ε, τροπολογίες ή εν πάση περιπτώσει δημοσία στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να αιτιολογήσει την απόρριψη κάποιων τροπολογιών. Έτσι αυτός είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου στο υπάρχον πλαίσιο. Και αυτό εννοώ ότι θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει πριν εγκριθεί μία πρόταση από το Κολέγιο των ε, ε, επιτρόπων ε, και να γίνει μια θεσμική διευθέτηση συμφωνία ε, μεταξύ, Κοινοβουλίου και Κομισιόν πριν. Τώρα, τρίτη ερώτηση είναι βεβαίως εάν μπορεί κάποιος να κάνει δύο δουλειές, ναι γιατί όχι, αλλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες, έχω κάποια, κάποια προβλήματα υπάρχουν. Ο πρόεδρος Εκοφίν θα πρέπει να είναι υπουργό Οικονομικών στο Eurogroup γιατί θα πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο, άρα ε, μένουν απ' έξω πολλές χώρες, αποκλείονται πολλές χώρες. Ε, δεν νομίζω ότι θα ήταν η καλύτερη λύση και αυτό είναι το μόνο ο μόνος περιορισμός τον οποίο εγώ θα μπορούσα ε, να φανταστώ γιατί, είναι, γιατί αποκλείει χώρες οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιήσει το Euro. Η... Έλμαρ θες να πεις κάτι? Στο θέμα της ενισχυμένης συνεργασίας Αυτό είναι περιορισμένο στην ε, εσωτερική αγορά γιατί ε, έχει να κάνει με τη λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία και το Κοινοβούλιο δεν έχει κατανόηση γι' αυτό και επίτηδες έχει περιοριστεί. Γιατί δεν θέλησαν να υπάρξει ένα ξύλωμα στην εσωτερική αγορά ε, που θα υπήρχε με την ομοφωνία. Αλλά διαπιστώνουμε στην πράξη ότι τα Υπουργικά Συμβούλια σε όλο και αυξανόμενο ρυθμό και ε, ε, ταχύτητα αρνούνται να αποφασίσουν. Συμφωνούν να μην ε, χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία να το παραπέμπουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που καλείται πάντα να αποφασίζει ομόφωνα δηλαδή με την πρακτική συμπεριφορά των Υπουργών ε, καταργείται ουσιαστικά η δυνατότητα της ε, αποφάσεων κατά πλειοψηφία συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων των Υπουργών Οικονομικών. Βλέπετε καμία δυνατότητα να υπενθυμίσουμε στους Υπουργούς Οικονομικών ότι έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και να αναλάβουν την ευθύνη τους. Και αν ε, αυτό το αρνούνται δεν συνιστά παραβίαση της συνθήκης. Ε, το, συμφωνώ 100% με αυτό που λέτε και εγώ το ίδιο θα επιθυμούσα το Κοινοβούλιο ε, ακριβώς να προσφύγει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Βάσει του άρθρου 114 για την εσωτερική αγορά. Και το Συμβούλιο αυτό το έχει κόψει, το έχει βγάλει ε, σε μια διεθνή σύμβαση, που, ε, συνθήκη μάλλον που ζητάει ομοφωνία, ακριβώς αυτό που εσείς περιγράψατε. Και εδώ το Συμβούλιο από τεχνική σκοπιά και μόνο απέρριψε συνολικά σε λίβδιν την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά έβγαλε ένα κομμάτι και είπε αυτό θα το συνεχίσουμε. Αυτό δεν γίνεται. Η Ευρωπαϊκή έχει τρομοθετική πρωτοβουλία και είτε απορρίπτεται η σύνολη πρόταση, είτε πάμε στη συναπόφαση και πάμε μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τριμερή διάλογο κτλ. Εδώ όμως το ε, Συμβούλιο ε, μπλόκαρε και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Κοινοβούλιο ε, άρχισαν τη διαδικασία επιπαραβάση ακριβώς για να θυμίσουν στο Συμβούλιο όπως είπατε την ευθύνη του και την υποχρέωσή του. Εγώ θα το θεωρούσα προηγούμενο. Το είχαμε και στα εσωτερικά και δικαιοσύνης που ε, έκανε το ίδιο νομεράκι το Συμβούλιο ε, από τη συναπόφαση το έκανε απλή ακρόαση του Κοινοβουλίου διαβούλευση. Και ε, το ίδιο πρόσωπο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και το δεν το δεχόμαστε. Ε, τι διαπιστώνω εγώ ως αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις το Κοινοβούλιο δεν προσέφυγε ε, στο δικαστήριο. Υπάρχουν δυνατότητες που έχει το Κοινοβούλιο προσφέρει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το ΔΕΚ έχει μεγάλα προβλήματα όταν ε, έτσι καταργείται η νομοθεσία χωρίς συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η καθηγήτρια um, Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλια και ερωτήσεις σας. σα ευχαριστώ. Καταρχάς, το θέμα του δημοκρατικού ελλείμματο και τη εξωτερική πολιτική και πώ μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Συμφωνώ πολύτως ότι στην εποχή του διαδικτύου Έχουμε αυξημένη πολιτική της ε, ε, συμμετοχής συγγνώμη, της κοινωνίας των πολιτών ε, στις διαδικασίες διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προσμετρήσουμε και αυτή τη δυναμική και να βρούμε και θεσμικούς μηχανισμούς προκειμένου να επιτευχθεί. Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να συζητήσουμε την επισημοποίηση ε, στις συζητήσεις για δυνητικές συμφωνίες, κυρίως όσον αφορά τους εξωτερικούς μας Να υπάρχει μια πρώτερη εντολή, αν θέλετε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η συζήτηση και στο Κοινοβούλιο, αλλά και ευρύτερα. Ακόμα και πριν συμφωνηθεί η εντολή θεωρώ ότι μετά την εντολή και ε, εφόσον έχουν ξεκινήσει και διαπραγματεύσεις υπάρχει όλη αυτή η δυναμική περιθεωρία συνωμοσία που αναπτύσσεται στην ευρύτερη κοινωνία και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την αποφύγουμε. Κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται αλλαγή τη συνθήκης. Θα μπορούσαμε ίσως να υπάρχουν κάποιες ε, κοινέ ε, ε, στρατηγικές κατευθύνσεις που θα συμφωνούνται από κοινού, κυρίως για ε, νομοθετικά ζητήματα. Και θα μπορούσαμε ίσως εδώ να αποτίσουμε και φόρο τιμής ε, στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δείξει ότι κάνει ένα άνοιγμα για τις διαπραγματεύσεις. Ίσως όμως αυτό το άνοιγμα θα μπορούσε να γίνεται ακόμα νωρίτερα. Να περάσω τώρα στην ερώτηση περί τρομοκρατίας. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε εργαλεία εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, ασφάλειας, ε, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το ερώτημα, διότι σαφώς μπορεί κάποιος να ταχθεί υπέρ μιας πιο συνεκτικής πολιτικής που θα συγκεράσει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Αλλά υπάρχουν δύο τεινά. Καταρχάς θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των οποίων εμπίπτουν στη δικαιοσύνη και στον εσωτερικών υποθέσεων και αυτά που εμπίπτουν σε θέματα ε, ασφάλειας και άμυνας ε, και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει και φυσικά υπάρχουν πολύ σοβαρέ θεσμικέ συνέπειε, ιδίω για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι όπου έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι υπάρχει πρόβλημα. Το δικαστήριο κινείται προς μια κατεύθυνση ότι μέτρα τα οποία αφορούν την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτουν σε θέματα δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων, αλλά μέτρα τα οποία αφορούν ε, διεθνή ασφάλεια εμπίπτουν στην κοινή εξωτερική ασφάλεια και άμυνα. Δεν μπορούμε όμω ε, στην πράξη να κάνουμε διακρίση μεταξύ διεθνού ασφάλεια και εσωτερικής ασφάλειας Ευρωπαϊκή Ένωση και η τρομοκρατία, ιδίω όταν βρίσκεται δίπλα στα σύνορά μα, είναι ε, μία από αυτές τις περιπτώσεις. Και θεωρώ ότι εδώ έρχεται να προσθεθεί και το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένε ε, θεσμικές ε, δομές ε, στην ΚΕΠΑ και στην κοινή πολιτική, στην ΚΕΠΑ και στην κοινή πολιτική ασφάλειας και Θεωρώ ότι αυτό είναι σαφώς σημαντικό ζήτημα και θα ήταν χρήσιμο εάν μπορούσαμε να κινηθούμε προς μια σύγκληση στη λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι κάτι βέβαια που πολλοί θα πούν ότι δεν θα συμβεί ποτέ. Αλλά ίσως θα έπρεπε να πούμε ότι ε, θα ήταν το επιθυμητό σε κάποιες περιπτώσεις. Να υπάρχει μια σύγκληση στις πρακτικές μας μεταξύ της ΕΠΑ και της ε, ε, δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων θέματα που δεν είναι θέματα ΕΠΑ. Γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία συζητούνται αυτή τη στιγμή ιδίως όσον αφορά τη σχέση ε, ε, και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυκλοφορεί ένας μύθος ότι αυτό δεν είναι δυνατόν και όπως ε, γίνεται και με τα θέματα της συμμετοχής του δικαστηρίου, νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Θα υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στη χάραξη πολιτικής, χωρίς να θυσιάσουμε και τη δημοκρατική νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται. Και θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό. Θέστε και μία ερώτηση για την ενισχυμένη συνεργασία ε, μια μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Βέβαια αυτή η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία είναι μια ευκαιρία η οποία προσφέρθηκε από τη συνθήκη της Λισαβόνας και δεν την εκμεταλλεύτηκε κανείς. Ε, και ίσως εδώ η ενισχυμένη συνεργασία στην επάκις και ΕΠΑ υπήρχε στη συνθήκη της Λισαβόνας και δεν την εκμεταλλευτήκαμε. Υπάρχει ανεπίσημα, υπάρχουν ανεπίσημοι τρόποι με τους οποίους ε, ε, η πολιτική ασφάλειας και άμυνας εκφύσεως είναι μια περίπτωση ενισχυμένης συνεργασίας, διότι θα υπάρχει συνεργασία ε, και κάποια κράτη-μέλη θα συμμετέχουν και κάποια άλλα όχι με φυσικό τρόπο και σε κάποιο βαθμό ίσως λειτουργεί ήδη αυτό το σύστημα. Αλλά κάτι το οποίο ίσως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε εδώ είναι και ο συνάδελφος ο καθηγητή Καρέρα γνωρίζει περισσότερο επί του ζητήματο, στην περίπτωση τη νόμιμη μετανάστευση υπήρξαν κάποια ενδιαφέροντα πειράματα εντό αγωγικών, διεθνείς συμφωνίες, πολύ ανεπίσημες, σε επίπεδο μνημονίου συνεννόησης. Υπήρχαν κάποιε τρίτε χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια κράτη-μέλη που ενδιαφέρονταν φυσικά για αυτές τις συμφωνίες. και εδώ θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μορφή συνεργασίας και σε άλλους τομείς, όχι μόνο στον τομέα της μετανάστευσης, αλλά και σε περίπτωση αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και ή προβλήματα ασύλου και ε, παράνομης μετανάστευσης, περισσότερο από ό,τι έχει γίνει μέχρι τούδε. Αυτό είναι ίσως ένα μοντέλο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, να έχουμε ομάδες ενδιαφερομένων κρατών μελών και άλλων ενδιαφερομένων τρίτων χωρών στην περιοχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα-δυο σχόλια τώρα προς την κυρία Χούμπνερ και τις ερωτήσεις που έθεσε για τα όρια αυτής της κατακαιρματισμένης Ευρώπης. Σαφώς και δεν έχω απάντηση στο ερώτημα του πόσο ε, πρέπει να κατακαιρματιστεί η Ευρώπη πριν διαλυθούμε, αλλά νομίζω ότι είναι ε, ένα πολύ καλό ρητορικό ερώτημα που πρέπει να τίθεται. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι δημιουργώντας όλες αυτές τις ε, αέναες παραλλαγές για το opt-in και το opt-out, ορισμένες φορές δεν σκεφτόμαστε και τι συνέπειες υπάρχουν για την εξωτερική πολιτική. Και αυτό το διαπιστώνουμε πολύ με τη δυνατότητα του ε, opt-out του Ηνωμένου Βασιλείου στο άρθρο 21 και τη δικαιοσύνη και στις εσωτερικές υποθέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί φόβοι ε, για το τι μπορεί να συμβεί. Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογή του άρθρου 21 ε, και πώς μπορεί να έχει opt-out το Ηνωμένο Βασίλειο σε διεθνείς συμφωνίες. Πώς μπορούμε να έχουμε μια ρήτρα δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων σε μια ευρύτερη ε, συμφωνία, συμφωνία σύνδεσης ή αναπτυξιακή συμφωνία. Και υπάρχουν ε, ερωτήματα για την εξωτερική ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υπάρχουν πολλαπλά opt-outs. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε και δεν αφορά μόνο τον εσωτερικό κατακαιρματισμό μας, αλλά και την ε, ε, εξωτερική ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ ε, συνδέεται ίσως και κάτι τελευταίο. Θα μπορούσαμε ίσως να περάσουμε προς την για το QNV για τη διαδικασία λήψη αποφάσεων με ε, ειδική πλειοψηφία. Υπάρχει θέμα λήψης αποφάσεων ε, σε άλλους τομείς πολιτικής. Εδώ όμως υπάρχουν ε, η δυνατότητα επικοδομητικής αποχής, η οποία δεν χρησιμοποιείται όμως. Όταν περνάει σε ψηλότερο επίπεδο πολιτική, μια ε, απόφαση που θα είναι ομόφωνη και ενοποιημένη δίνει άλλο μήνυμα και ίσως αυτό είναι το τίμημα το οποίο πρέπει να πληρώσουμε ως προς το ε, ε, επίπεδο στο οποίο μπορεί κάποιος να αποφασίσει, σε ποια σύνθεση μπορούμε να λάβουμε απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το τίμημα που πληρώνεται. Θεωρώ φυσικά ότι η ειδική πλειοψηφία είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί για άλλους τομείς πολιτικής. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, λυπάμαι. Ε, ε, φυσικά απαντήστε με την ησυχία σας, απλώς ε, θυμηθείτε ότι μας πιέζει και ο χρόνος. Σας ευχαριστώ. Να συνεχίσω στη τροχιά των σημείων που ανέφερε η ε, κυρία Κρεμόνα. Υπάρχουν εσωτερικά και εξωτερικά ε, ε, ζητήματα. Ε, ωραία, αυτό το δεχόμαστε. Το ζήτημα είναι ποιες είναι οι υποθέσεις. Και εδώ υπάρχουν κάποιες ασυναρτησίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε διάφορους υπουργούς και διάφορα υπουργεία τα οποία ασχολούνται με αρκετά ζητήματα και ενδεχομένως δεν ακολουθούν πάντα το σωστό τρόπο έτσι ώστε να έχουμε μια πραγματικά ελεύθερη δημοκρατία. Αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και σε όλους τους τομείς. Ε, η ερώτηση κλειδί λοιπόν είναι η όροι και οι προϋποθέσεις. Δεύτερο, όσον αφορά τα δικαιώματα, ε, θα πρέπει να εφαρμόζεται ταυτόσημα για όλα τα δικαιώματα. Ναι, εγώ αναφέρομαι βεβαίως σε οτιδήποτε σχετίζεται με την ελεύθερη κυκλοφορία. Όταν ελευθέρως κυκλοφορούν οι πολίτες σε άλλες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ είναι για μία ακόμα φορά παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο εν μέρη ε, ε, συμμετέχει στις αρχές για την ποινική δικαιοσύνη, αλλά ας πούμε δεν συμμερίζεται όλες τις αρχές των δικαιωμάτων των υπόπτων. Και αυτό μπορεί να είναι ε, προβληματικό ε, γιατί σχετίζεται ας πούμε και με θέματα της ε, έλλειψης διακριτικής μεταχείρισης που απαιτούμε να έχουμε μετακινούμενοι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην λησμονούμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία και ένα τελευταίο, ποια είναι τα όρια του κατακαιρματισμού, ας πούμε τα δικαιώματα των πολιτών θα μπορούσε να είναι ένα καλό παράδειγμα. Η μη ε, υπονόμευση αυτών των δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελέσει κόκκινη γραμμή για μας. Ε, θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον Πέντρο Περέιρα να ξεκινήσει, να εισαγάγει μάλλον το δεύτερο πάνελ. Uh, Θα συνεχίσουμε. Καλημέρα σε όλους. Όπως ξέρετε το δεύτερο πάνελ αφορά πτυχές της δημοκρατίας, λογοδοσίας και τη θεσμική διευθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσκεκλημένοι μας είναι ο καθηγητής Αντώνιο Παντόα Σκιώπα από, από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου καθηγητής Κρίστιαν Κάλης από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και ο κύριος Άντριου Ντάφ, πρώην μέλος του Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής Ταγματικών Υποθέσεων. Θα περάσω αυτής αμέσω στις ομιλίες των προσκεκλημένων μας και όπως είπα, πρώτος ομιλητής θα είναι ο καθηγητής Πάντουα Σκιώπα. με πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο της Παδίας το 1961, δίδαξε από το 1970, μέχρι το 1979 όπου έγινε και καθηγητής με ε, διδασκαλία στην μεσαιωνική και σύγχρονη νομική ιστορία στο Πανεπιστήμιο των Μεδιολάνων στην νομική σχολή από το 82 στο 99. Έχετε το λόγο κύριε Πάντοα και ευχαριστούμε που ήρθατε Αντώνιο. Ένα ευχαριστώ προς την ε, Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου που με προσκάλεσε και βεβαίως εδώ να εκφράσω μία συγκίνηση γιατί παρακολουθώ την ζωή του Ευρωκοινοβουλίου από τη σύλληψή του, όχι από τη γέννησή του, από την δεκαετία του 50, όταν το Ευρωκοινοβούλιο δεν ε, υπήρχε ως εκλεγμένο όργανο. Η διάρθρωση που μας παρουσιάστηκε από τους τρεις συθήνοντες της ε, Επιτροπής ΑΦΚΟ μου φαίνεται άψογη. Διότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις προκλήσεις και τα προβλήματα για να καταλήξουμε στις λύσεις περνώντας από αυτό που μας επιτρέπουν να κάνουμε προς στιγμή οι συνθήκες. Οι προκλήσεις, για να είμαι συνοπτικός, είναι τουλάχιστον τρεις. Η πρώτη είναι ότι το ευρώ παρά την πολιτική πολιτική, την ε, πιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν βρίσκεται ακόμη σε ασφαλή κατάσταση. Το ε, ευρώ ε, εφόσον δεν προστατευθεί αρκετά, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή ολόκληρου του οικοδομήματος τη Ένωση. Έπειτα, σε δεύτερη φάση, και έχει αναγκαστικά με σειρά σημασία, η πρόκληση της ανάπτυξης ή της ανεργία περισσότερο είναι τρομακτική. Οι προοπτικές, οι πρόσφατες τουλάχιστον εξελίξεις δείχνουν ότι τουλάχιστον για πολλά χρόνια θα μένει γύρω στο 10% η ανεργία αλλά ιδίως για τους νέους μπορεί να ξεπεράσει και το 20%. Όχι σήμερα αλλά και στο μέλλον. Αυτή είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Όχι μόνο από κοινωνικής ε, σκοπιάς αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως σωστά θυμίστηκε ότι υπάρχει και το άρθρο 9 άρθρο που μεταξύ των στόχων της Ένωσης συγκαταλέγει την πλήρη απασχόληση. Σε τρίτη φάση και για πρώτη φορά μετά από 60, από 60 χρόνια ειρήνης ακόμα και η ειρήνη αυτή τη στιγμή απειλείται στην Ευρώπη, όχι μόνο λόγω των πιέσεων στα ανατολικά και στα νότια, στη Μεσόγειο, αλλά και λόγω της τρομοκρατίας και της κατάστασης στην Ουκρανία. Τρεις μεγάλοι κίνδυνοι, τρεις μεγάλες αιστείες κινδύνου για τις οποίες πρέπει να αναρωτηθούμε τι πρέπει να γίνει. Δεν υποτιμώ καθόλου την ε, σημασία της λιτότητας στους εθνικούς προπολογισμού και αυτό επειδή Θεωρώ ότι το να χρεώνεται κανείς υπέρμετρα σημαίνει ότι βαρύνει υπερβολικά και υπερογκά ε, τους νέους και τις πλάτες των νέων. Φορτώνει την ευθύνη δηλαδή στους νέους. Η πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσουν στο προπολογισμό τους οι λιγότερο οι χώρες που δεν έχουν χρηστή διαχείριση ως προς τα δημοσιονομικά τους σε σχέση με αυτά που έχει ορίσει η πολιτική του Μάστριχτ είναι αυτό που μας οδηγεί στην αναζήτηση μιας ορθής πολιτικής η οποία είναι ικανή αλλά όχι αναγκαία για να λύσει τα προβλήματα αυτό μπορούμε να το πούμε μετά από κάμποσα χρόνια κρίσης δεν έχουμε θεραπεύσει την όσο οι προκλήσεις που προανέφερα και ως προς το ευρώ και ως προς την απασχόληση και την ανάπτυξη ακόμη δεν έχουν επιληθεί. Δεν έχουν βρεθεί απαντήσεις. Κάτι δεν έγινε. Το ε, πρόγραμμα Juncker προφανώς οδεύει στη σωστή κατεύθυνση και να υπογραμμίσω ότι δεν θα είχε υπάρξει πρόγραμμα Juncker εάν στις εκλογές του 2014 για πρώτη φορά δεν είχαμε τα θεμέλια για μία ε, δομή δημοκρατική και κοινοβουλευτική με την διτή νομιμοποίηση τόσο του Κοινοβουλίου όσο και των κρατών. Δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει λοιπόν τέτοιο πρόγραμμα και αυτό είναι ένα βήμα προόδου επί της ουσίας. Ως προς το Ευρωπαϊκό ε, Σύνταγμα και θα χρησιμοποιήσω αυτήν την έκφραση σκοπίμως. Λείπουν λοιπόν πολλά στοιχεία, ιδίω ως προς την οικονομία. Εκεί λείπει η, το δεύτερο σκέλος της οικονομικής διακυβέρνησης. Υπάρχει σίγουρα το κοινό που είναι υπερκρατικό, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά μέτρα για μια ευρωπαϊκή ε, οικονομική διακυβέρνηση. Δεν υπάρχουν πόροι και ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων ουσιαστικά δίνει το προβάδισμα στο διακρατικό στοιχείο, το διακυβερνητικό στοιχείο. Το πρόγραμμα Juncker Στόχο έχει να προσελκύσει τις ιδιωτικές επενδύσεις και είναι γνωστό ότι οι ιδιώτες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, αλλά θα επενδύσουν εκεί όπου υπάρχουν προοπτικές κερδοφορίες, ανάκτηση των επενδύσεών τους. Ε, υπάρχει μια σειρά όμως από δημόσια αγαθά που είναι σημαντικά για τους πολίτες και έχουν τέτοιο χαρακτήρα που μόνο με δημόσιες επενδύσεις μπορούν να αναπτυχθούν όπως η προστασία του ε, περιβάλλοντος ή η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή κάποιες πτυχές της βασικής έρευνας ή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ χρειάζονται πόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και χρειάζεται και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Να μην ε, ξεχνάμε επίσης ότι ο συντονισμός δεν σημαίνει και διακυβέρνηση. Είναι δύο, διαφορετικό, δύο διαφορετικά πράγματα κάποιο πρέπει να ενισχυθεί. Ως προς την άμυνα υπενθυμίστηκε ότι κατά την άποψη των τριών τετάρτων της κοινή γνώμης θα κόστιζε λιγότερο στους πολίτες η κοινή άμυνα. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να μην υπάρχει ε, ευρωπαϊκός μηχανισμός άμυνας, τουλάχιστον για τις χώρες που, που το θέλουν. Δεν μπορεί να επιβληθεί κάτι από στους υπόλοιπους. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν σε επίπεδο συνθήκων. Πολλά υπόθηκαν ήδη σήμερα το πρωί, οπότε θα είμαι ταχύς να περιοριστώ στο εξής. Ε, στην άμυνα. Η διαρθρωμένη συνεργασία είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ ισχυρό ως προς την οικονομία. Η ενισχυμένη συνεργασία είναι ένα ε, στοιχείο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη επαρκώς. Έχει τεράστιες δυνατότητες που, επιτρέπουν να αναλάβει ένα συγκεκριμένο ρόλο και το Ευρωκοινοβούλιο. Διότι όπως ορίζει το άρθρο 333 και το οποίο ακούστηκε ήδη, μπορεί να αποφασιστεί ομοφόνος μεταξύ των χωρών της ενισχυμένης συνεργασίας να υιοθετήσουν την τακτική νομοθετική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωκοινοβούλιο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να παρέμβει. Και μετά θα πω δυο λόγια για το πώς. Διότι εδώ προφανώς υπάρχει και ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα αρκετά περίπλοκο. Διότι αν μιλάμε για ενισχυμένη συνεργασία, αυτό αφορά ορισμένα μόνο κάτι μέλη και όχι όλα. Πέραν αυτών, και δεν στέκομαι περαιτέρω στο τι μπορεί να γίνει, υπογραμμίστηκε και υπόθηκε σήμερα το πρωί, ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες Αυτά σίγουρα δεν αρκούν. Απαιτείται και αναθεώρηση των συνθήκων. Δίπλα μου έχω έναν πρώην Ευρωβουλευτή, για τον οποίο έχω έναν τεράστιο σεβασμό, τον Άντριου Νταφ, ο οποίος στην περασμένη θητεία βρέθηκε στην καρδιά της ε, συζήτησης για την ε, νέα συνθήκη. Κάτι που θα μπορούσε να συζητηθεί. Θα μπορούσαν να ακουστούν και επικριτικά σχόλια. Αλλά τα όσα έγιναν από τη συνέλευση του 2003 και από το σχέδιο Σπινέλη του 1984 φαίνεται που καταλήξαμε. Πάντως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σήμερα και να επικεντρωθούμε σε λίγα σημεία. Το είπε και ο κύριος Φεχόφστατ. Μετά θα δούμε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε ποια ακριβώς είναι αυτά τα σημεία θα ήθελα να αναφέρω τέσσερα κυρίως. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται ευρωπαϊκή διακυβέρνηση με περισσότερες εξουσίες και αρμοδιότητες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι οι στόχοι μας είναι δύο. Η αποτελεσματικότητα και η δημοκρατία. Αποτελεσματικότητα ε, μπορεί κανείς να έχει με δύο τρόπους. Με ε, μια κυβέρνηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ενισχύοντα το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και με τη λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λογικός κανένας λόγος, ίσως για λόγους ιστορικούς ναι, αλλά όχι για λόγους λογικής, να αρνηθούμε την αρχή της λήψης αποφάσεων με την πλειοψηφία. Είναι καθοριστική σημασία όταν πρέπει να αποφασίσουμε για κοινέ υποθέσει. Βεβαίω, ομιλούμε για αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνον. Αλλά όταν πρόκειται για αρμοδιότητε αποκλειστικές ή μικτές. Η ανθρώπινη ιστορία τα τελευταία 2.500 χρόνια δύο συστήματα έχει ε, δείξει ότι επικρατούν. Πρώτα απ' όλα την κλήρωση που δεν είναι και κάτι τόσο αποτελεσματικό και μετά την καταμέτρηση. Ε, εγώ θα θυμηθώ ότι το 1079 η Εκκλησία ε, για την εκλογή του Πάπα αποφάσισε ότι χρειάζονται μόνο τα δύο τρίτα των καρδιναλίων να εγκρίνουν και ε, το υπόλοιπο το καλύτερο το Άγιο Πνεύμα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ότι γιατί για θέματα τόσο περισσότερο επίγεια και κοσμικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε τόσο πιο απαιτητικοί από το Άγιο Πνεύμα. Ε, δεν βλέπω λόγο που να προκύπτει από τον λογικό νου. Α, κατά τα άλλα, δεν λαμβάνονται αποφάσεις εφόσον περιμένουμε όλοι να συμφωνήσουν για μερικά θέματα και μερικούς τομείς. Δεν θα λαμβάνονται αποφάσεις. Ε, το ότι δεν χρησιμοποιείται το σύστημα αυτό ή δεν υπάρχει ε, τελικά λήψη απόφασης επειδή κάποιοι διαφωνούν και δεν ψηφίζουν κατά ή δεν απέχουν, βλέπουμε ότι το σύστημα ακόμα δεν είναι αποτελεσματικό και έπειτα χρειάζεται ευρωπαϊκή φορολογία. Κάτι που δεν το προβλέπουν οι συνθήκες. Εκεί θα πρέπει να έχει συμμετοχή με ψηφοφορία και το Κοινοβούλιο. Και το τρίτο που συνδέεται με το δεύτερο είναι ότι το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει πάντοτε να ε, συμμετέχει με τη διαδικασία της συναπόφασης. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ε, νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μην έχει περάσει από τη διαδικασία συναπόφασης στο Κοινοβούλιο. Διότι αλλιώ δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Το τέταρτο σημείο είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο ενός διτού ε, θεσμικού οικοδομήματος, διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε Όποιος δεν θέλει να συμμετέχει σε, αυτόν τον πιο, ε, σε αυτή την αυξημένη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην το κάνει. Όπως η Μεγάλη Βρετανία. Μπορεί να, και έχει το δικαίωμα η Μεγάλη Βρετανία να θεωρεί ότι η υπόλοιπη Ήπειρος είναι απομονωμένη. Όμως ε, δεν μπορεί να αποφασίζονται πολιτικές και να τις εμποδίζει, να μην μπορούν να προχωρήσουν οι άλλοι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι τι θα κάνουμε. Δεν είναι τόσο δύσκολο να διατηρήσουμε την ενιαία αγορά, το single market που με τη σειρά της έχει ε, τις απαιτήσει της. Δηλαδή, αν αρχίσουν όλοι τις εξαιρέσεις, το opting out, ε, αποδυναμώνεται η ενιαία αγορά. Το θεσμικό πρόγραμμα, το, το πιο ε, ευαίσθητο θεσμικό πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό του Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήταν επιζήμιο και επικίνδυνο να δημιουργηθεί και ένα τρίτο σώμα. Το είπαν πολλοί εδώ. Ε, νομίζω ότι οι εκπρόσωποι, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού λαού είναι μόνο τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και το άλλο σκέλος της δημοκρατικής νομιμοποίησης είναι τα συμβούλια, τα οποία μας θα πρέπει να αποφασίζουν πάντοτε, πάντοτε κατά, κατά πλειοψηφία. Αυτά τα δύο σημεία αρκούν. Αρκούν για να μπορέσουμε από θεσμικής ε, σκοπιάς να φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στον στόχο που θέλουμε. Τώρα, μην ξεχνάμε το εμπόδιο του άρθρου 48. Να θυμίσω ότι αν οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν το άρθρο 48 στο Σύνταγμά του, δεν θα είχαν ουδέποτε δημιουργηθεί. Θα ε, ε είχαν μείνει 9 απικίες από τις 13 τις αρχικές. Οι βασικές λοιπόν αυτές αρχές υπονοούνται ούτω ή άλλω από την αρχή τη επικορικότητα, τη δημοκρατία και τη αλληλεγγύη. Αυτέ οι αρχέ είναι ε, θεσμικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που νομικώ θα έπρεπε να υπηρεσχύουν όλων των άλλων. Και εν τέλει να ολοκληρώσω λέγοντας ότι τα στατιστικά στοιχεία που ανέφερε ο κύριος Φερχόφστατ είναι για μένα το θεμέλιο των πάντων. Υπάρχει μια επί της ουσίας συμφωνία ακόμη και σήμερα παρόλα όσα έχουν γίνει, παρά τα σφάλματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια που είναι βαρύτατα, παρόλα αυτά η ευρωπαϊκή προοπτική είναι κάτι που το θέλουν οι ευρωπαίοι πολίτες το περιμένουν από την τάξη των πολιτικών ηθινόντων. Πρέπει απλώς να την κάνουμε πραγματικότητα, να τη δώσουμε σάρκα και ωστά. Εδώ λοιπόν ε, η συνεννόηση μεταξύ των κυβερνήσεων, όχι μόνο της Γαλλίας και της Γερμανίας αλλά και των υπολείπων, είναι κάτι απαραίτητο. Η Γερμανία κατά ε, ε, παραδοσιακά ήταν πάντοτε ομοσπονδιακής κατεύθυνση. Και υπάρχει τροχοπέδιος προς τη διάθεση που εκφράζει η Γαλλία. Θα πρέπει λοιπόν και η γερμανική κυβέρνηση να καθίσει και να συζητήσει την, ε, το ενδεχόμενο μιας πραγματικής ομοσπονδιακής διάρθρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία ενώ στο εσωτερικό της το εφαρμόζει το σύστημα αυτό δεν έχει προχωρήσει στο ευρωπαϊκό. Η Γαλλία δεν θα μπορούσε πλέον να αρνείται και στο επίπεδο της οικονομικής διακυβέρνησης και στο επίπεδο της άμυνας κάτι που θα έφερνε περισσότερη ασφάλεια στους και θα κόστιζε σε κάθε περίπτωση λιγότερο. Οπότε ο δρόμος είναι ανοιχτός. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα απλώς πρέπει να υποθούν ώστε να ε, υπάρξει και μία αντιστοίχηση με τις ε, πραγματικές σημερινές ανάγκες. Δεν νομίζω ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να την αφήσουμε και να την αναβάλουμε για την επόμενη γενιά. Αυτή η γενιά πρέπει να λάβει τις αποφάσεις. Εάν δεν αναλάβει δράση αυτή η γενιά, νομίζω ότι αυτό το οικοδόμημα, αυτός ο καθεδρικός που έχουμε ε, κατασκευάσει, αλλά δεν έχουμε τοποθετήσει ακόμη τον θόλο του, θα καταρρεύσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει σημειώσει κάποιες επιτυχίες ε, ορισμένες φορές, αλλά οδέποτε έχει φτάσει τόσο κοντά στην πλήρη αποτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Δόκτωρ Παντοασιώπα. Με μεγάλη χαρά σας ακούσαμε και είμαι βέβαιος ότι θα σας γίνουν και ερωτήσεις στο τέλος. Θα ήθελα να καλωσορίσω το δεύτερο μιλητή μας, τον καθηγητή Δ. Κρίστιαν Κάλλιες από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Έχετε μέσα στο λόγο σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση ε, να έρθω και να συζητήσω μαζί σας. Καταρχάς θα ήθελα να σας κάνω κάποια σχόλια για το υπόβαθρο της παρουσίασής μου. Όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο το 1984 ήταν η έκθεση Σπινέλη εκείνη που κυριαρχούσε ε, στο Κοινοβούλιο. Το 1990 συνεχίσα στο Κολέγιο της Ευρώπης και κυριαρχούσε η συνθήκη του Μαστρίχτ. Και τα δύο ε, βασίστηκαν στην ε, αρχή της ολοκλήρωσης του Ζαν Μονέ και στην ιδέα ε, της μετάδοσης που αυτόματα οδηγεί σε πολιτική ένωση. Το spillover δηλαδή. Και στην αρχή ε, του Βάλτερ Χάλσταϊν ότι γίνεται ολοκλήρωση δια νόμου, δια δικαίου. Ε, Rechtsgemeinschaft στα γερμανικά λέγεται αυτό, για να ενωθούν διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμοί, νομικοί, κοινωνικοί, πολιτισμικοί, δια του δικαίου. Ε, κατά τη διάρκεια και την πάροδο των ετών άλλαξε ε, η φύση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα είμαστε 28 κράτη-μέλη με μεγαλύτερη ετερογένεια και είναι αυτό πρόκληση και λόγω της ευάθυσης η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ε, θίγει βασικούς τομείς πολιτικής. Αυτό που βλέπουμε και μάλιστα κυριαρχεί η σημερινή κρίση για την νομισματική ένωση. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση λοιπόν γίνεται και πιο πολιτική. Δεν μπορώ να σας δώσω νέα θεωρία, αλλά έχουμε νέες προκλήσεις. Πρόκληση ε, για ολοκλήρωση, ενώ ταυτόχρονα επικρατεί και διάλυση. Αυτό είναι ε, καινοφανές, τουλάχιστον στο βαθμό που διαπιστώνεται. Και υπάρχει ανάγκη διαφοροποίησης και ευελιξίας. Θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Και για ενισχυμένη συνεργασία. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα με την ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η ενισχυμένη συνεργασία έχει τους περιορισμούς της, περιορίζεται στις αρμοδιότητες της συνθήκης. Καμιά φορά θα πρέπει ακόμα και να δεχθούμε διακυβερνητικέ συμφωνίε αν δεν συνεργάζονται όλα τα κράτη-μέλη. Και λυπάμαι που οφείλω να το ομολογήσω αυτό, αν θέλουμε να είναι εγγυημένη η ε, επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια έχουμε και νέα ζητήματα και ερωτήματα που, θίγονται, που τίθεται ε, συγγνώμη, προς την νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τη δημοκρατία σε σύγκριση με τις περιόδους που σας προανέφερα 1984 και στη συνέχεια τη συνθήκη του Μαστρίχτ στο άρθρο 9 της συνθήκης υπάρχει μια αρχή που κατοχυρώνεται και τα επόμενα ε, ότι θα πρέπει να ενσωματώσουμε τουλάχιστον τα εθνικά κοινοβούλια στη διαδικασία της ολοκλήρωσης και αυτό το λέει και το άρθρο 10 εδάφιο 2 και αυτό είναι ε, μια αρχή των συνθήκων και θα πρέπει να ε, το παραδεχτούμε και να το αποδεχτούμε ότι θα έχουμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ε, και πολυεπίπεδη και κοινοβούλια. Μπορούμε να το συζητήσουμε κύριε Μπρόκαρα. έρχομαι τώρα στο έγγραφό μου. Ε, ο σχεδιασμός λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε το έγγραφο ενδεχομένως στα χέρια σας, ε, δεν ε, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τρία βασικά στοιχεία της κρίσης. Η τραπεζική κρίση, η κρίση δημοσίου χρέους και η κρίση ανταγωνιστικότητας που σε τελική ανάλυση ε, οδήγησε και σε κρίση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και τα τρία αυτά στοιχεία χρειάζεται να άλληλο ενισχύονται και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Και αυτό ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί. Η κρίση δηλαδή βλέπουμε ε, το πρόγραμμα της ε, ποσοτικής χαλάρωσης στα όντη της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και φοβούμε ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη κρίση και εκεί να κάνουμε θεμελιώδεις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το λεγόμενο παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγεται. Έρχομαι τώρα στη σελίδα 3 στις προτάσεις να υπάρχει ένα δεσμευτικό ε, πλαίσιο, δεσμευτικό οδικός χάρτης για να λυθεί η κρίση με τρόπο βιώσιμο, για να έχουμε αποκατάσταση και να ε, λάβουμε μελλοντικές κρίσεις χρειάζεται εμβάθυνση στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ε, ολοκλήρωση μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, βήμα-βήμα σταδιακά. Για μια ε, νέα ένωση χρειάζεται δημοσιονομική ένωση, μια γνήσια οικονομική ένωση και μια πιο βαθιά πολιτική ένωση. Οι, πέμπτη, οι πέντε πρόεδροι ε, θα κάνουν ε, μια έκθεση που θα ζητάει ε, βήματα, ας πούμε με βάση το σχέδιο του Ντελόρ, για να προχωρήσουμε και αυτό θα αποφασιστούν τέλη του έτους και αυτό θα ορίζει όχι μόνο τα απαραίτητα βήματα, αλλά και ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τις μεταρρυθμίσεις ίσως μέχρι το 2022. Είναι μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική που συμπεριλαμβάνει βήματα εντός των συνθήκων, αλλά και πέρα των συνθήκων και επέκεινα αυτών. Βασικές αρχές λοιπόν, κατευθυντήριες ε, για τη συνθήκη Λισαβόνας θα πρέπει να είναι οι ε, αρχές δημοκρατίας, κράτους δικαίου, αρχή της επικουρικότητας αλλά και αρχή της αλληλεγγύης. Ε, και, ε, στην ε, Ομισματική Ένωση θα πρέπει να γίνεται σεβαστή αρχή της σταθερότητας. Οι μηχανισμοί, η Τραπεζική Ένωση, ο νέος μηχανισμός εξυγίανσης κτλ και η Δημοσιονομική Ένωση χρειάζεται ε, συντονισμό στη διαμόρφωση των εθνικών ε, δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών. Οι εθνικές αρμοδιότητες θα παραμείνουν, αλλά θα πρέπει να συνδέονται με δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές και πιο αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο που θα απορρέει από αυτή την ευρωπαϊκή προσπάθεια. Αφετηρία θα μπορούσε να είναι ε, ε, το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ε, το δημοσιονομικό σύμφωνο όμως δεν δίνει τη δυνατότητα δεσμευτικά, νομικά δεσμευτικής παρέμβασης στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό θα πρέπει να κατοχυρωθεί ακόμα. Τέτοια νομικά μέσα βέβαια μπαίνουν στα χωράφια των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι κυρίαρχα για τον προπολογισμό. Ε, θα πρέπει να γίνουν σεβαστές εδώ οι αρχές της επικορικότητας και της αναλογικότητας. Εντός της συνθήκης της Λισαβόνα, εντός της συνθήκης επαναλαμβάνω μπορεί να υποστηρίζεται ένα κράτος μέλος για να κάνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και βασίζονται σε διμερείς συμφωνίε Ευρωπαϊκή Επιτροπής κρατών μελών. Αυτό μπορεί να είναι διοικητική υποστήριξη που είναι πολύ σημαντικό, αλλά και οικονομική βοήθεια για τις συγκεκριμένες πάντα μεταρρυθμίσεις. Πέρα τώρα από τις συνθήκες Λισαβόνας, έχουμε δικαιώματα παρέμβασης στην ε, δημοσιονομική αυτονομία των κρατών μέλων. Αυτό είναι κάτι δυνατό από πλευράς και συνταγματικής για μένα στα κράτη-μέλη. Να το δούμε ως εξής. Ε, Όσο ένα κράτος μέλος συμμορφούνται προς τις υποδείξεις και τις υποχρεώσεις, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο υπάρχουν κάποιες ε, ρυθμίσεις μη δεσμευτικέ. όπως γίνεται τώρα. Αν ωστόσο ένα κράτος μέλος παραβιάζει τα κριτήρια σταθερότητας, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να γίνονται αφηρημένες μεν πλην νομικά δεσμευτικές ε, συστάσεις ε, το κράτος όμως διατηρεί πάντα τις ε, αποφάσεις για το πού θα γίνουν οι οικονομίες. Και όταν ένα κράτος εξαρτάται από οικονομική βοήθεια του μηχανισμού σταθερότητα θα πρέπει να υπάρχουν ρητές και συγκεκριμένες ε, υποχρεώσεις όπως ισχύει και τώρα. Ένα κράτος μέλος που παίρνει λεφτά από το μηχανισμό σταθερότητας έχει χάσει ήδη τη δημοσιονομική του κυριαρχία και η απόφαση είναι είτε θα χρεοκοπήσεις είτε θα πάρεις λεφτά από τον ESM, το μηχανισμό σταθερότητας, υπό όρους. Είναι ελεύθερη απόφαση, κυρίαρχη ενός κοινοβουλίου πάντα εθνικού, ε, αλλά έτσι λαμβάνεται η απόφαση, δηλαδή η αλληλεγγύη συνοδεύεται και από όρους και υποχρεώσεις και συνδυάζεται. Ε, στην Ευρωζώνη λοιπόν Έχουμε τη Δημοσιονομική την Ένωση και την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Αυτά θα πρέπει να είναι αλληλένδετα. Ήδη από τώρα, στο άρθρο 2, ε, αναφέρεται η οικονομία της αγοράς, η κοινωνική όμως οικονομία της αγοράς και θα πρέπει αυτό να γίνεται πάντα σε συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Τα πρώτα βήματα στη συνθήκη της Λισαβόνας θα μπορούσαν να είναι τα εξής μια οδηγία για την κινητικότητα των εργαζομένων εντός των πλαισίων της συνθήκης πάντα που θα μπορεί να συνδυάζεται με την οδηγία για την ελευθερία των υπηρεσιών. Παρά το γεγονός ότι το άρθρο 45 ήδη εγγυάται τα ατομικά δικαιώματα ε, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων ε, δεν έχουν αρθεί όλα τα εμπόδια και κάθε φορά χρειάζεται απόφαση του ΔΕΚ για να επιβληθεί. Αντίστοιχα για την ελευθερία των υπηρεσιών η ιδέα είναι να έχουμε μια γενική ε, οδηγία που θα απελευθερώσει τις και θα υπάρχει ένας γενικός κανόνας αμοιβαίας αναγνώρισης. Μια οδηγία ε, όμως γενικής ε, απελευθέρωσης κυκλοφορίας θα μπορούσε να σπάσει τα εμπόδια που ακόμα υπάρχουν. Ε, επιπλέον, τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να, διαρθ... να αναμορφωθούν έτσι ώστε να υποστηρίζουν τις ε, διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Πώς θα αντισταθμιστηθούν τώρα οι οικονομικοί κραδασμοί εκτός της συνθήκης. Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα ήταν μέσα στη συνθήκη. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα μηχανισμό ασφάλισης ως μαξιλαράκι για να απορροφήσει τις ανετικές συνέπειες. Θα μπορούσε η Ευρωζώνη για παράδειγμα να έχει ένα σύστημα ασφάλισης ανεργίας κοινό ε, που θα έρθει να ε, επικουρήσει τα εθνικά συστήματα. Όλα τα συστήματα και όλες οι εθνικές αγορές εργασίας ε, που εντάσσονται στο ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι επιλέξιμα ενδεχομένω να συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα. Σε περίπτωση και ε, χρεοκοπίας μιας χώρας με όλα τα συμπεραμαντούντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διεθνείς χρηματαγορές θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα εργαλείο με αποτρεπτικό χαρακτήρα και ισχύ και με ε, προθεσμίες για την χειρότερη περίπτωση. Ο μηχανισμός σταθερότητας έτσι θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο που μαζί με τα θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να έχει τα δικαιώματα επέμβασης και παρέμβασης ε, στους εθνικούς προϋπολογισμούς και σε όλα αυτά που προανέφερα. Επιπλέον, αυτό το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να είναι σε θέση να αρχίζει μια διαδικασία πτώχευσης, χρεοκοπίας ε, ε, διαρθρωμένης και συντεταγμένης ενός κράτους μέλους της Ευρωζώνης. Θα πρέπει κάπως να θεσμοθετηθεί αυτή η δυνατότητα. Στην Ευρωζώνη, ε, πέρα πάντα από τη συνθήκη όλα αυτά που λέω, χρειάζεται μια νέα εκτελεστική εξουσία να μπορεί να δρά ανεξάρτητα όχι ΕΚΟΦΗΝ και Ευρωσύνοδος, θα πρέπει να είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το εργαλείο. Ε, θα μπορούσε να είναι ο πρόεδρος της και πέντε επίτροποι που έχουν να κάνουν με τα αντίστοιχα πεδία πολιτικής. Για παράδειγμα, της εσωτερικής αγοράς, νομισματικής ένωσης, ε, χρηματοοικονομικής σταθερότητας και εμπορίου να είναι αυτή η Επίτροπη και πάλι εκτός συνθήκης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται με τα ρυθμιστικά πακέτα και να υπογράφουν διμερείς συμφωνίες με τις χώρες, θα ε, απαντούν για απώλειες των τραπεζών και για τα δημόσια αγαθά, θα προτείνουν νομοθεσία για ε, ζητήματα οικονομικά και νομισματικά. Ε, μαζί με το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα μπορούσαν να αποτελούν αυτά εργαλεία σταδιακής επέμβασης κανονικά στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Επίσης η οικονομική κυβέρνηση χρειάζεται έναν προϋπολογισμό για να ε, υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις στις χώρες που έχουν συνάψει δεμερείς συμφωνίες. Ο προϋπολογισμός θα χρηματοδοτείται από ένα τέλος μέλους 0,5% του ΑΕΠ της κάθε χώρας. Τώρα, για τη δημοκρατική λογοδοσία, η οικονομική κυβέρνηση θα πρέπει να ελέγχεται από ένα κοινοβούλιο. Μία δυνατότητα είναι να απαρτίζεται αυτό το σώμα από βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου από κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Μπορείτε να το διοργανώσετε εντός του Κοινοβουλίου, το έχουμε ήδη συζητήσει, είναι μια δυνατότητα αυτή. Όταν γίνεται μια νομοθεσία πλαίσιο και που οθήγουν ευαίσθητα ε, σημεία πολιτικής, οικονομικά, δημοσιονομικά, προϋπολογισμού και κοινωνική πολιτική, ίσως ήταν φρόνιμο να συσταθεί και ένα τρίτο σώμα επιπλέον, όπου να συμμετέχουν και μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων ή μάλλον μόνο μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου θα έχει αρμοδιότητες μόνο σε αυτούς ευαίσθητους τομείς. Έχω την αίσθηση ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τα κράτη-μέλη και τα Εθνικά Κοινοβούλια να γίνει αναθεώρηση της συνθήκης, ενσωματώνοντάς τους σε αυτή τη διαδικασία νομοθεσίας σε, μόνο σε αυτά τα ευαίσθητα ε, πεδία το, τομείς πολιτικής όπου αλλάζει κοινωνική πολιτική, δημοσιονομική πολιτική όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συμμετέχει πουθενά αλλού το κοινοτικό κεκτημένο ε, είναι εξασφαλισμένο από πλευρά της νομοθεσία με τη σημερινή κατάσταση. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρακαλώ να μην με παρανοήσετε. Άλλη δυνατότητα. Εντός της συνθήκης θα μπορούσε να είναι δικαίωμα βέτο, κόκκινη κάρτα εθνικών κοινοβουλίων ε, σε θέματα πολιτικής αυτά τα ευαίσθητα που σας ανέφερα. Ε, για να μην μπλοκάρει όμως όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, στο ε, το βέτο μιας χώρας θα μπορεί να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να σκεφτούν και να λάβουν υπόψη την αιτιολόγηση του Εθνικού Κοινοβουλίου και αν δεν βρεθεί ένα συμβιβασμός εντός εξαμήνου, δύο είναι τα τεινά που διανοίγονται. Είτε το 1 τρίτο τουλάχιστον των υπολείπων εθνικών κοινοβουλίων υποστηρίζουν το βέτο αυτό του ενός εθνικού κοινοβουλίου και αφαιρείται η πρόταση από την ημερήσια διάταξη, είτε εάν δεν βρεθεί το 1 τρίτο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να υπερβούν αυτή την, και να παρακάψουν την απόφαση. Οπότε χρειάζεται από εκεί και πέρα ε, ομοφωνία στο Συμβούλιο. Ολοκληρώνω. Για να λειτουργήσει σωστά η νομισματική ένωση πρέπει να ευρωπαϊκή ξευρωπαϊστούν οι πολιτικές, οι κοινωνικές, οι οικονομικές, οι δημοσιονομικές, να είναι πραγματικά πολιτική ένωση, να μεταφερθούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά ε, αυτό το θεσμικό πλαίσιο και τελικά ε, αναπόφευκτα πρέπει να αλλάξουν και οι συνθήκες. Αν δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη, το παράδειγμα του Δημοσιονομικού Συμφώνου μπορεί να αποτελέσει μια ευφετερία για την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων, όπου κάποια κράτη-μέλη ε, πρωτοπορούν και έχουν τη δυνατότητα όταν μπορούν ή όταν θελήσουν τα άλλα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κρίστιαν Κάλλης. Κάντε μια σειρά από συγκεκριμένε προτάσεις και θέσατε μια σειρά από ενδιαφέροντα ζητήματα. Αυτή η τρίτη βουλή βέβαια που αναφέρεται είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Θα επανέλθουμε σε αυτό με βέβαιος. Και να δώσω τώρα το λόγο στον τελευταίο μιλητή, στον κύριο Άντριο Νταφ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις, άλλωστε είναι πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην μέλος της Επιτροπής μας. Χαιρόμαστε που είστε και πάλι εδώ και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι και πάλι εδώ. Και πρέπει να υπενθυμίσω ότι έχουν περάσει ακριβώς 12 μήνες από τις ευρωεκλογέ. Τότε με πέταξαν έξω, αλλά το λέω αυτό για να σας υπενθυμίσω ότι έχετε μόνο τέσσερα χρόνια μπροστά σας. Ο χρόνος μετράει και με ανησυχεί η απουσία ενδείξεων από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι ε, προετοιμάζεται μέχρι τώρα να αντιμετωπίσει με ιδιαίτερα ζωηρό τρόπο τα ε, πολύ σοβαρά προβλήματα διακυβέρνηση που αντιμετωπίζουμε. Ελπίζω ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα φροντίζει συνεχώς να προστατεύει την εντολή και τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ιδίω να δω ότι θα εκμεταλλευτείτε τις έξι συνταγματικές εξουσίες που διαθέτεται βάσει της παρούσας συνθήκης. Είναι σημαντικές και ίσως θα έπρεπε να τις εξετάσουμε ε, έστω για λίγο. Η πρώτη είναι στο άρθρο 14.2 της Συνθήκης, ε, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σας υποχρεώνει να ξεκινήσετε να κατανομή των εδρών μεταξύ των ε, κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω να υπάρξει κάποια πρόοδος επ' αυτού και να συμφωνήσετε ότι θα υπάρχει μια συγκεκριμένη προσέγγιση βάση τύπου η οποία θα είναι δίκαιη και ε, διάφανη. Δεύτερον, βάσει του άρθρου 223 παράγραφος 1 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλεται μια πρόταση για ένα ενιαίο εκλογικό νόμο. Το αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος στις εργασίες που έγιναν στο παρελθόν. Στην πρόταση για μια πανευρωπαϊκή έδρα δηλαδή έναν υπερεθνικό, μια υπερεθνική λίστα από την οποία θα εκλέγονται ε, αρκετά μέλη. Αυτό είναι κάτι αντίστοιχο με το Spitzen Καντιντάν, τον επικεφαλής υποψήφιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά θεωρώ ότι είναι και λογική του συνέπεια. Η τρίτη εξουσία που έχετε είναι στο άρθρο 48. Και ο Αντώνιο Πάντουα Σόρπα αναφέρθηκε σε αυτό το εξαιρετικό ε, πλάσμα του άρθρου 48 έχει πολύ σημαντικά στοιχεία. Στο 48.3, στην πρώτη παράγραφο, έχετε τη δυνατότητα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφέρετε αρνητική άποψη για την περίπτωση αναθεώρησης της συνθήκης. Έχει άλλωστε γίνει κάτι τέτοιο όσον αφορά το προτινόμενο πρωτόκολλο για το άρθρο 30 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτό έγινε με αποτελεσματικό τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχει, σε περίπτωση μάλλον που υπάρξει πρόταση αλλαγής της συνθήκης, την οποία εν μέρη θα ευνοεί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, έχετε το ελεύθερο να εκφράσετε την αναζητική σας άποψη και σας προτρέπω να το κάνετε. Επίσης, στο άρθρο 48.6... Μπορείτε να έχετε και πάλι αρνητική άποψη, με ακόμα μεγαλύτερο σθένος, για την έναρξη μιας απλουστευμένης διαδικασίας για την αλλαγή του τμήματο 3 τη συνθήκη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι πολύ σημαντική εξουσία, ιδίω εάν ένα κράτο μέλος προσπαθεί να αλλάξει ή να μετριάσει την πρακτική νομοθετική έκφραση της αρχής ελευθερίας κυκλοφορίας των ανθρώπων. Στο 48.3 δεύτερη παράγραφος έχετε τη δυνατότητα να επιμείνετε για τη σύγκληση συντακτικής συνέλευση για να αλλάξει η συνθήκη. Σε κάποιες περιπτώσεις, τις οποίες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το να επιμείνετε το να υπάρξει συντακτική συνέλευση θα είναι κάτι το οποίο δεν θα αρέσει στο λαό, θα είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσετε. Ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μεταφορική πανδώρα και θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσετε πώς θα οργανωθείτε εσωτερικώς ώστε να υπάρξει μια συντακτική συνέλευση, ε, να συζητηθούν θέματα του ε, αριθμού της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, της ε, ε, την εκχώρηση εξουσιών που θα απαιτεί μια συντακτική συνέλευση, ε, συγκεκριμένες διαδικασίες και το καθεξής. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να έχει εξετάσει το Κοινοβούλιο εκ των προτέρων, πριν ξεκινήσει η διαδικασία για τη σύγκληση συντακτικής συνέλευσης. Τέλος, φυσικά, Υπάρχει η εξαιρετική εξουσία του άρθρου 48.2 δηλαδή τη δυνατότητα να προτείνεται τροποποίηση της συνθήκης. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η όλη ουσία της έκθεσης Φερχόφστατ, την οποία αναμένουμε εναγωνίως το φθινόπωρο. Ε, φαντάζομαι ότι το Κοινοβούλιο στα πλαίσια της συζήτησης για το Brexit ε, και τις ε, συζητήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο για να αλλάξει τους όρους συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ελέγξει με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο οποιαδήποτε απόπειρα να υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο θα είναι ουσιαστικά μια υποσχετική εντολή. Ε, και θα γίνει μία απόπειρα να το προσκολήσουμε και αυτό στη συνθήκη. όταν θα γίνει επισήμως η επόμενη τροποποίησή της. Επίσης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επικριτικό και σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία εκτός πλαισίου κοινοτικού δικαίου για να μπορέσουμε να ε, κατευνάσουμε το, ε, ε, την Βρετανική κυβέρνηση. Επίσης, ξέρετε ότι έχετε και ε, το άρθρο 267, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όταν υπάρχουν επίμαχα και ευαίσθητα ζητήματα. Η άποψή μου όμως είναι ότι παρά τι ιδιαίτερα ευφυείς ιδέες που ακούσαμε από τους αναλύσαντες για τις δυνατότητες που έχετε βάσει της παρούσας συνθήκης, δεν είμαστε σε θέση να παραγνωρίσουμε και το γεγονός ότι τελικώς, και νομίζω ότι αυτό θα έρθει πάρα πολύ σύντομα, θα υποχρεωθούμε να επανέλθουμε σε πλήρη διαδικασία νέας συνθήκης. Και ελπίζω ότι αυτό θα έχει στο επίκεντρο το νέο πλαίσιο να μην είναι τόσο απογορευτικό όπως είναι οι προηγούμενες συνθήκες. Αν δείτε τις συνθήκες, τα πρώτα 2, 3, 4 άρθρα είναι εξαιρετικά, είναι διάφορε διάφορες προσδοκίες, οι ελπίδες μας, οι στόχοι μας για το τι θέλουμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όλα τα υπόλοιπα άρθρα στις συνθήκες είναι αυτά που απαγορεύεται να κάνετε τι περιορισμοί υπάρχουν, τι ε, πιέσεις, ε, τι προσκόμματα για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα έχει και μεγάλο περιθώριο ε, αποτελεσματικής δράσης σε όλα τα θέματα πολιτικής. Επομένως, αυτό το οποίο είναι επιτακτικό για την επόμενη διαδικασία είναι να πάψουν οι συνθήκες να είναι τόσο απαγορευτικές και να αρχίσουν να επιτρέπουν περισσότερα πράγματα. Και πρωτίστως βεβαίως πρέπει να ξεκινήσει μια αναζήτηση, μια πορεία ε, προς μια κυβέρνηση. Και σε σχέση με τα όσα είπε ο προλαλής σας, ε, όπως ξέρετε εγώ είμαι υπέρ ε, του ομοσπονδιακής δομής, είμαι φεντεραλιστής και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ενισχυμένες εκτελεστικές εξουσίες ώστε να μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη τις εξουσίες που έχει αυτή τη στιγμή. Έγινε μια συζήτηση στο παρελθόν για το πόσο αδύναμη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μπορεί να εφαρμόσει ε, τους ε, κανόνες συμμόρφωσης που ισχύουν. Επομένως θα πρέπει μόνο να επεκταθεί νομικός ε, η εκτελεστική εξουσία που θα είχε ούτως ή άλλως ε, μία κυβέρνηση. Παραδείγματο χάρη το να καθορίσει ε, επίσημες ποσοστώσεις. Είναι παράλογο να υπάρχουν ακόμα δυνατότητες και εξουσίες στο Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Και επίσης θα πρέπει να δώσουμε και τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκτήσει εμπιστοσύνη. Μια εμπιστοσύνη την οποία δεν έχει εδώ και πάρα πολλά ε, χρόνια. Νομίζω ότι η περίπτωση του speech and candidate βοήθησε, αλλά δεν είναι παρά το πρώτο βήμα. Και θεωρώ ότι είναι αφελές να πιστεύουμε ότι μετά από όλα όσα συνέβησαν, ότι το Συμβούλιο θα εφαρμόσει ενισχυμένη πλειοψηφία όπως θα έπρεπε με διάφανο και δημοκρατικό τρόπο. Εάν θέλει να σεβαστεί το πνεύμα της Λοσοβόνας όσον αφορά τις εξουσίες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ποτέ δεν θα διασχίσει αυτό τη ρήτρα, αυτή την πασαρέλα που έχουμε τόσο προσεκτικά συμπεριλάβει στη συνθήκη. Δεν θα συμβεί ποτέ αυτό και δεν θα συμβεί εάν δεν υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να έχει πλήρη εξουσία για διακυβέρνηση της πολιτικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ένα Υπουργείο Οικονομικών και έναν Υπουργό Οικονομικών. Αν έχουμε Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορούμε να έχουμε Υπουργείο Οικονομικών και δεν μπορούμε να έχουμε Υπουργό Οικονομικών αν δεν μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε τη διαδικασία λήψη αποφάσεων για να σχεδιάσουμε τους πόρους μας. Ε, ε, χρειαζόμαστε ένα σύστημα για τις πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και φορολογικός φεντεραλισμός. Πρέπει λοιπόν να μεταρρυθμιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να μειωθεί το μεγεθός της βεβαίως, αλλά αυτό θα αρέσει σε κάποιους γιατί θα εξοικονομήσουμε χρήματα, αλλά δεν θα επιτρέπει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, λειτουργεί σαν ειρηνευτικό σώμα. Υπάρχουν αρκετά όργανα εδώ, σε αυτή την πόλη, που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των κρατών μελών ούτως ή άλλως. Εάν γίνουν αυτά και αλλάξει έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαφώς θα πρέπει να αυξηθούν και οι εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να δρά πλήρως βάση του πεδίου εφαρμογή της παρούσας συνθήκης και με αυτό το οποίο θα περιμέναμε από μια ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα που θα έχει ε, δυνατότητες δανεισμού ως ίστατη λύση. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο διαχείρισης κρίσεων Έχουμε διάφορους νόμους που πέρασαν, ε, υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει το, η δέσμη των 6 μέτρων και τη δέσμη των 2 μέτρων, το 6-pack και το 2-pack, υπάρχει το δημοσιονομικό σύμφωνο, το οποίο συμφωνήθηκε εκτός πλαισίου κοινοτικού δικαίου και μετά το ξεχάσαμε. κωδικοποίησαμε αυτά τα που έπρεπε να ε, κωδικοποιηθούν σε πρωτογενές δίκαιο, όπως για παράδειγμα το θέμα της ε, ειδική ε, πλειοψηφίας και το πώς θα γίνονται οι ψηφοφορίες και έχουμε και τη δυνατότητα να ξανασκεφτούμε λίγο την ποιότητα αλλά και την ουσία κάποιων νομοθετημάτων. Ελπίζω ότι αυτή η διαδικασία θα μας οδηγήσει στη συνέχεια και σε μια νέα εκτίμηση αυτή τη ε, βολική ε, τριμερού κατηγοριοποίηση των αρμοδιοτήτων που έχουμε αυτή τη στιγμή στη συνθήκη. ότι ο κανόνας θα πρέπει να είναι κοινή αρμοδιότητα, αλλά να μην περιορίσουμε πάρα πολύ τις εξουσίες των κρατών μελών να δράσουν. σε τομείς ε, οι οποίοι καλύπτονται από το ε, ευρωπαϊκό δίκαιο. Και αν φυσικά γίνουν αυτές οι αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σίγουρα θα πρέπει να επεκανεξετάσουμε και τις ε, σχέσεις της με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα εδώ. Αυτή η διπλή προεδρία δημιουργεί σύγχυση, αλληλοεπικαλύψεις και ο μόνος ο οποίος το απολεμβάνει είναι ο κύριος Πούτιν. Και από πλευράς δημοκρατικής λογοδοσίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ανοησίες. Τι θα έκανα εγώ αν με ρωτούσατε, και νομίζω ότι με ρωτάτε αφού με καλέσατε εδώ σήμερα, είναι, λοιπόν, να είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αρμόδιο και το Συμβούλιο των Υπουργών. Να εφαρμόζει συγκεκριμένη συνοχή και συγκεκριμένε κατευθύνσεις για ε, το Συμβούλιο και αυτό διότι χρειάζεται. Δεν θα υπήρχε περιτροπή προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών. Νομίζω ότι έχει αποδειχθεί ότι είναι παντελώς δυσλειτουργική. Θα μπορούσαμε να τις πούμε για χαρά, σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνατε, αλλά καιρό είναι να προχωρήσουμε. Και όσον αφορά το χάρτη και έγιναν και ενδιαφέρουσα συζητήσεις. για το πώς κινδυνεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα από τον ε, κατακαιρματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ θεωρώ ότι ο χάρτης θα έπρεπε να βρίσκεται κανονικά εγγεγραμμένο στη συνθήκη και θα άλλαζα τις διάφορες οριζόντιες ρήτρες ώστε να επιτρέψουμε ε, και λίγο στο χάρτη να πάρει μια ανάσα. Και επιπλέον, επειδή ε, το δικαστήριο μας έχει υποχρεώσει, θα πρέπει να διευκρινίσουμε περαιτέρω τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του του Στρασβούργου. Όλα αυτά σημαίνουν ότι θα πρέπει να αλλάξει η εκβάθρον συνθήκη. Και θα πρέπει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο και αυτό δεν θα έπρεπε να μας αγχώνει, ίσα ίσα θα, θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε. Όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια, γι' αυτό θα γίνει η μάχη, αλλά εγώ θα ήθελα να διαγράψω το πρωτόκολλο 2 της συνθήκης που αναφέρεται σε αυτό τον ε, μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για λόγους επικουρικότητας και νομίζω ότι το βάλαμε απλώς για να ευχαριστήσουμε τα εθνικά κοινοβούλια και να νομίζουν ότι έχουν κάποια κοινοβουλευτική άποψη. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει κάποιο αποτέλεσμα εν μέρη διότι δεν καταλαβαίνουμε τι είναι επικουρικότητα. Και επίσης γιατί δεν έχουμε άποψη για το τι ακριβώς είναι κοινοβούλια. Τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν τελείως διαφορετικούς ρόλους σε κάθε περίπτωση. Και αυτό το οποίο θα έκανα εγώ, με πάσα ειλικρίνεια, είναι να τους αποδεσμεύσω από την όλη αυτή διαδικασία. Θα έλεγα ότι είναι πρόσδεκτα, μπορούν κάλλιστα να εκφράσουν την άποψή τους για όλα τα ζητήματα, να πάσα στιγμή τη, τη διάρκεια της ε, νομοθετικής και πολιτικής διαδικασίας και ίσως θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κάθετη έννοια της δημοκρατίας που είναι το πολιτικό κόμμα ώστε να είναι πιο αποτελεσματική και πιο ισχυρή η συνεισφορά τους. Αν ξεκινήσουν όλα αυτά και πάνε όλα πάρα πολύ καλά, θα πρέπει από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε να εξυγχρονίσουμε και τις κοινέ πολιτικές. Κάποιες ε, ε, επ όπως για παράδειγμα οι μεταφορές ε, δεν είναι πολύ σημαντικές, αλλά η ασφάλεια εφοδιασμού στην ενέργεια, για παράδειγμα, θα έπρεπε ε, να ε, έρθει και με σημαντική χώρωση αρμοδιοτήτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να προσπίσουμε τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών και όλων των πολιτών μας. Και κάτι τελευταίο, διότι θα βαρεθήκατε και να μ' ακούτε να μιλάω, κάτι για το Brexit. αν κρατήσουμε την, το Ηνωμένο Βασίλειο θα τους έχουμε δώσει συνέχεια να γκρινιάζουν και να απειλούν ότι θα φύγουν. Ή θα μπορούσαμε να τους βάλουμε κάπου αλλού, να τους παρκάρουμε κάπου, να τους απελευθερώσουμε για ένα διάστημα τουλάχιστον και να είναι τέτοιες οι προϋποθέσεις ώστε να καταλάβουν οι πολίτες της χώρας μου, άνδρες και γυναίκες, ότι θα θελήσουν τότε να επιστρέψουν στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ενότητας, εκεί που ανήκουν. Ευχαριστώ. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, έχουμε τέσσερις συγγεγραμμένους, αλλά πρέπει σαν πρόεδρος ε, να ε, σας ζητήσω κάτι. Δυστυχώς Στη μια μισή θα έπρεπε να είμαι στην ε, συνεδρίαση της ομάδας εξωτερικής ε, δράσης έτσι ώστε να τους πείσω να έχουμε ε, αντιπρόσωπο της Επιτροπής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα και θα ήθελα να σας ε, ζητήσω ε, να ε, επιτρέψουμε έτσι ώστε ο συνάδελφος Σέπλινγκ, ο οποίος μάλιστα από αυτόν ξεκίνησε η ιδέα μέλους της ΑΦΚΟ να πάει στις Ηνωμένε Πολιτείε να μας εκπροσωπήσει σε αυτή τη συνεδρίαση για το ταξίδι στις Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί εγώ δεν θα μπορώ να είμαι. Συμφωνείτε όλοι, είναι κανείς κατά, όχι, επομένως το συμφωνήσαμε και αυτό. Επανερχόμαστε στα σημερινά μας ζητήματα. Ο Κίφερ Χόφστατ ε, είναι μέλος της ε, Επιτροπής ε, της Διάσκεψης των Προέδρων. Επανερχόμαστε λοιπόν στα δικά μας. Έχουμε τον κύριο Μαρκούλα μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ από την Επιτροπή των Περιφερειών. Ευχαριστώ πολύ ε, τους εισηγητές ευχαριστώ και την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να σας πω πρώτα απ' όλα ότι εμείς στηρίζουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου για τη σύνταξη αυτών των δύο εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας ε, και χαιρόμαστε που έχετε έρθει σε επαφή και με την Επιτροπή των Περιφερειών για τη σύνταξη αυτών των εκθέσεων. Να σας θυμίσω ότι τον Ιούλιο στην Ολομέλη μας θα ασχοληθούμε ασχοληθούμε ε, και με το θέμα αυτό και με έκθεση ε, με παρόμοιο σχετικό θέμα. Ε, ε, η συνθήκη της ε, Λισαβόνας αποτελεί θεμελιώδες σημείο κίνησης έτσι ώστε να βελτιωθεί η νομοθετική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λαμβάνοντας υπόψη την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, η αρχή της ε, επικουρικότητας αναφέρεται ρητά στο άρθρο 5 ενώ ταυτόχρονα αυτή αναφέρεται και στο τοπικό και στο περιφερειακό επίπεδο. Ε, η Επιτροπή των Περιφερειών έχει ενισχύσει την συνεργασία της ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης ε, και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη φάση της νομοθετικής διαδικασίας. Τώρα πρέπει να δούμε το μέλλον για να χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα επιτεύγματα του παρελθόντος. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιες ιδέες. Πρώτον, να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά αυτή την έννοια, το, ε, η Επιτροπή των Περιφερειών ε, είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί μέσω διαβουλεύσεων ε, στην προσενταξιακή φάση καθώς επίσης και στη φάση των ε, ε, ε, μελετών επιπτώσεων. Επίσης, ε, σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να μελετά στις πρώτες φάσεις την επίπτωση των νομοθετημάτων. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξουν ομάδες μελέτης και στο Συμβούλιο, καθώς επίσης και μια διαδικασία υποχρεωτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Επίσης, εμείς θα θέλαμε να συμμετάσχουμε σαν παρατηρητές στις τριμερείς διαλόγους και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης. Ε, να είναι υποχρεωτική η παρουσία του εκπροσώπου ε, του δικού μας θεσμικού οργάνου σε όλες τις διαθεσμικές συζητήσεις για την ε, νομοθεσία οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, σε όλες τις πολιτικές ε, και η εδαφική ζημία. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει πιο αποτελεσματικό το ευρωπαϊκό εξάμεινο, ε, δηλαδή μέσω της συμμετοχής τοπικών και περιφερειακών αρχόντων, καθώς επίσης και την συμμετοχή εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων στις κοινοβουλευτικές εβδομάδες οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της εδαφικής συνοχής σε όλες τις πολιτικές. Εμείς προτείνουμε τρεις συγκεκριμένε βελτιώσεις, δημιουργία ειδικού συμβουλίου για την πολιτική συνοχή, ένα ε, χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα σχετίζεται και με τις υποδομές. Δεύτερον, ε, να αναγνωριστεί ως επίσημος παρατηρητής στο Συμβούλιο των ε, περιφερειών για θέματα συνοχής και επενδύσεων. Τρίτον, να δοθεί στο Συμβούλιο των Περιφερειών ε, η δυνατότητα να ε, κάνει ε, προτάσεις όσον αφορά την οικονομική και εδαφική συνοχή. Αυτό κάτι τέτοιο βέβαια θα προϋπέθεται τροποποίηση των συνθήκων. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή των συνθήκων. Αυτές, αυτή η πρόταση αλλαγή συνθήκων θα πρέπει να βασίζονται ε, σε ισχυρή πολιτική βούληση αλλά ε, και σωστές ε, μελέτες επιπτώσεων. Το Συμβούλιο των Περιφερειών θα ήθελε να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση για μελλοντική τροποποίηση των συνθήκων. Εμείς έχουμε πολλούς ε, εκπροσώπους ε, πέραν των 700 μέλων ε, μας και αυτή τη στιγμή είμαστε πανέτοιμοι έτσι ώστε να συμμετάσχουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει διάλογος με τους πολίτες έτσι ώστε να εγκαθιδρυθεί αποκεντρωμένη συνεργασία του Κοινοβουλίου με τους πολίτες. Περαιτέρω βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί μέσω τροποποίησης των ε, αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη ε, απασχολεί το Συμβούλιο των Περιφερειών ε, και έχει ξεκινήσει εσωτερικές διαδικασίες έτσι ώστε να βελτιώσει την δωρατότητα αλλά και την πραγματική συμμετοχή των, του Συμβουλίου των Περιφερειών. Ε, μία δομή η οποία θα μπορούσε να προσωμιώνεται με την, ε, ε, με την, με την συμμετοχή του Συμβουλίου των Περιφερειών εν είδη γερουσίας που θα μπορεί να συν ε, συζητάμε με το Κοινοβούλιο τα θέματα αυτά θα μπορούσε να αποτελέσει ε, μια ε, πρώτη, ένα πρώτο καλό βήμα. Παρόλα αυτά και πριν φτάσουμε σε αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλα βήματα εάν θέλει πραγματικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλύψει το δημοκρατικό έλλειμμα θα μπορούσε να δώσει και μεγαλύτερη ε, ορατότητα στην Επιτροπή των Περιφερειών. Ε, θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, επιτυχία στην εργασία των τριών συνεισηγητών ε, και να, να σας πω ότι ήδη την επόμενη εβδομάδα έχουμε ε, συνεδρίαση της Ολομέλειας Επιτροπής των Περιφερειών το θέμα που θα συζητήσει το θέμα και θα φτάσει μέχρι την Ολομέλεια του Ιουλίου. Ευχαριστώ συναδέλφοι, δεν έχουμε πολύ χρόνο οπότε που να προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι. Ο κύριος Σεψίλτ. Yes. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ. Καλώς όρισες Άντρου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω και δεν είναι η πρώτη φορά. Ε, θέλω να αναφερθώ καταρχάς και στην παρουσίασή σου και στο κείμενό σου. Όσο γίνεται πιο σύντομα θα προσπαθήσω. Ε, στη σκέψη σου και στον προβληματισμό σου. Πόσο σημαντικά και θεωρείς τη λαϊκή ε, ε νομιμοποίηση. Ποιος δίνει την νομιμότητα, ο κυρίαρχο λαό, η τεχνοκρατία, οι φιλελεύθερε αρχές και αξίε βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, αλλά εσύ πού εστιάζεις. Εγώ νομίζω ότι ε, τίνεις να υποστηρίξεις στεναρά την τεχνοκρατική κατεύθυνση και αυτό ενέχει τον κίνδυνο του να εξεγερθεί ο κόσμος κατά της Ευρώπης. Βλέπουμε ήδη τα μηνύματα. Το δεύτερο, τα Εθνικά Κοινοβούλια, πάνω κάτω απάντησε στην ερώτησή μου ήδη ε, γι' αυτό. Αλλά εάν ε, και καταργήσεις τη σχέση που υπάρχει ήδη, καλά κανείς δεν ξέρει την επικουρικότητα, ε, φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει τη δυνατότητα τριβών και θα αυξηθεί η απόσταση μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια σχέση κρατών μελών ένωσης θα πρέπει να περνάει μέσα από τα εθνικά κοινοβούλια. Μπορούμε να συζητήσουμε το μηχανισμό, δεν λέω. Ε, τρίτο θέμα. Ε, αυτό που ανέφερες ε, για την ποιοτική ή ποσοτική μείωση ε, ε, της εκπροσώπησης των μικρών και μεσαίων κρατών μέλων θα οδηγήσει σε μεγάλη ε, διάσταση και στους ευρωσκεπτικιστές. Την έχουμε ξανασυζητήσει αυτή τη συζήτηση για την αναλογική εκπροσώπηση. Και για το πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο Θυμάσαι ότι στο κοινοβούλιο δεν διακριθήκαμε για τις επιδόσεις μας. Εγώ ήμουν και παραμένω υπέρ, αλλά δεν έχω δει τίποτα να προωθεί ε, την ιδέα αυτή στο κοινοβούλιο. Δεν έχει αλλάξει κανένα ιδέα ούτε με ε, άποψη, ούτε με κάνει να πιστεύω τίποτα το αντίστοιχο. Θα έχουμε μεγάλα εμπόδια και μεγάλα ερωτηματικά μπροστά μας. Ο Έλμαρ Μπροκ. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα της νομιμοποίησης. Σίγουρα χρειάζεται κάπου να καλυφθεί ένα έδαφος και όχι στις δομές και μόνο. Δεν έχουμε καταφέρει να εξηγήσουμε στους πολίτες ποια είναι η δημοκρατική νομιμότητα. Νομιμότητα δεν είναι πώς διαρθρώνεται κάτι, αλλά πώς το αντιλαμβάνει το πολίτης. Και εκεί νομίζω εν μέρη μάλλον δεν ανταποκριθήκαμε απολύτως στην υποχρέωση παράδοσης στον πολίτη του αγαθού αυτού. Κοιτήστε ένα θέμα διαφάνειας, αποτελεσματικότητας και νομιμοποίησης. Εκεί πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, ένα συμβιβασμό σε αυτές τις διαδικασίες. Τι σημαίνει αυτό κατά Κάθε θεσμικό όργανο θα πρέπει να αποφασίζει στο επίπεδο που της αναλογεί και βρίσκεται και όχι στα διάφορα άλλα επίπεδα. Με άλλα λόγια, τα εθνικά κοινοβούλια αποφασίζουν σε εθνικό επίπεδο και ελέγχουν τις κυβερνήσεις ω μέλη του Συμβουλίου. Κάνουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και μια που μιλάτε για θέματα νομιμοποίηση, που εκπροσωπούνται ε, ε, τα κράτη δια του Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει μια γερουσία ε, ή να αντικατασταθεί από μια γερουσία. Υπάρχει το Συμβούλιο, εκπροσωπείται ε, το κάθε κράτος. Δηλαδή ο πολίτης θα καταλάβει ακόμα λιγότερο αν ε, έχει να πει και τι έχει να ορίσει. Λέμε δεν είναι αποτελεσματικό όταν θα πρέπει να συμφωνούν και οι κοιτηρείς. Δεύτερον, δεν ξέρω το Συμβούλιο πώς θα παραμείνει ε, ως σώμα που ε, απορρέει από τα εθνικά κοινοβούλια, ε, πώς θα παραμείνει ο Συμβούλιο αν συμμετέχουν και τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό είναι θέμα έθνους κράτους. Και το τρίτο είναι ο πολίτης θα χάσει τον μπούσουλα τελικά ποιος έχει ποια αρμοδιότητα για τις ανοησίες που εμείς ψηφίζουμε. Και νομιμοποίηση σημαίνει ότι θα πρέπει και ο πολίτης να καταλαβαίνει ποιος φέρει ευθύνη γιατί. Αν δεν το καταλάβει αυτό ο πολίτης δεν υπάρχει καμία ε, δημοκρατική νομιμοποίηση. Αν βάλουμε τώρα και νέα θεσμικά όργανα, άκουσα κι εγώ την ιδέα να έρθει λέει μια γερουσία από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωραία. Τέταρτη βουλή λοιπόν πάμε. Καλή σας νύχτα. Έχω μόνο να προσθέσω. Να κατεβάσουμε ρολά, να το κλείσουμε το μαγαζί και χαίρετε σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Μπορεί να το συζητήσουν ε, και μετά τα ομόσπονδα κρατήδια στη Γερμανία για το πώς θα παρισφρήσουν στο Συμβούλιο. Πράγμα που ήδη κάνουν. Γιατί έχουν αρμοδιότητα, α πούμε, Υπουργεία Πολιτισμού ή Παιδεία, ε, έχουμε μόνο σε ομοσπονδιακό επίπεδο και ήδη εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο. Αυτό δεν μπορούμε να το θεσμοθετήσουμε τώρα για όλες τις αρχές τοπική αυτοδιοίκηση. Καήκαμε, χαιρετίσματα. Αυτό που θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ για την νομιμοποίηση και θα πρέπει ίσω να το μελετήσουμε είναι πώ εσεί ε, φτάνετε στη σύνθεση αυτή του Συμβουλίου. Θεωρώ τη σημερινή λειτουργία του Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται, ε, αντισυνταγματικό, κατά των συνθηκών. Εκεί λέει το Συμβούλιο, δεν λέει τα Συμβούλια, διάφορα Ευρωπαϊκά Συμβούλια δηλαδή. Υπάρχουν επιμέρους υπουργικά συμβούλια ε, και θα πρότεινα αυτά ε, να γίνουν επιτροπές. Να υπάρχει ένα συμβούλιο και να συνεδριάζει άπαξ εβδομαδιαίως ή κάθε δύο εβδομάδες, κάθε 15 μέρες και τα επιμέρους συμβούλια, ε, τα θεματικά, να είναι επιτροπές. Αυτό αλλάζει χωρίς τροποποίηση των συνθήκων με απλούστατη ε, και αμυγή τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργία του Συμβουλίου. Και πολλά από αυτά που ζούμε ως δυσφορίες και κακό κείμενα στα κράτη-μέλη και βλέπουμε και στις εκλογές, ε, απορρέουν από αυτό. Πάνε στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη και αποφασίζουν και μετά γεννά στη χώρα τους και κάνουν τις παρθένες. Αντί να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Πρέπει να αλλάξει η δομή για να είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους στη συνταγματική συνέλευση στη Ρώμη. Μισή ώρα, την πρώτη μισή ώρα το σβήσανε. Το θυμάστε στη διακυβερνητική ε, διάσκεψη που έγινε μετά τη συντακτική συνέλευση. Το πρώτο πράγμα που κάνανε οι κυβερνήσεις στη Ρώμη είναι να σβήσουν αυτή την παράγραφο. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν ε, είμαστε εμείς εμπόδιο ε, στην νομιμοποίηση. Το, Συμβούλιο είναι και θα πρέπει να το καταλάβει ο πολίτης αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο για μια δεύτερη παρέμβαση. Το πάνελ αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα θέματα, σε ένα θέμα που είναι προσφυλές και σε μένα και σε εσά. Και είναι και ο λόγος ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Το συμβουλευτικό το όργανο που προβλέπεται από τις συνθήκες και θέτει σε εφαρμογή την αρχή της αναλογικότητας, συμμετοχής και διαβουλευσής. Μιλάω για το άρθρο 11, κυρίες και κύριοι, που μιλά για μια αρχή ενίσχυσης όλων αυτών δημοκρατική συμμετοχή μοναδική στον κόσμο και ε, ενίσχυση της ε, δημοκρατίας όπως από το άρθρο 10 και 12 της συνθήκης. Αυτό που ονομάζουμε στην Επιτροπή μας ε, Δημοκρατικό Τρίπτυχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως για να υλοποιηθούν οι διατάξεις αυτές ε, έχουμε για την ώρα ε, περιορισμένες δυνατότητες. Ιδίω για τις δημόσιες διαβουλεύσεις που ε, φαίνεται να εντείνονται αλλά θα πρέπει να οργανώνονται με πιο διαφανή τρόπο και να μην προαπλασιάζονται απλώς ή ταχώς να μετατρέπονται σε διαβουλεύσεις μέσω του διαδικτύου. Οι διαβουλεύσεις με τους πολίτες στόχο έχουν να καθιστούν γνωστά σε όλους τα Αλλά εδώ απαιτείται η συμμετοχή και της Επιτροπής των Περιφερειών και της ε, ΕΟΚΕ για να αντιμετωπίσουμε τα επικριτικά σχόλια και τις ε, αντιρρήσεις που μπορεί να προκύπτουν από τον ε, κανονισμό. Εδώ υπάρχουν μηχανισμοί για να γίνει πιο αποτελεσματική η υλοποίηση του άρθρου 11. Πρώτα απ' όλα ρητός να προβλεφθεί η ε, εφαρμογή του άρθρου αυτού βάσει της οριζόντιας επικουρικότητας, ώστε να αναγνωριστεί η σημαντική θέση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών φορέων σε όλες τις διαδικασίες. Δεύτερον, να χρησιμοποιηθεί ε, ο ΙΕΟΚΕ στο θεσμικό της ρόλο για να δημιουργηθούν φόρουμ και διαδικασίες διαβουλεύσεων ε, σχεδόν μόνιμες που ούτως ή άλλως διαρκώς επιλαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με όλη αυτή την προσπάθεια ε, για τη δημιουργία προστατευμένης αξίας, όπως το Φόρουμ για το Άσυλο, τη μετανάστευση, την ενέργεια. Επιτά, στο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να προβλέψουμε την υλοποίηση της ε, διερθωμένης συνεργασίας των πολιτών, συνεργασία με την κοινωνία δηλαδή των πολιτών και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δηλαδή αυτό να γίνει η κινητήριος δύναμη για την υλοποίηση του άρθρου 11. Μία της πρότασης αυτής βρήκα ήδη στην ε, γνωμοδότηση που ζήτησε το Ευρωκοινοβούλιο από από την ΕΟΚΕ το 2004 για την ε, υλοποίηση της συνθήκης της Ρώμης. Τέταρτη πρόταση η ΕΟΚΕ να συμμετέχει όλο και περισσότερο με διαφορεμένο τρόπο στις εξπόστα αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης μέσω μιας διαρκούς μόνιμης ε, διαδικασίας διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών ε, των κρατών μελών, ώστε να υπάρχει συμπληρωματική ερμηνεία όλων αυτών των θεμάτων. Αυτά βάζει και το πρωτοκόλλο του Ιανουαρίου του 2014 που υπογράφηκε μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και ΟΚΕ. Και τώρα το σημα... η σημαντική δεσμή μέτρων που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον στόχο καλύτερη νομοθεσία. Ένα τεράστιο πρόγραμμα με ένα στόχο που και εμεί συμμεριζόμαστε. Δηλαδή να ελαφρυνθεί καλυφθούν οι πολίτες και οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων από όλο το περιττό άχθος με δύο γραμμές που πρέπει να συμπληρωθούν. Πρώτον, να χρησιμοποιούνται καλύτερα μελέτε αντικτύπου σε όλου του νομοθετικού κύκλου και στάδια και έπειτα να διευρυνθούν οι διαβουλεύσει με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εδώ δύο παρατηρήσεις επικριτικού χαρακτήρα από την πλευρά μας. Πρώτα απ' όλα το έχω πει στον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς ε, ότι πρώτον γιατί να μην έχουμε προβλέψει σε αυτή τη φάση ένα συγκεκριμένο ρόλο για τι δύο επιτροπέ, τα δύο συμβουλευτικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΟΚΕ και την Επιτροπή των Περιφερειών. Στην πρόταση για τη νέα συμφωνία, τη νέα διαθεσμική συμφωνία με, την, με στόχο την καλύτερη νομοθεσία. Λόγω χάρη στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού. Κάτι που η Επιτροπή μα με το πρωτόκολλο που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το παρακολουθεί και ανάδει και κατάδει. Ε, δεύτερον, η δέσμη μέτρων προτείνει να δημιουργηθεί ένα νέο φόρουμ για τους ενδιαφερομένους. Δηλαδή ένας διαρκής ε, μόνιμος συνομιλητής όσων θα συμμετέχουν στη διαδικασία της καλύτερης νομοθεσίας. Εκεί καλούνται οι ΟΚΕ και οι Επιτροπή των Περιφερειών να ονομάσουν δύο εμπειρογνώμονες. Οι ΕΟΚΕ ήδη ε, είναι σε θέση να ε, το κάνει αυτό χωρίς να γίνει κάποια ιδιαίτερη διευθέτηση. Θα ήταν περίεργο, Πρόεδρε, ένα τέτοιο σημαντικό ρόλο απλούστευσης να τον υλοποιούμε πολλαπλασιάζοντας ε, τις θεσμικές διαστάσεις και τους διάβλους συμμετοχής των θεσμικών οργάνων. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο μέσα στην σημερινή διευθέντηση για να υπάρξει καλύτερη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων όπως προβλέπονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας με τις διατάξεις του άρθρου 11 και ρόλο της ΕΟΚΕ. Και... Προφανώς στο πλαίσιο του, διαδικασία της διαδικασίας αναθεώρησης της συνθήκης αυτή η διάσταση θα πρέπει να ενισχυθεί και να αποσαφινιστούν καλύτερα οι πρακτικές διαδικασίες για να γίνουν όλα αυτά. Και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι από τους συναδέλφους της ΕΟΚΕ και από πλευράς μου θα είμαστε απολύτως πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας στα πλαίσια της οποιαδήποτε συνέλευσης, ε, όπως και γίνει και στο παρελθόν, ή με την ε, συνέλευση του Λάκεν, ή με μια συντακτική συνέλευση για την επεξεργασία της νέας συνθήκης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Σπινέλη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως σκιώδης συγγήτρια για τις δύο εκθέσεις, ε, θα ήθελα να εκφράσω κάποιες αμφιβολίες ε, όσον αφορά την μη περατότητα των θεσμικών συζητήσεων που κάνουμε σε σχέση με τις πολιτικές ε, που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που εφάρμοσε τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να προσπαθήσω δηλαδή να ενοποιήσω αυτά τα δύο επίπεδα διότι ο τεχνοκρατικός κίνδυνος τον οποίο αναφέρθηκε ο συνάδελφος Σεφλίνγκ ε, καθώς επίσης και ο κίνδυνος της νομιμότητας που ανέφερε ο συνάδελφος Μπρόκ έγκυται σε αυτήν την έλλειψη ενοποίησης των πολιτικών από τη μία και των θεσμικών συζητήσεων από την άλλη. Λέω εξ αρχής ότι οι πολιτικές που ασκήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης υπήρξαν ε, κοινωνικά ε, βαθιά ε, άδικες και σίγουρα όχι απαραίτητες το νομισματικό ταμείο από το 2012-2013 έκανε μεγάλα λάθη υπολογισμού κυρίως όσον αφορά τις επιπτώσεις αυτών των πολιτικών λιτότητας επί της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Είδαμε επίσης πολλά από τα δικαιώματα τα οποία καταγράφονται στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, να ε, παραβιάζονται και σε πολλές χώρες έγινε αισθητή ε, η ανάγκη πραγματικής ένταξης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κατά την άποψή μου η πρακτική ήταν εσφαλμένη και αντιφατική και πιστεύω ότι ήταν λάθος που πιστέψαμε ότι η έλλειψη του πολιτικού πυλώνα ε, δεν θα γινόταν αισθητή ή ότι θα γινόταν αισθητή με ε, τόσο μεγάλο τρόπο ώστε να ακολουθήσει και την οικονομική πολιτική του ευρώ. Ήταν ε, εσφαλμένη θέση και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν δυσχέραναν ακόμα περισσότερο την πολιτική ένωση. και έστω και αν ε, η θεσμική μάχη είναι απαραίτητη, κατά την άποψή μου πλέον θα είναι πιο δύσκολη. Θέλω να πω ότι έχοντας ένα ευρώ το οποίο ταυτοχρόνως ε, ε, θα είχε δημιουργηθεί με την πολιτική ε, θα είχε αποτελέσματα διαφορετικά από αυτά που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Δύο ερωτήσεις. Τις αναρωτιέμαι και εγώ και τις αναφέρω και σε εσά. Πρώτον όσον αφορά την κοινή άμυνα. Συμφωνώ απολύτως με την ιδέα ότι είναι απαραίτητη η κοινή άμυνα Αναρωτιέμαι εάν τα λάθη που έγιναν με το ευρώ, δηλαδή ότι πρώτα έγινε τομεακή ενοποίηση με την ψευδέστηση ότι η πολιτική ένωση θα έρθει αργότερα, μήπως λέω κινδυνεύουμε να κάνουμε το ίδιο λάθος με την άμυνα, δηλαδή να ενοποιηθούν οι στρατοί αλλά να μην υπάρχει ε, ταυτόχρονα ή πιο πριν ακόμα η πολιτική ένωση. Θα ήθελα να σας καλέσω όλους ε, να μην ε, πιστεύουμε πάρα πολύ το ευρωβαρόμετρο. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον στις χώρες που γνωρίζω εγώ, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, ε, Αγγλία, ε, τα ε, στοιχεία είναι εσφαλμένα και οι προβλέψεις είναι εσφαλμένες εδώ και χρόνια, ιδίως δεν τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι το ευρωβαρόμετρο δεν μπορεί να είναι ε, η μόνη δημοσκόπηση, ας πούμε, η μόνη σφιγμομέτρηση που είναι σωστή. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί λοιπόν, το λέω και το ξαναλέω, το πρόβλημα της πολιτικής ένωσης ε, και καλό και της νομιμότητας και καλό την Επιτροπή μέσα στα πλαίσια των συνταγματικών προβληματισμών να μην αναφερθεί μονάχα ε, στην, στο ενδεχόμενο του Brexit αλλά και του Grexit γιατί η έξοδος ε, της Ελλάδας από το ευρώ θα μπορούσε να αποτελέσει μια συζήτηση πολύ πιο δύσκολη από ότι μια συζήτηση για το Brexit, για την έξοδο της ε, Μεγάλης Βρετανίας. Σάλς Γκέρενς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μία απλή ερώτηση στον Άντριο Ντάφ που αναφέρθηκε στην ε, κατάσταση της, ε, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπολείπων 27 μετά από τις γενικές εκλογές και που μας κάλεσε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην ξεπουλήσουμε τις αρχές της Ένωσης και σε αυτό συμφωνούμε όλοι και έτσι ώστε να δημιουργήσουμε αυτήν την νέα αναπτέρωση του ηθικού μεταξύ των πολιτών της χώρας του ε, ε, δηλαδή πώς μπορεί να γίνει αυτό με συγκεκριμένο τρόπο. Ευχαριστώ, ο Γκίφερ Χόφστατ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρώτον, ευχαριστώ για τις διαφορές παρεμβάσεις και χαίρομαι πάρα πολύ που σημειώνω ότι υπάρχει ένα σταθερό στοιχείο στη Βρετανική πολιτική είναι οι φιλελεύθερες πεπιθήσεις του Άντρου Νταφ και που δεν εθίγησαν καθόλου από τις εκλογές. Τρία πράγματα έχω να πω, σχόλια και ερωτήσεις. Πρώτον, εκπλήσουμε λίγο. Από το νέο θεσμικό οικοδόμημα που προτείνουν οι διάφοροι παρεμβαίνοντες, δεν υπόθηκε τίποτα εκεί για κάτι που για μένα είναι το βασικό καθήκον ενός κοινοβουλίου. Δηλαδή, να εγκρίνει τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Ποια, οποιαδήποτε θα είναι η δημόσια αρχή. Γιατί έχουμε κοινοβούλια, γιατί δημιουργήθηκε στην αρχή μια βουλή. Γιατί είπαμε ότι δεν νοείται φορολόγηση χωρίς εκπροσώπηση. Εμείς όμως έχουμε εκπροσώπηση χωρίς φορολόγηση τώρα. Και αυτό το πρόβλημα μέχρι τώρα δεν έχει λυθεί. Υπάρχει ομάδα υψηλού επίπεδου Μόντι που έκανε τις εκτιμήσεις της, αλλά πρέπει να το συνδέσουμε και με αυτό. Και κάπως έχω απογοητευτεί, δεν σας κρύβω. Καθηγητά κάνεις στο σημείο 20 του εγγράφου σας Μιλάτε για νέο προπολογισμό για την ε, χρηματοδότηση ενός Ταμείου Ανάπτυξης επανέρχεστε στις εθνικές συνεισφορές. Αυτό το έχουμε ξαναδεί και είναι σκέτο χάλι. Όλος ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός σήμερα είναι κατά 80% βασιζόμενος σε εθνικές συνεισφορές. Και είναι, γίνεται παζάρι κάθε φορά 6-7 χρόνια. Ε, και βλέπουμε εκεί τι γίνεται, πώς παζαρεύουν τα κράτη-μέλη. Και παντού βάζουν εξαιρέσεις, ε, εκπτώσεις, ε, όχι μόνο για τη Βρετανία, σημειώσεις και για μια σειρά άλλες χώρες ισχύει αυτό. Αυτό θα πρέπει να το ξεφορτωθούμε, να απαλλαγούμε, εν περιπτώσει, από αυτό. Έτσι κάπως έχω απογοητευτεί περίμενα να πείτε κάτι. Και πάλι εθνικός προϋπολογισμός. Ε, τουλάχιστον μιλήστε για ιδίους πόρους. Είτε με άμεση φορολόγηση των πολιτών, είτε ε, ε, οι εταιρείε να συνεισφέρουν ένα ευρωπαϊκό φόρο και με πλήρη φορολογική αυτονομία, αρμοδιότητα και για το κοινοβούλιο φορολογικό έλεγχο. Στο δεύτερο, δεν μπορώ παρά να για τον προπολογισμό έλεγχο ε, Το είπε ο Έλμαρ. Είμαστε η μόνη δημοκρατία στον κόσμο που χρειόμαστε τρία σώματα βουλής. Βρείτε μου ε, αν υπάρχει άλλη δημοκρατία που να έχει τρία σώματα. Εγώ ξέρω στις δημοκρατίες είναι, έχεις μία βουλή, βουλή και γερουσία. Και όταν έχεις δύο σώματα, το δεύτερο σώμα κοιτάει την ποιότητα της νομοθεσίας του πρώτου σώματος, την ελέγχει, και ο άλλος τύπος ή το άλλο είδος είναι στα ομοσπονδιακά κράτη που η γερουσία εκπροσωπεί τις ομόσπονδες ε, ενότητες. Ξέρω εγώ τα ομόσπονδα κράτη ίδια της Γερμανίας, περιφέρειες κτλ. Μόνο αυτά τα δύο ξέρω. Υπάρχει και τρίτο. Έχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε, τη Γερμανία, τον Καναδά ως ομοσπονδιακά κράτη. Υπάρχουν αρκετά. Ακόμα και η Γαλλία, γιατί και αυτοί έχουν Γερουσία ως δεύτερο σώμα, που εξετάζει περισσότερο την ποιότητα της νομοθεσίας. Άλλο στυλ είναι αυτό. Αλλά τρίτο σώμα δεν έχω ξαναδεί πουθενά. Είναι μοναδικό. Είναι κλασικό, χαρακτηριστικό, ευρωπαϊκό ε, παράδειγμα. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα και δεν μπορούμε να το λύσουμε, λέμε α, ας το μεγενθύνουμε. Έχουμε δύο έδρες Έχουμε δύο έδρες. Και για να λύσουμε, ας πούμε, την ΕΦΣΑ, νομίζω ότι λύσαμε το πρόβλημα. Ε, όχι, φτιάξαμε και άλλο οργανισμό. Μία για τη Φιλανδία και μία για τον κύριο Μπερλουσκόνη στην Πάρμα. και δεν είναι μόνο το ζαμπόν της Πάρμα, όχι αυτό ήταν η αιτιολόγηση ε, στο Συμβούλιο του Λάκεν όταν το συζητήσαμε. Δεν ήταν για το πρόσωπο το καθόλου. Αυτή ήταν η δικαιολογία. Ναι, τα ξέρουμε όλα αυτά. Και τελικά τι κάναμε. Ο Ευρωπαϊκός Έλεγχος γίνεται στην Πάρμα και ο συντονισμός των εθνικών ε, ε, οργανισμών τροφίμων είναι στο Ελσίνκι. Έτσι λύνουμε τα προβλήματα, τα πολλαπλασιάζουμε. Και αυτό είναι τώρα δεύτερο παράδειγμα, επειδή έχουμε πρόβλημα να φτιάξουμε ένα τρίτο σώμα. Και μετά θα έρθουν και προτάσει για τέταρτο και τα λοιπά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και που μας χρειάζεται είναι τα συμβούλια να συγχωρευτούν σε ένα συμβούλιο και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορεί αυτό το συμβούλιο το δεύτερο να γίνει το δεύτερο σώμα της Ευρωπαϊκής Βουλής. Και αυτή είναι η λύση και όχι να προσπαθήσουμε να βρίσκουμε κάθε φορά. μπορούμε να βρούμε το πρώτο σύνταγμα στην Ευρώπη του Χάινριχ Φον Πραντάνο ε, το 1852. Ε, το δικό σας, καλό ήταν. Το 1952 και το 1953 εγκρίθηκε από όλους τους εκπροσώπους ε, των έξι ιδρυτών ιδρυτικών κρατών μελών των χωρών που τότε συνέστησαν την ευρωπαϊκή κοινότητα. Δεν χρειάζεται να φέρουμε τίποτα. Αυτό το τρίτο σώμα το ξεχάσουμε καλύτερα, γιατί αρκετή σύγχυση επικρατεί. Γιατί τελικά ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος και υπεύθυνο. Εμείς που θα εκπροσωπούμε τους πολίτες ή ένα τρίτο σώμα που θα εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη. Και θέλω να ρωτήσω όλους σας το τρίτο τώρα. Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε τώρα προφορικά, δεν πειράζει. Μπορείτε να μου το στείλετε γραπτός. Αρχίσαμε πριν την νίκαια, κατά τη διάρκεια μετά την νίκαια και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να έχουμε ενισχυμένη συνεργασία. Έχουμε τις ρήθρες ευελιξίας και τις νέες πασαρέλες και δεν συμμαζεύεται. Ε, opt-out που υπήρχε εδώ και καιρό, όλα αυτά. Για ποιο λόγο τα χρειαζόμαστε. Και γιατί εφευρίσκουμε κάθε φορά και ανακαλύπτουμε περισσότερα τέτοια εργαλεία κάθε φορά. Διότι έχουμε το όρθο 48 της συνθήκης. Την ομοφωνία. Η ομοφωνία είναι ακόμα κανόνα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κάποιο τρόπο. Εγώ ήμουν μέλος των διαπραγματεύσεων με τον Μπροκ για το δημοσιονομικό σύμφωνο που ήταν μια συνθήκη εκτός της συνθήκης. γιατί δεν μπορούσαμε να τροποποιήσουμε τη συνθήκη γιατί διαφωνούσε η Βρετανία. Και ποιοι ήταν οι διαπραγματευτές. Βρετανική αντιπροσωπεία, αλλά την ώρα μας απ' έξω. Και κάθε φορά ήταν οι πρώτοι που έπαιρναν το λόγο. <laughs> Βέβαια και δεν ψηφίζαμε ποτέ. Και τελικά το δημοσιονομικό σύμφωνο έγινε δεκτό, εγκρίθηκε από την Βρετανική αντιπροσωπεία. Εγώ έτσι το κατάλαβα τουλάχιστον. Αυτό είναι επίση χαρακτηριστικό. Και εγώ τι φοβούμαι. Ότι όλα αυτά τα εργαλεία, opt-out, πασαρέλες, ενισχυμένη συνεργασία και δεν συμμαζεύεται, δεν οδηγούν προς περισσότερη ολοκλήρωση, αλλά προς περισσότερη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από σύνθεση. Η αρχική ιδέα ήταν ότι α, χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός με την ολοκλήρωση, αλλιώς χρειάζεται ομοφωνία. Τώρα βλέπουμε να ξυλώνεται η κατάσταση. Και διαλύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο λόγο? Γιατί εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο αυτό 48 και τα ε, συμπαραμαρτούντα, ομοφωνία, είναι αδύνατο να τροποποιηθούν οι συνθήκες χωρίς αυτή κτλ. Και αντί να συνεχίσουμε να θρίζουμε ειδικά συστήματα και εξαιρέσει και ρήτρε, αυτό που χρειάζεται είναι να συζητήσουμε το άρθρο 48 επί της ουσίας και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Όπως είπε και ο κύριος Παντώας Χιώπα, σαν τις αν είχαν το 48 άρθρο Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν 13 Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα. Έτσι δεν είναι. Δεν θα μπορούσε. 9 από 13 είπα. Εντάξει. Ε, και στη Φιλαδέλφια Α, να σας πω θα πάω στη Φιλαδέλφια. Ε, μάλλον προτείνω να πάμε με την ΑΦΚΟ, όχι στην Ουάσιγκτον. Εκεί συνέβησαν τα πράγματα, εκεί γράφτηκε η ιστορία, όχι στην Ουάσιγκτον. Εκεί είναι το πνεύμα της Φιλαδέλφια. Και ε, θέλουμε σούπερ ειδική πλειοψηφία. Τι είναι αυτά. Σε κάθε μεγάλο ομοσπονδιακό μόρφωμα παγκοσμίω ισχύουν τέτοια πράγματα. Για να απαλλαγούμε λοιπόν από όλες αυτές τις εξαιρέσεις, τις ειδικέ ρυθμίσεις, σημειώσεις, πασαρέλες και πάει λέγοντας, ε, ρήτρα ευελιξίας και όλα αυτά που τα τελευταία 20-30 χρόνια εφευρίσκαμε γιατί δεν είχαμε το θάρρος να ε, πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρα. Το βλέπετε κι εσείς έτσι. Και αν έχετε προτάσεις για το άρθρο 48 για να τροποποιηθεί, με χαρά να τις ακούσω. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία παρέμβαση πριν δώσουμε το λόγο στους ομιλητές, η Mercedes Μπρέσο, πολύ σύντομα παρακαλώ. Δύσκολα μπορώ σε ένα-δυο λεπτά να απαντήσω στις ερωτήσεις. Με τις τελευταίες ε, <laughs> δύο-τρεις ε, παρεμβάσεις αντιμετωπίσαμε περισσότερο πολιτικά ζητήματα. Οι ερωτήσεις μου επικεντρώνονται σε τρία σημεία. Πρώτον, μέσα από τη συνθήκη ίσως ο μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκε ο Γκίφερ Χόφστατ και πριν από λίγο και τα οποία θίξατε κι εσείς είναι ίσως να καταλήξουμε σε μια ενισχυμένη συνεργασία η οποία όμως θα περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο πολιτικό κύκλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι λοιπόν ένα μέσο το οποίο θα χρησιμοποιείται ε, αποσπασματικά και εμβαλωματικά. Θα έχουμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό κύκλο, δύο κύκλους που θα αφορούν την ε, Ευρωζώνη και την ενία αγορά. Συμφωνώ με τα όσα επενθύμησε πριν η Μπάρμπαρα Σπινέλη, εγώ θεωρώ ότι αυτός ο πολιτικός κύκλος, τουλάχιστον αυτός ο πρώτος πολιτικός κύκλος, θα πρέπει ε, κατά προτεραιότητα ε, με βάση και ίσως και μια διαρθρωμένη συνεργασία να γίνει για την ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, μια Ευρωπαϊκή Ένωση σε, χωρίς μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και το αντίστροφο. Δεύτερον, αυτό το θέμα της επόμενης, του επόμενου σώματος. Συμφωνώ απολύτως ως προς το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα μόνο νομοθετικό συμβούλιο. Αυτό έγραφε και η πρώτη εκδοχή της συνταγματικής συνθήκης. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω, αλλά μία σύνθεση νομοθετική και στα πλαίσια εντός αυτής της ε, ε, νομοθετικής δομής θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εάν τα, οι κυβερνήσεις οι οποίες υπερεκπροσωπούνται τώρα στο ε, Συμβούλιο θα μπορούσαμε να έχουμε εκπροσώπηση από πλευράς Κοινοβουλίου. Ίσως αυτό θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε. Πρέπει όμως, και νομίζω ότι αυτό είναι σαφές, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον μια νέα συντακτική συνέλευση. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να μας βοηθήσετε να καθορίσουμε το στόχο μας, να υπάρχει δηλαδή σαφής εντολής για αυτή την συνταγματική ε, συντακτική συνέλευση. Δεν θα μπορούσαν να δεχτούν ε, τα κρατη μια ανοιχτή συνέλευση και επομένως το σημείο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε είναι ακριβώς μια σαφής εντολή για αυτή τη νέα συντακτική συνέλευση για το τι δεν μπορεί να γίνει εντός της συνθήκης Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους διερμηνείς, παρά το γεγονός ότι σε λίγο θα σταματήσει η διερμηνία. Να δώσω το λόγο στους ομιλητές για τις τελευταίες παρατηρήσεις τους. Ο Αντώνιο Παντοσόπα καταρχάς. Ευχαριστώ. Δύσκολο να είμαι σύντομο. Διότι οι απόψεις που εκφράστηκαν από τους τρεις υπευθύνους της Επιτροπής σας θα πρέπει να πω ότι συνολικά συμφωνώ σε όλα. το θέμα της τρίτης, ε, του τρίτου σώματος που θα μπορούσε να δημιουργηθεί είναι κάτι που και εγώ το βλέπω έτσι. Για τα εθνικά λοιπόν κοινοβούλια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσει μια δυτή κατεύθυνση. Να δούμε πού ε, είναι το πεδίο εφαρμογή μιας οδηγίας και πώς ε, ελέγχεται η υλοποίηση από τα εθνικά κοινοβούλια. Κάποια κοινοβούλια ε, συμφωνούν ε, ως προς το σημείο μέχρι το οποίο πρέπει να πάνε και κάποια άλλα όχι. Και μετά το να δημιουργηθεί ένα τρίτο επίπεδο θα ήταν μια τεράστια αλλαγή. Για το άρθρο 48 δεν υπάρχουν αμφιβολίες. Το είπα ξεκάθαρα. Πιστεύω όμως ότι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις δεν θα γίνουν έτσι κι αύριο. Ελπίζω να γίνουν, ελπίζω ότι θα προκύψουν από εδώ από το Ευρωκοινοβούλιο, αν όλα πάνε καλά, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε χρόνια, δεν μπορούμε γιατί τρει προκλήσεις που εντοπίσαμε, του ευρώ, των κοινωνικών θεμάτων και της ασφάλειας σήμερα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όχι σε 6 χρόνια. Οπότε πρέπει να αξιοποιήσουμε τα ε, εργαλεία που μας προσφέρουν οι συνθήκες. Να επισημάνω για τις ε, μορφές ενισχυμένης συνεργασίας που ανέφερε και ο κ. Φερχόφστατ. Έχουν το ίδιο ψεγάδι, διότι απαιτούν την ομοφωνία σε όλους τους τομείς και τα παιδεία, πάνω από 50 όπου απαιτείται η ομοφωνία από τη συνθήκη, μπορεί να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία. Αλλά εκεί απαιτείται ομοφωνία, εκτός και χρησιμοποιηθεί η λεγόμενη πασαρέλα. Η πασαρέλα όμως κατά τους, ε, 28 δεν θα μπορέσει ποτέ να ε, αξιοποιηθεί. Πάντοτε μία κυβέρνηση, ξέρουμε ποια είναι αυτή, θα λέει όχι. Και ε, ισοδυναμεί αυτό με αυτοκτονία. Για να υπάρξει λοιπόν ενισχυμένη συνεργασία πρέπει όταν θέλουμε να χαράξουμε τέτοια πολιτική να περάσουμε από την πασαρέλα. Πράγμα που σημαίνει τακτική νομοθετική διαδικασία και κατά πλειοψηφία απόφαση. Το πρόβλημα είναι ότι το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες να βρεθούν λύσεις. Οι συνθήκες θα έπρεπε να προβλέπουν συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των ε, μελών της πολιτικής αυτής και αυτό θα ήταν μια ενδεχόμενη μεταρρύθμιση. Και θα πρέπει βεβαίω να δούμε τι απόψει έχουν και οι υπόλοιποι εμπειρογνώμονε. Όμω υπάρχουν και άλλα εργαλεία, λόγω χάρη συντονισμό από μια επιτροπή. Αυτό είναι το σημείο κλειδί, όπου εμεί θα έπρεπε να βρούμε μια λύση και να προχωρήσουμε. Όμω φτάνει με την ομοφωνία. Ενισχυμένη πλειοψηφία πάντοτε για όλε τι αποφάσει. Ειδικά εκεί που ισχύει ενισχυμένη συνεργασία. Και εν τέλει, γιατί πιέζει και ο χρόνο, να πω εν είδη συμπεράσματο ότι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, μία μόνο δυνατότητα νομιμοποίησης και πρόσδοσης κύρους μία μόνο τέτοια δυνατότητα διαβλέπω για να θέσουμε αυτά τα προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ευρωκοινοβούλιο. Εάν δεν αναλάβετε αυτό το ρόλο εσείς οι ευρωβουλευτές, Πραγματικά δεν έχω καμία ελπίδα, διότι οι κυβερνήσεις από μόνες τους δεν θα κάνουν τίποτα. Καθυστερούν, κάνουν σφάλματα, τα εντόπισε τα σφάλματα η κυρία Σπινέλη, με την συνηθισμένη της ε, ακρίβεια, κάνουν αυτό που θεωρούν απαραίτητο οι κυβερνήσεις και το νομίζουν αρκετό αλλά ποτέ δεν αρκεί το Κοινοβούλιο διαθέτει και τα εργαλεία αυτά του προπολογισμού, του ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά δεν μπορεί να σας τα κανένας και πρέπει να ασκούνται ως δικαιώματα. Πρέπει να ασκούνται και μάλιστα και με αυστηρότητα ε, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Για τις δημοσκοπήσεις πολλά μπορούν να υποθούν, όμως είμαι βέβαιος ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών θέλουν κοινή άμυνα, θέλουν κοινή εξωτερική πολιτική και θα κατανοούσαν και να τον και το να υπήρχε μια οικονομική πολιτική με αντικυκλική προστασία και με εργαλεία που σήμερα δεν διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα επιμέρου κράτη δεν τα διαθέτουν, διότι δεν υπάρχουν κυρίω λογαριασμοί. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό που μπορεί να καλυφθεί και αυτό μπορεί να το καλύψει μόνο η Ευρώπη. Οι πολίτε τα καταλαβαίνουν αυτά, αλλά τα καταλαβαίνουν καλύτερα από του πολιτικού κιόλα. Και σαφώ πολύ καλύτερα από τον τύπο και του δημοσιογράφου. Οπότε νομίζω ότι το στοιχείο, ε, το κομβικό σημείο σε όλα αυτά είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους διερμηνείς για τη συνεργασία τους. Θα συνεχίσουμε τώρα αποκλειστικά με αγγλικά για τις τελευταίες ε, παρεμβάσεις. Ε, maybe there was a misunderstanding with regard to the chamber, because ε,